Αγαπητοί συνάδελφοι, όσοι τουλάχιστον είστε παρόντες, ας αρχίσουμε την ε, συνάντηση της Επιτροπής μας και σας καλωσορίζω στην τελευταία μας συνεδρίαση για φέτος. Στο σημείο 1, στην ημερήσια διάταξη, στην έγκριση της ημερήσιας διάταξης, έχουμε κάποιες αλλαγές. Στο σημείο 13 πρέπει να πούμε ότι θα το συζητήσουμε σήμερα. Την έμεση αλλαγή χρήση της γης και βιοκάψιμα είναι ένα θέμα που θα το συζητήσουμε σήμερα. Ε, αύριο το πρωί αναμένουμε τον ε, πρόεδρο Μπούζεκ Και θα ήθελα και εγώ να πω δύο λόγια για τη διάσκεψη του κλίματος στο Κανκούν. Επειδή έχει διάφορες ε, συναντήσεις, ε, δεν ξέρουμε τι θα γίνει σε σχέση με την ψηφοφορία. Θα αφήσουμε χρόνο ε, για τη συνάντηση αυτή σε σχέση με τις ψηφοφορίες που έχουμε να κάνουμε. Για το, 6, για το σημείο 6, για τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης, θα το συζητήσουμε και μετά θα ακολουθήσει στο σημείο 7 που είναι το συναδέλ, για το, από το συνάδελφο Σκυλακάκη που θα πρέπει να πάει στο σημείο 17 της ημερήσιας διάταξης ε, σε σχέση με τα διάφορα ε, σημεία περιεφαρμογής. Στις, ε, στη μία θα παρουσιαστεί στην 6Q2 στη Γιάννη. 4 2, äh, θα παρουσιαστεί το θέμα αυτό που έχει με την Επιτροπή και θα το συζητήσουμε το απόγευμα στην Επιτροπή μας. Την Τετάρτη, 1η Δεκεμβρίου, στις 2, στην αίθουσά μας εδώ, στο 2Q2, θα γίνει ένα workshop για την Πράσινη Βίβλο για την Προστασία των Βασών. αποφάσισαν οι συντονιστές να διοργανωθεί ένα σεμινάριο και αυτό θα γίνει την Τετάρτη. Την 1η Δεκεμβρίου είναι η Παγκόσμια ημέρα για το AIDS και έχουμε και μία νέα έκθεση των Ηνωμένων Εθνών. Η κατάσταση δεν φαίνεται ιδιαίτερα καλή, το αντίθετο μάλιστα. 33 εκατομμύρια ε, είναι τα κρούσματα του AIDS σε ολόκληρο τον κόσμο και το μεγαλύτερο τμήμα αυτών ε, στην υποσαχάριο Αφρική. 22,5 εκατομμύρια άτομα ε, έχουν πληγεί από το AIDS στην υποσαχάριο Αφρική. Πραγματικά διαστάσεις επιδημίας λοιπόν έχει λάβει το AIDS. Στην έκθεσή μας διαπιστώνουμε ότι και στην Ευρώπη συνεχίζει να είναι οξύ το θέμα, στις βαλτικές χώρες, στην Ουκρανία, στη Ρωσία η κατάσταση είναι δραματική σε σχέση με το AIDS. Ακόμη θα ήθελα να αναφέρω το θέμα των σκουπιδιών, της κρίσης των σκουπιδιών στην Ιταλία, στην καμπάνια. Έστειλε μία αποστολή διερευνητική επιτροπή για να δει πώς πάνε τα πράγματα και η επικεφαλής της ομάδας αυτής, η κυρία Πία Μπουτσέλα, διευθύντρια, θα μιλήσει στην Επιτροπή μας την 1η Δεκεμβρίου στο σημείο που αφορά την εφαρμογή της νομοθεσίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης για το περιβάλλον. Τώρα όσον αφορά τη διάσκεψη του κλίματος στην Κανκούν, την περασμένη εβδομάδα στο Στρασβούργο ψηφίσαμε το σχετικό ψήφισμα. 299-254 ψήφων. Ε, ελπίζαμε ότι θα έχουμε μεγαλύτερη πλειοψηφία, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα. Στη συνέχεια είδα διάφορα ανακοινοθέντα στον τύπο. Και πρέπει να σας πω ότι ένα θέμα ε, μου έκανε εντύπωση. Δεν χρειάζεται να είναι κανείς ε, πάντοτε υπέρ της πλειοψηφίας, υπέρ αυτού το οποίο ψήφισε ε, η πλειοψηφία. Αλλά ο συνάδελφο ρόλο από την Επιτροπή Βιομηχανία έκανε μια δήλωση ω πρόεδρο τη Επιτροπή ε, Βιομηχανία που μιλάει για το ψήφισμα αυτό ε, που λέει ότι πρόκειται για οικονομική αυτοκτονία όταν μιλάμε για τέτοιο ψήφισμα. και είναι κάτι το οποίο θα επιτύχει αυτό που δεν έχει επιτευχθεί μετά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, δηλαδή να μεταμορφώσει τη Γερμανία σε αγροτική χώρα. Αλλά και ακόμη όσον αφορά την πολιτική του κλίματος είναι πολιτική ανοησία. Αλλά πραγματικά πιστεύω ότι οι δηλώσεις αυτές είναι λίγο υπερβολικές ως παρατραβηγμένες. Δεν νομίζω ότι μπορούμε να διατυπώνουμε τέτοιου είδους ε, κριτικές. Είναι υπερβολικές και δεν νομίζω ότι αυτή είναι και η άποψη της Επιτροπής Βιομηχανίας. Αυτές ήταν οι δικές μου ανακοινώσει. η κυρία Ντάγμαρ Ροτ Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ακριβώς αυτήν την ερώτηση ήθελα να κάνω. Το να είναι κανεί ε, πρόεδρο τη Επιτροπής είναι ένα από τα υψηλότερα αξιώματα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Μια τύχη που δεν έχει δοθεί σε όλου από εμά ή σε πολλού από εμά και αυτοί που έχουν τέτοια τιμή ε, εκφράζονται και εκ μέρου τη επιτροπή την οποία προεδρεύουν. Και γι' αυτό θα ήθελα να σα ε, παρακαλέσω να δείτε αν αυτό αυτές οι δηλώσεις είναι απόψεις επί τις οποίες έχει ψηφίσει και αποφασίσει η Επιτροπή Βιομηχανίας για αν ήταν προσωπικές απόψεις του συναδέλφου Ρόιλ, οπότε και θα πρέπει να το δηλώσει αυτό. Νομίζω ότι πραγματικά ε, είναι ανάρμοσες τέτοιες δηλώσεις. Chris Davis. Αυτά τα σχόλια σίγουρα δεν ευθυγραμμίζονται με τις απόψει του Κοινοβουλίου που έχουν εκφραστεί πολλέ φορές. Ο πρόεδρος της Επιτροπής Βιομηχανίας μπορεί να κάνει ό,τι θέλει βέβαια, με, από προσωπικά, αλλά δεν μπορεί να τα λέει εκ μέρου της Επιτροπής. Στην ομάδα μου μου λένε συνέχεια ότι τέτοια πράγματα δεν μπορεί να τα πει, Δεν μπορεί να ε, βάζει όλη την ομάδα. Δεν είναι η πολιτική αυτή που ακολουθούμε όλοι. Φαντάζομαι ότι το ίδιο που ισχύει στη δικιά μου πολιτική ομάδα ισχύει και γενικότερα στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Κάτλιν Φαν Μπρέντ, θέλεις κάτι? Είμαι μέλος πλήρες της Επιτροπής Βιομηχανίας της ΣΥΤΡΕ. Αυτή τη βδομάδα συνεδριάζουμε μάλιστα. Και είναι πολύ καλό που το είπατε αυτό. Θα το θίξω και θα το συζητήσω και με άλλα μέλη της Επιτροπής Ήτρε της ομάδας μου και από άλλες πολιτικές ομάδες για να δούμε τι θα κάνουμε. Σας ευχαριστώ πολύ. Θα ακολουθήσουμε λοιπόν αυτήν την τακτική. Είναι πραγματικά ασύνηθες να αναφέρεται κατά αυτόν τον τρόπο ένα συνάδελφο, αλλά νομίζω ότι έπρεπε να το συζητήσουμε σήμερα, δεν έπρεπε να το αφήσουμε χωρίς ε, να το σχολιάσουμε. Δεν μπορούμε να μιλάμε ε, για ε, αυτοκτονία, για ένα θέμα το οποίο ε, έχει τεθεί και ως στόχος και από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο εξάλλου η τιμή των εκπομπών διοξιδίου του άνθρακος. Είναι ένα θέμα λοιπόν το οποίο νομίζω ότι αξίζει να συζητήσουμε και να επικρίνουμε. Περνάμε στο σημείο 4 της ημερήσιας διάταξης, προφορική ερώτηση του Γιάννο Σάντερ και Άνια Βάισκερβερ και Jim Higgins. Το σημείο 3 το ξέχασα όμως, έγκριση των πρακτικών της 6 Σεπτεμβρίου. Έχουμε τα πρακτικά. Αν δεν θέλει κανείς να ζητήσει κάποια αλλαγή, θεωρούμε ότι εγκρίθηκαν τα πρακτικά και όντως περνάμε στο σημείο 4, προφορική ερώτηση για την έλλειψη βιταμίνης D. Εδώ έχουμε ανταλλαγή απόψεων με εκπροσώπους της Επιτροπής. Καταρχήν θα δώσω όμως το λόγο στο Γιάννο Σάντερ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ετός ε, τον ε, Απρίλιο, πάνω από 6 μήνες πριν δηλαδή, υλοποιήσαμε μια συνδιάσκεψη ιδιαίτερα επιτυχή στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και μπορέσατε να δείτε μια μπροσούρα. Έχουμε εδώ όλες τις συνέπειες. αυτήν η διάσκεψη ήταν μια πολύ καλή ευκαιρία για να ασχοληθώ με ένα θέμα, καθώς εγώ είμαι νομικό. Έτσι λοιπόν, κατόπιν αυτής ε, της συνδιάσκεψης, ασχολήθηκα με το θέμα αυτό. Καταρχήν θα ήθελα να σας πω ότι η κυρία ε, Βάις και ο κύριος Χίγκιν μου ζήτησαν να απολογηθώ εκ μέρου του γιατί έχουν ανηλυμένε υποχρεώσει. Ήθελα να συμμετάσχουν ε, στην παρουσίαση αυτή γιατί από κοινού υλοποιούμε ε, αυτό το σχέδιο. Όμως, τι θέλω να πω εγώ τώρα, στείλαμε ένα έγγραφο επί της ουσίας σε όλα τα μέλη του Κοινοβουλίου. Υπάρχουν κάποιοι που το έχουν λάβει στην ασπρόμαυρη έκδοση, αλλά νομίζω ότι το ουσιαστικό τμήμα των πληροφοριών υπάρχει. Τουλάχιστον κάθε ομάδα έχει λάβει ένα αντίτυπο. Δεν θα σας παρουσιάσω τώρα όλα τα στοιχεία του εγγράφου, αρκεί να δείτε το έγγραφο. Απλώ θέλω να επικεντρωθώ στα πιο ουσιώδη. Ποιο είναι το πρόβλημα λοιπόν. Όσοι, ακόμη και όσοι δεν είναι γιατροί, ακόμη και οι κοινοί άνθρωποι ε, που ε, ε, ε, ε, μάλλον ακόμη και εκείνοι κοινοί άνθρωποι ενδιαφέρονται για τα ιατρικά ζητήματα και ξέρουμε ότι η βιταμίνη D είναι πάρα πολύ σημαντική έτσι ώστε όλοι οι άνθρωποι πάστα ηλικία να μπορούν να αναπτυχθούν σωστά. Και ξέρουμε ότι με ισορροπημένη διατροφή και αν υπάρχει ήλιος κατορθώνουμε να έχουμε την απαραίτητη ποσότητα βιταμίνης D. Όμως, τι δεν ξέρουμε, τουλάχιστον εγώ το αγνοούσα και πολλοί το αγνοούν ότι η έλλειψη βιταμίνης D αποτελεί την πηγή πολλών νόσων. Δηλαδή μπορεί να προκαλέσει διαβήτη, άσθμα, σκλήρηση κατά πλάκας, παραδείγματος χάρη και υπάρχουν και ορισμένες μορφές ε, καρκίνου που μπορούν να αναπτυχθούν λόγω της έλλειψης βιταμίνης D. Τι αγνοούμε ακόμη, ότι σύμφωνα με μία μελέτη που υλοποιήθηκε πρόσφατα, τουλάχιστον 50% του πληθυσμού στην Ευρωπαϊκή Ένωση υποφέρει από έλλειψη βιταμίνης D. Και κάτι που είναι εντελώ ε, νέο για μένα είναι ότι ορισμένες ε, νόσοι που θεωρούσαμε ότι δεν υπάρχουν πλέον στην Ευρώπη όπως ε, μειοσκελετικές ε, μειοσκελετικά προβλήματα έχουν εμφανιστεί στην Αγγλία λόγου χάρη. Και με πολύ λίγους πρόσθετους σπόρους, με πολύ λίγες δαπάνες μπορούμε να βελτιώσουμε σημαντικά την κατάσταση. Αυτό μπορεί να μας επιτρέψει να εξοικονομήσουμε δαπάνες στον τομέα της υγείας. Έτσι λοιπόν, στην παρουσίαση αυτή στη σελίδα 8 μπορείτε να δείτε ένα διάγραμμα βασίζεται σε μία μελέτη που υλοποιήθηκε πέρσι σε 17 ευρωπαϊκές χώρες και ποιο είναι το αποτέλεσμα ότι με 10 δισεκατομμύρια ευρώ αν δαπανίσουμε αυτό το ποσό για να μειώσουμε την έλλειψη βιταμίνης D στον ευρωπαϊκό πληθυσμό θα εξοικονομήσουμε 187 Έτσι λοιπόν καταλαβαίνετε, αν θα πενήσουμε 10 θα ξεκονομήσουμε 187. Αν ε, ακόμη και το 1 τέταρτο αυτών ε, των αριθμητικών στοιχείων αληθεύουν, τότε καταλαβαίνετε ότι αυτό είναι επαρκής λόγος έτσι ώστε στο εσωτερικό αυτής της ε, Επιτροπής να ακολουθήσουμε την εξίσοδο εδώ, να πάρουμε μέτρα σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση και να υλοποιήσουμε μια εκστρατεία σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Ένωση για να μειώσουμε την έλλειψη σε βιταμίνη D. Πρέπει να έχουμε μια πολιτική για τη δημόσια υγεία πολύ πιο εντατική. Ξέρω ότι ανυπομονείτε πρόεδρε, αλλά βλέπετε και τις ε, ερωτήσεις ε, στις τρεις τελευταίες σελίδες, μπορείτε να τις διαβάσετε. Θα ήθελα να υπογραμμίσω ότι αφενός πάνω από 50% του ευρωπαϊκού πληθυσμού φύγεται από αυτή την έλλειψη βιταμίνης D. Δεύτερον, μπορούμε να εξοικονομήσουμε σημαντικούς πόρους αν έχουμε μία πιο αποτελεσματική πολιτική υγεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Και τρίτον, θέλω να ζητήσω από ε, τους παρόντες, από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να μας υποστηρίξουν έτσι ώστε να μην ασχολούμαστε μόνο εμείς στη δική μας επιτροπή με το θέμα αυτό, αλλά να μπορέσει να συζητηθεί και στην Ολομέλεια. Ξέρετε ότι μια κοινοβουλευτική απόφαση διαφέρει τα μάλα αν συζητηθεί και στην Ολομέλεια και ληφθεί απόφαση εκεί. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον συνάδελφο Γιάννα Σάντερ. Εκπροσωπείτε από τον διευθύντη της DG Σάνκο, Ανδρέα Ρίς. Θα μας πείτε για αυτό το 50% του πληθυσμού με την έλλειψη βιταμίνης Δ και τι μπορούμε να κάνουμε από αυτού. Παρακαλώ, έχετε το λόγο. Thank you. Thank you, uh, Ευχαριστώ. Η Κομισιόν γνωρίζει αυτό το το πόσο σημαντική είναι η βιταμίνη D για διάφορε πτυχέ της δημόσιας υγείας ε, και εδώ μιλάμε για πρόληψη. Συμφωνούμε με την ε, παρουσίαση αυτή θεωρούμε ότι η βιταμίνη D είναι πολύ ουσιαστικό θεραπευτικό συστατικό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή καλωσορίζει τον ενδιαφέρον του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και την υποστήριξη στις δράσεις για την πρόληψη και Θέλω να σας προσθέσω ότι η Κομισιόν γνωρίζει τα πολύ ε, καλά επιδημολογικά δεδομένα που υπάρχουν, ε, όμως ε, τα, δεν έχουμε ακόμη δεδομένα σε σχέση με τις μειοσκελετικέ νόσους και βλέπετε τα αυτά τα στοιχεία στις μελέτες που έχουν γίνει. Και αναφέρθηκε σε αυτά και ο κ. Γιάννος ε, έχουμε την οδηγία 2002-406 και του κανονισμού 1925-2006 όπου προβλέπουν ελάχιστο αριθμό ε, κάποιων θρεπτικών συστατικών και ανόργανων στοιχείων και αυτά ε, θα καθοριστούν σε κάποιες μελέτες που θα γίνουν από την ΑΦΣΑ και από άλλους φορείς και λαμβάνονται από διάφορες πηγές. Επίσης, ε, ε, θα ληφθούν ε, δεόντως υπόψη οι αναφορές που υπάρχουν σε αυτά τα κείμενα. Ε, η Κομισιόν ε, έχει υλοποιήσει σημαντικέ διαβουλευσει με τα κράτη-μέλη και έτσι ενδιαφερόμενε τομεί στον τομέα αυτό. Θα γίνει περαιτέρω προσπαθή να δυσφαλίσουμε ότι είναι διαθέσιμα για τους καταναλωτές ασφαλή προϊόντα προ κατανάλωση και να αποφύγουμε ε, και τις υπερβολικές προσλήψεις αλλά και την έλλειψη βιταμίνη D. Η Ευρωπαϊκή η Αρχή Ασφάλειας των Τροφίμων ζητήθηκε να παράσχει επιστημονικά δεδομένα για την επικαιροποίηση ε, των στοιχείων που είχαμε από το 1992 για την πρόσληψη του πληθυσμού για τα όργανα στοιχεία και τις βιταμίνες και το τέλος του 2012 ε, ε, αναμένεται να ελοποιηθεί αυτό το έργο. Όταν η Κομισιόν θα έχει λάβει τη γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ, θα σκεφτεί αν οποιαδήποτε δράση χρειάζεται να ληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης και για τις πρόσθετες μελέτες που σκεφτόμαστε να συζητήσουμε στο σημερινό πρόγραμμα για την υγεία θα είναι δύσκολο να έχουμε περαιτέρω μελέτες, κυρίως αν ε, ε, θέλετε να έχουμε νέες κλινικές δοκιμές, γιατί έχουμε περιορισμένους πόρους για τα επόμενα έτη. Αλλά θα πρέπει να το σκεφτούμε αυτό και για το μελλοντικό πρόγραμμα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Ρης. Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Η πρώτη μου αντίδραση όταν διάβασα αυτό το κείμενο ήταν ότι εξεπλάγην για το κείμενο της ερώτησης. Σκέφτηκα μήπως πρόκειται για διαφήμιση ή για τα συμπληρώματα διατροφής. Γιατί έχουμε συζητήσει πόσο προσεκτικά πρέπει να δίνουμε πληροφορίες στους ασθενείς παραδείγματο χάρη και εξεπλάγει από τη διατύπωση αυτής της ερώτησης και αυτό πρέπει να το δηλώσω καταρχήν. και δεν συζητώ αυτή τη στιγμή το ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και το ρόλο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής μετά τη συνθήκη της Λισαβόνας. Ε, θέλουμε να έχει αρμοδιότητα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή για θέματα υγείας. Αλλά μπορεί να είμαι εγώ η μόνη που το επιθυμώ αυτό και αναρωτιέμαι τι θέλουμε. Θέλουμε να έχει αρμοδιότητα η Επιτροπή και σε ποιους τομείς. Είναι δύσκολο το ερώτημα και πρέπει να προσέξουμε ε, να δώσουμε μια ειλικρινή απάντηση. Τώρα θα ήθελα να περάσω στο περιεχόμενο, στην ουσία της ερώτησης. Αρκετοί συνάδελφοι, ο συνάδελφο Λίζη, ο Κρίς Ντέιβις, πριν από λίγα χρόνια θα θυμάστε ότι κάναμε μια συζήτηση για τα συμπληρώματα διατροφής Και είχαμε συζητήσει και το θέμα της επιτρεπόμενη ημερήσιας ποσότητα. Η Εμίλια Μιούλερ ήταν η εισηγήτρια εκείνη την εποχή και θυμάμαι ήταν λίγες εκθέσεις που ήταν τόσο αντιφατικές, όπου δημιουργήθηκε τόσο μίσος ε, και τόσες επιθέσεις ε, εναντίον του εισηγητού, εναντίον της κυρίας Μιλή προσωπικά εκείνη την εποχή. Η συνιστόμενη ημερήσια ε, ποσότητα για μια συγκεκριμένη βιταμίνη, για κάποιες ανόργανες ουσίες, πώς πρέπει να καθορίζονται. Αρχίζουμε τώρα μέσα σε μια υφιστάμενη νομοθεσία να βγάζουμε κάποια συστατικά, διότι υπάρχει σχετική νομοθεσία. Εδώ αφορά την βιταμίνη Δέλτα Και το ερώτημα ποιες ε, βιταμίνες ε, βοηθούν και μια μεγαλύτερη δόση τους θα βοηθούσε ε, την θεραπεία του καρκίνου ή την πρόληψη του καρκίνου. Αυτά είναι θέματα τα οποία επιστημονικά είναι ιδιαίτερα αντικρουόμενα. Και ρώτησα και γιατρούς τι πρέπει να κάνει κανείς, να πάρει βιταμίνη Δ, να πάρει βιταμίνη Ε, τι να πάρει. Και η απάντηση ογκολόγων ήταν πάρα πολύ κατά περιπτώσεις διαφορετική. Δεν είμαι γιατρός και είμαι πάλι πολύ προσεκτική σε αυτά τα οποία λέω. Εάν πιστεύουμε ότι η οστεοπόρωση μια νόσο των οστών είναι μεγάλο πρόβλημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, θεωρώ ότι είναι σωστό να ασχοληθούμε με το σοβαρό πρόβλημα και να βάλουμε στο κέντρο της συζήτησης την ασθένεια, όχι μια πιθανή λύση, και αν βάλουμε την ασθένεια στο επίκεντρο των συζητήσεων και πούμε ότι το πρόβλημα είναι η οστεοπόρωση και μπορούμε να πούμε ότι ε, μπορεί η βιταμίνη Δ να αντιμετωπίσει την έλλειψη ασβεστίου, θα ήταν προτιμότερο και θα προτιμούσα να δω κάτι τέτοιο στα υποστηρικτικά έγγραφα. Να μιλάμε 10 λεπτά ηλιακό φως ε, το χειμώνα μπορεί να φτάνει για την απορρόφηση της βιταμίνης Δ για τους ασθενείς. Δεν διαφωνώ να ασχοληθούμε με συγκεκριμένες ασθένειες, αλλά διαφωνώ να βγάζουμε από την νομοθεσία ένα συγκεκριμένο κομμάτι και να ασχολούμεθα με αυτό. Γιατί τη βιταμίνη Δ και όχι τη βιταμίνη Σ τη βιταμίνη Ε, γιατί να θέλουμε κάτι συγκεκριμένο για τη βιταμίνη Δ. Ε, αν πιστεύουμε ότι πρέπει να αναθεωρήσουμε την οδηγία για τα μέσα διατροφής, να το κάνουμε, να ζητήσουμε από την Επιτροπή να μας υποβάλει μια νέα πρόταση και να συζητάμε και τη βιταμίνη Δ και τη βιταμίνη Ε και τη βιταμίνη Σ που έχουμε πολλά να πούμε να το βάλουμε στην ημερήσια διάταξη και να το συζητήσουμε. Διαφορετικά θα σας έλεγα να είμαστε πάρα πολύ προσεκτικοί και σας παρακαλώ να μην φτάσει στην Ολομέλη. Να το συζητήσουμε στην Επιτροπή πρώτα. Ευχαριστώ πολύ. Θυμάμαι και εγώ τη μάχη για τη βιταμίνη C πριν από χρόνια. Οι υπέρμαχοι της βιταμίνης C είχαν ε, ε, κατακλείσει με 10.000 email ε, τους υπολογιστές του Κοινοβουλίου ήταν ιδιαίτερα αντιφατικό το θέμα και η οδηγία για την ε, συνιστόμενη ημερήσια ποσότητα ή την εγκεκριμένη ημερήσια ποσότητα ε, είχε δημιουργήσει ε, μεγάλες εντάσεις. Δεν βλέπω κανέναν άλλον όμως να θέλει το λόγο για αυτό το συναρπαστικό θέμα. Να δώσω ξανά το λόγο στον κύριο Ρίς. Όχι, ο Κρίς Ντέιβις. Εδώ με την κυρία Μάνα συζητάω που είναι αναπληρώτρια εδώ, που στην ομάδα μου παίζει σημαντικό ρόλο. Εδώ άκουσα για την βιταμίνη Δέλτα στην Ευρώπη. Στη Φιλανδία δεν είναι έτσι, από ό,τι μου λέει. Λέμε ότι μπορεί να χρειάζονται κάποια πρόσθετα αλλά αυτά είναι εντελώ διαφορετικά ανάλογα με τη χώρα στην οποία βρισκόμαστε. Είναι δύσκολο λοιπόν για όλη την Ευρώπη να πούμε το ίδιο. Διαφέρουν οι κλιματικές συνθήκες, η ηλιοφάνεια. Οπότε πρέπει όλοι να έχουμε βαζάκια με συμπληρώματα διατροφής. Εσείς, Πρόεδρε, σε κοινοβουλευτικό επίπεδο, τι πρέπει να οργανώνετε. Μήπως ότι πρέπει να οργανώνετε λίγο γυμναστική το μεσημέρι έξω στον καθαρό αέρα για τους ευρωβουλευτές. Θέλω να πω ότι υπάρχουν τόσο πολύ διαφορετικές πρακτικές που θα μπορούσε κανείς να προτείνει σαν σημείο εκκίνησης πριν προχωρήσουμε περισσότερο. Uh, ισορροπημένη διατροφή και ισορροπημένος ε, τρόπος ζωής ε, σίγουρα βοηθάνε ε, στην απορρόφηση των βιταμινών, αλλά υπάρχουν πολλοί άνθρωποι που δεν έχουν ούτε ισορροπημένο τρόπο ζωής, ούτε ισορροπημένη διατροφή. Και γι' αυτό μια καμπάνια ενημέρωσης, μια εξαιρετική ενημέρωσης δεν είναι κακό. Τώρα δεν ξέρω αν μας βοηθάει και αν μας οδηγεί στο να επιτύχουμε τους στόχους μας. Αυτό είναι άλλο ερώτημα η πρόληψη ε, των ασθενειών και η ε, διατήρηση καλής υγείας είναι σαφώς μια προτεραιότητα. Θέλει κανείς το λόγο για τη βιταμίνη Δ, κυρία Μάνερ, από τη Φινλανδία όπως ακούσαμε, όπου αντιμετωπίζεται το θέμα εντελώς διαφορετικά από ό,τι στο Ηνωμένο Βασίλειο, όπως μας είπε ο κ. Ντέιβις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πράγματι, μόλις έφτασα στην Επιτροπή αυτή, δεν γνωρίζω καλά το περιεχόμενο της συζήτησής σας. Άποψή μου όμως είναι ότι είναι περίεργο να συζητάμε τόσο πολύ για μία βιταμίνη. Και συμφωνώ με τη συνάδελφο Ροτ Μπέρεντ ότι αυτό το ζήτημα πρέπει να συζητιέται γενικότερα. Όπως λέει και ο κύριος Στεφής, συζητάμε για πρακτικές που είναι διαφορετικές από χώρα σε χώρα. Εξάλλου, τα πρώτα χρόνια ζωής του κάθε παιδιού είναι πολύ σημαντικά, ανάλογα με τη δόση σε βιταμίνη Δ που παίρνει δηλαδή. Στη Φιλανδία, τα ανώτατα όρια, οι συνιστόμενες δηλαδή μερίσιες τροφικές δόσεις, είναι πολύ πιο χαμηλές από ό,τι σε άλλες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Οπότε πρέπει να δούμε πρώτα ποιε είναι οι συστάσει για τι σωστές δόσεις που δίνονται σε κάθε χώρα. Μην ξεχνάμε ότι αν υπάρξει παραπάνω δόση βιταμίνης από όσο πρέπει, μπορεί να προκληθούν βλάβες. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε μια γενικότερη συζήτηση το πόσο βιταμίνη Δ πρέπει να παίρνουμε είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί και το χαιρετίζω. Αλλά πρέπει πρώτα να γίνει συζήτηση και για αυτή τη βιταμίνη αλλά και για άλλες. Σας ευχαριστώ πολύ για την παρέμβασή σας. Να δώσω το λόγο ξανά στον κύριο Ρης. Θέλετε να απαντήσετε κύριε Ρης. Uh, Συμφωνώ απόλυτα για το ότι πρέπει να περιμένουμε μελέτες. Υπάρχει ΕΦΣΑ από τη μια μεριά που κάνει μελέτες, η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων, αλλά όχι μόνο. Όντως πρέπει να δούμε ποια είναι η καλή ισορροπία ανάμεσα στον ήλιο, στην έκθεση στον ήλιο δηλαδή, ε, να δούμε τι μπορεί να προσφέρουν ε, δίαιτες με συμπληρώματα διατροφής και άλλους παράγοντες πρέπει να λάβουμε υπόψη μας. υπάρχουν ε, και ειδικέ κατηγορίες στον πληθυσμό, όπως είναι οι ηλικιωμένοι ή τα μωρά. Ε, η κάθε περίπτωση απαιτεί μια διαφορετική λύση. Πώς να το πετύχουμε αυτό, εμείς θέλουμε στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή να συνεχίσουμε να δουλεύουμε, να ενημερωνόμαστε από την Ευρωπαϊκή Αρχή και έτσι να προχωρήσουμε προς το μέλλον. Ο Γιάννος. Έχει το λόγο ο Γιάννος Άντερ. Ευχαριστώ. Μετά από τις παρατηρήσεις που άκουσα, έχω να πω το εξής. Πολλοί είπαν ότι υπάρχει έλλειψη και σε άλλες βιταμίνες. Οπότε δεν ε, πρέπει να ασχοληθούμε μόνο με την έλλειψη σε βιταμίνη Δ, αλλά να καλύψουμε και άλλες βιταμίνες. Σε αυτό έχω να απαντήσω ότι δεν είμαι καθόλου κατά του να εξετάσουμε και την έλλειψη σε άλλες βιταμίνες. Όμως το γεγονός ότι υπάρχει ένα συγκεκριμένο πρόβλημα για το οποίο έχουμε μια λύση, υπάρχουν επιστημονικά Ινστιτούτα που έχουν εκπονήσει μελέτες. Υπάρχει το έγγραφο αυτό το οποίο σας ε, μοίρασα, το οποίο βασίζεται σε επιστημονικές μελέτες. Άρα δεν είναι κάτι στο οποίο έχω καταλήξει έτσι μου ήρθε Όχι. Το ότι υπάρχουν και άλλα προβλήματα δεν σημαίνει ότι εμεί δεν πρέπει να ασχοληθούμε με αυτό το ειδικό πρόβλημα. Εξάλλου, δεν ασχολείται μόνο η Ευρωπαϊκή Ένωση. Από όσο γνωρίζω εγώ, αρχές Δεκεμβρίου θα δημοσιευθεί μία μελέτη και στις Ηνωμένε Πολιτείες στις Ηνωμένες Πολιτείες μπήκε στην ημερήσια διάταξη τον τελευταίο καιρό αυτό το θέμα και θα έχουμε τα αποτελέσματα μιας πολύ προθυμένης επιστημονικής μελέτης. Γι' αυτό σκέφτηκα ότι θα έπρεπε και οι ευρωβουλευτές να μπορέσουν να εξετάσουν το θέμα αυτό. Πρόκειται για μια ρύθμιση που την αποκτήσαμε πριν από 20 χρόνια και που κατέληξε σε μια οδηγία όχι για την υγεία, αλλά για κάτι άλλο. Για να καθοριστεί η ποσότητα που χρειάζεται σε βιταμίνη Δ ο οργανισμός μας. Όλοι οι ερευνητές συμφωνούν ότι χρειαζόμαστε τουλάχιστον 3 με 4 φορές παραπάνω ποσότητα. Άλλοι, μάλιστα, μιλάνε για 10 φορές παραπάνω. Οπότε, τη στιγμή που 50% του ευρωπαϊκού πληθυσμού παρουσιάζει έλλειψη σε βιταμίνη Δ και που η έλλειψη βιταμίνα Δ οδηγεί σε διαφορετικές ασθένειες, ε, αυτό σημαίνει ότι αποτελεί παράγοντα κινδύνου η έλλειψη σε βιταμίνη Δ. Εγώ δεν ε, θέλω εδώ να μιλήσω όμως για ασθένειες, θέλω να μιλήσω για πρόληψη. Γιατί είμαστε πεπισμένοι ότι η πρόληψη είναι πάρα πολύ χρήσιμη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να έχει μια ενιαία πολιτική με εκστρατεία ενημέρωσης του κοινού, αλλάζοντας τους κανόνες εκεί που χρειάζεται, γιατί όπως είπαμε η ρύθμιση αυτή είναι... ξεκινήσει από 20 χρόνια. Αλλάζουν τα πράγματα, αλλάζουν τα δεδομένα. Και από την άλλη η έλλειψη αυτή κοστίζει και εκατομμύρια στον Ευρωπαίο φορολογούμενο. Γι' αυτό σας ζήτησα να ζυγίσουμε τα υπέρ και τα κατά. να δούμε το υγειονομικό αποτέλεσμα από τη μια και το οικονομικό αποτέλεσμα από την άλλη. Πρέπει να τα μελετήσουμε και τα δύο για να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ελπίζω η Ευρωπαϊκή Επιτροπή να προχωρήσει. Σας ευχαριστώ πολύ για τις ερωτήσεις και για την ενδιαφέρουσα συζήτηση. Θα ασχοληθεί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή με το θέμα και θα ακούσουμε τα σχετικά αποτελέσματα. Για την υγεία για να μπορέσει να ασχοληθεί και η Επιτροπή μας με το θέμα της ε, υγείας. Περνάμε στο στο επόμενο σημείο της μέσης διάταξης, το σημείο 6 ε, για τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης που το συζητάμε μαζί με το σημείο 5. Ίσως ε, να μπορέσουμε σήμερα να ρίξουμε λίγο φως στο θέμα και επειδή εδώ έχουμε ανταλλαγή απόψε με την Επιτροπή, ο κύριος Ρίς μπορεί να μας πει τι μπορούμε να κάνουμε. Έχετε το λόγο και πάλι. Uh, try to combine Πρόεδρε, θα προσπαθήσω εδώ να απαντήσω από κενού στα δύο θέματα αυτά η οδηγία που τροποποιεί την οδηγία 2009 κάθετος 883 σε σχέση με τα φαρμακευτική προέλευση για την ε, ανθρώπινη χρήση και παρέχει μια απλή διαδικασία καταχώρησης για τη θέση στην αγορά. Σήμερα έχει μεταφερθεί στο εσωτερικό δίκαιο οδηγία για όλα τα κρατημέλη και η Κομισιόν θεωρεί ότι τα εμπόδια έχουν ε, αρθεί για αυτά τα φάρμακα, φάρμακα προέλευσης. Ε, ε, τα τελευταία κράτη-μέλη που μετέφεραν το οδηγία στο ιστορικό της δίκαιο ήταν το 2008. Έτσι λοιπόν όλα τα κράτη-μέλη σήμερα ε, στο καθεστώς λειτουργεί η δυνάμη αυτής της οδηγίας. Σε ό,τι αφορά τώρα τα δεδομένα που μελετούμε για τη διαδικασία αυτή, Η Κομισιόν εξέδωσε μία ανακοίνωση το 2008 την 584 ότι η συστηματική αίτηση για γενικά στοιχεία αγώνιδιο τοξικότητας έκανε δύσκολη την καταχώρηση γιατί γενικά αυτά τα στοιχεία δεν ήταν διαθέσιμα. Η Κομισιόν θεώρησε ότι αυτή η προσέγγιση οδήγησε στο μικρό αριθμό των αιτήσεων που έχουν ληφθεί μέχρι τώρα έτσι λοιπόν, το Δεκέμβριο του 2009 η Επιτροπή για τα φυτικά φάρμακα εξέδωσε μια κατευθυντήρια γραμμή όπου προτείνει να εισαχθούν κάποιες δοκιμές ε, για μια αντιπροσωπευτική σειρά ε, υλικών προκειμένου οι παρασκευαστές να κάνουν μόνοι τους τις δοκιμές για συγκεκριμένα σκευάσματα μια συνεργασία πρωτοβουλίας ε, με τον τομέα για γενικά στοιχεία γονιδιοτοξικότητας υποστήριξε τη διαδικασία για τις ε, καταχωρήσεις σε εθνικό επίπεδο και ελπίζουμε ε, έτσι η διαδικασία αυτή να κινηθεί στα πλαίσια της Επιτροπής και σε επίπεδο εθνικού φορέα χορήγηση τη άδεια. Ε, η ερώτηση αφορά τις απλοποιημένε διαδικασίες καταχώρηση για τα προϊόντα. Η τελική έκθεση ε, στάλει από την Κομισιόν στο Συμβούλιο και στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο το Σεπτέμβριο ε, το 2010 περιμένουμε απαντήσεις από Συμβούλιο και Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Κομισιόν ε, δεν έχει κάνει κάποια περαιτέρω δράση σε σχέση με την απλοποιημένη διαδικασία και δεν προβλέπεται τώρα τροποποίηση της οδηγίας. Σε ό,τι αφορά τα παραδοσιακά προϊόντα για την κυβερνητική και την ε, Κινηζική ιατρική, ο κανόνας που αφορά την εφαρμογή της οδηγίας του 2004-24 ε, διευκολύνει την θέση στην αγορά των φυτικών προϊόντων, όμως θα πρέπει αυτά τα προϊόντα να χρησιμοποιούνται εδώ και 30 χρόνια και να υπάρχουν στην αγορά της Ευρωπαϊκής Ένωσης για 15 χρόνια. Αυτή είναι η μόνη διαφορά σε σχέση με τα άλλα προϊόντα με τα ευρωπαϊκού τύπου προϊόντα. Σε ό,τι αφορά τώρα πρόσθετες ερωτήσεις για το πόσα προϊόντα εξακολουθούν να συμπεριλαμβάνονται στις διαδικασίες. Η απλή απάντηση είναι ότι δεν γνωρίζουμε. Γιατί η διαδικασία είναι αποκεντρωμένη τους επόμενους μήνες θα προσπαθήσουμε να συνεργαστούμε με την Επιτροπή για να έχουμε μια πλήρη εικόνα και αυτό συζητήθηκε την περασμένη εβδομάδα στο Λονδίνο, δηλαδή πώς θα οργανώσουμε τη διαδικασία για να έχουμε μια πλήρη εικόνα σε σχέση με την εφαρμογή. Σε ό,τι αφορά τώρα στα προϊόντα, τα αριθμητικά στοιχεία που λάβουμε στο τώρα είναι τα εξής στην ανακοίνωση που δημοσιεύσαμε το 2008 μιλούσαμε για 110 αιτήσει σε 17 κράτη-μέλη και σύμφωνα με, τη βιομηχαν... με τις ενώσεις ε, της βιομηχανίας του τομέα περίπου 200 ε, προϊόντα φυτικής προέλευσης έχουν εγγραφεί σήμερα, έχουν καταχωρηθεί σήμερα αλλά δεν είναι ίση κατανομή σε στα κράτη-μέλη. Κάποια κράτη-μέλη είναι πιο ενεργά και χρησιμοποιούνται περισσότερο αυτά τα προϊόντα για την καταπολέμηση διαφορών νόσων, ενώ σε κάποια άλλα κράτη-μέλη δεν υπάρχει τέτοια ισχυρή παράδοση. Έτσι λοιπόν, σε αυτό το στάδιο αυτές τις πληροφορίες έχω να δώσω. Ευχαριστώ να απαντήσω σε πρόσθετες ερωτήσεις αν υπάρχουν. Ευχαριστώ. Θα δώσω το λόγο στο Μπασάικ Χουντ. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Επιτροπή για τις απαντήσεις της. Όμως νομίζω ότι παραμένουν ε, κάποια ζητήματα παρά όλες αυτές τις απαντήσεις που μας έδωσε. Γιατί τι ακούμε, ακούμε ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή συμφωνεί ότι το συστηματικό αίτημα που γίνεται, ότι ακόμα δηλαδή και με την απλουστευμένη διαδικασία καταχώρησης εξακολουθούν να μπαίνουν εμπόδια, Συγχρόνως, από τον Απρίλιο του 2011, όλα τα φάρμακα και τα παραδεσιακά πρέπει να καλύπτουν τις προϋποθέσεις. Άρα υπάρχει ένα πρόβλημα από τον Απρίλιο και μετά. Είπατε ότι η Επιτροπή αναγνωρίζει ότι το 2008 ήδη και δεν υπήρχε απάντηση από την Επιτροπή μας και το Κοινοβούλιο ίσως να είναι αλήθεια. Πάντως σήμερα οι πολίτες εκφράζουν ιδιαίτερη ανησυχία. Τι θα γίνει με αυτά τα προϊόντα. Και δεν έχω καταλάβει συγκεκριμένα, δεν άκουσα συγκεκριμένα τι θα γίνει μετά τον Απρίλιο του 2011 εφόσον η οδηγία αυτή τεθεί πλήρως εφαρμογή. Ποια θα είναι η συνέπεια για προϊόντα όπως για παράδειγμα παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής που ακολουθούν μια πιο ολιστική προσέγγιση. Δεν θα επιτρέπεται η πρόσβασή του στην αγορά. Αυτή είναι η συγκεκριμένη ερώτηση. Και αν η απάντηση είναι πως δεν θα μπορούν να έχουν πια πρόσβαση στην αγορά, τότε γιατί η Ευρωπαϊκή Επιτροπή δεν σκέφτεται αν μη τι άλλο να παρατείνει την περίοδο για την ρύθμιση αυτή, ώστε μετά τον Απρίλιο του 2011 να μπορούν τα προϊόντα αυτά να κυκλοφορούν στην αγορά. Ένα άλλο θέμα τώρα. Αναγνωρίζετε επίση ότι μπορεί να υπάρξει πρόβλημα για παραδοσιακά ε, προϊόντα, τα οποία χρησιμοποιούνται εδώ και πάρα πολύ καιρό εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση. Γιατί εσεί είπατε ότι πρέπει να κυκλοφορούν 15 χρόνια μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Αν όμως χρησιμοποιούνται περισσότερο εκτό Ευρωπαϊκή Ένωση, αυτό γιατί δεν μετράει. Γιατί δεν θεωρείται και αυτή μια χρήση. Γιατί πρέπει να είναι μόνο στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Το ερώτημα είναι, γιατί να μην εξετάζετε κατά περίπτωση το καθέτημα. Εσείς λέτε ότι πιστεύετε πως θα υπάρξει μια ομαλή προσαρμογή. Ναι, αλλά πρέπει να είμαστε σίγουροι ότι θα είναι έτσι, γιατί τον Απρίλιο θα έχει λήξει το ζήτημα. Και το άλλο, γιατί κοιτάτε αποκλειστικά τα φυτικά προϊόντα και τίποτα άλλο, όχι αυτά που έχουν ανόργανα συστατικά, και μήπως θα έπρεπε να κοιτάξετε όχι μόνο τα φάρμακα, αλλά και άλλα που να, ε, να έχουν μια άλλη προσέγγιση, σοφρολογική για παράδειγμα ή κάτι άλλο. Υπάρχει δυνατότητα αναβολής της προθεσμίας του Απριλίου. Είναι πολύ συγκεκριμένες οι ερωτήσεις μου και ελπίζω να πάρω και συγκεκριμένες απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ο κύριος Ρης. Συγγνώμη, Όντω θέλω να απαντήσω συγκεκριμένα. Προ το παρόν δεν θέλουμε να αναβάλουμε την ημερομηνία για αργότερα για την εφαρμογή τη οδηγία αυτή. Η οδηγία αυτή θα τεθεί σε εφαρμογή. Τα κράτη-μέλη έχουν θέσει τις ε, ημερομηνίες. Υπήρξε κάποια παρεξήγηση για τον τρόπο με τον οποίο προχωρούν οι καταχωρήσεις. Εμείς κάνουμε ό,τι μπορούμε να βοηθήσουμε και βοηθούμε τους ε, ετούντες Όντω, για να υπάρξει μια ομαλή διαδικασία από τη στιγμή που υποβάλλουν την αίτηση καταχώρησης των φοιτικών τους προϊόντων ε, στην αντίστοιχη επιτροπή. ώστε να μπορέσουν να προσαρμοστούν στην οδηγία. Στην οδηγία θέτουμε επίση και τον κανόνα για τα 15 χρόνια που πρέπει να κυκλοφορεί στην ευρωπαϊκή αγορά ή 30 χρόνια γενικότερα χρήση για την αγιουρβεδική και την παραδοσιακή κινέζικη ιατρική. Σε ορισμένε περιπτώσεις για τα ανόργανα συστατικά, αν δεν είναι η κύρια ουσία στο προϊόν, τότε μπορεί να εμπίπτει στον ε, κανόνα. Αν λοιπόν υπάρξουν επιπλέον προβλήματα με τον αριθμό των καταχωρήσεων, πρέπει να δούμε πώς θα προχωρήσουμε και πώς θα βοηθήσουμε τους ε, ετούντες για να περάσουν και από το εθνικό επίπεδο. Κύριε Ροτμπέρντ, ευχαριστώ πολύ. Ας προσπαθήσουμε να το ξαναδούμε το θέμα και από το παρελθόν. Ακούσαμε αυτά που μας είπε ο κύριος Ρης. Μας είπε ότι δεν νομίζω ότι μπορεί να παραταθεί η προθεσμία για την καταχώρηση. Εξάλλου, λογικό είναι αυτό, γιατί αυτό αποτελεί η νομοθεσία. Δεν μπορεί ο κύριος Ρή να μα πει τώρα μόνο του ότι θα αλλάξει νομοθεσία. Δεν θα ήταν λογικό να μα πει ότι κάτι που αποφασίσαμε στο πλαίσιο της συναπόφαση μπορεί να αλλάξει. Ε, εγώ ήμουν σκιώδη εισηγήτρια για την έκθεση τη και όχι μόνο η και αλλά εμείς είχαμε δώσει το έναυσμα για την νομοθεσία. Είχαμε ζητήσει από την Επιτροπή να καταρτήσει σχετική, σχετικό νομικό μέσο και η Επιτροπή δεν το έκανε με μεγάλη τη χαρά και διήρκεσε και μεγάλο χρονικό διάστημα. Και από τότε που είχαμε το νομικό μέσο στη διάθεσή μας πάλι σε μεγάλο χρονικό διάστημα μέχρι να μπορέσει μετά τη συζήτηση στο Λονδίνο ε, να περάσει σε μονογραφίες ε, για τα φυτικά μέσα. Όλα διήρκεσαν πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Και σε όσους δεν γνωρίζουν το θέμα θέλω να πω ότι έχω ασχοληθεί με πολλά θέματα. Ήταν ένα από τα πιο δύσκολα θέματα που μας είχε απασχολήσει. Υπήρχαν πολύ διαφορετικές απόψεις στο Κοινοβούλιο. Ε, υπήρχαν αυτοί οι οποίοι μιλούν για τη δυνατότητα επιλογής των ασθενών, οι οποίοι θα πρέπει να μπορούν να επιλέξουν μεταξύ διαφόρων μεθόδων παραδοσιακής ιατρικής, ολιστικής προσέγγισης κλπ. Και ε, είπαμε ότι για τα φυτικά ε, μέσα θα πρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα να συμπληρώνουν την ιατρική αντιμετώπιση και μάλιστα για ε, ήπια θέματα. Ο κύριος Λίζε θα μπορεί να μας τα επιβεβαιώσει αυτά και σε σχέση με αυτά τα οποία πιστεύει η παραδοσιακή ιατρική. Αυτά τα οποία, στα οποία καταλήξαμε έδειξαν ότι ο κύριος Νίστικο και εγώ χρειάστηκε να, επιβάλλουμε, να τα επιβάλλουμε. Είπαμε ότι είναι δύσκολο ε, να χειριστούμε τα φάρμακα φυτικής προέλευσης, οπότε ας μην ακουμπήσουμε καν τα θέματα ανθρωποσοφιστικής φιλοσοφίας και παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής. Έχω πολλούς φίλους που ασχολούνται με την ομοιοπαθητική ιατρική και ε, τα θέματα ε, αυτά αποτελούν αντικείμενο διαφορετικής ε, νομοθεσίας. Και ε, είναι άλλη κατηγορία αυτά τα οποία συζητάμε τώρα για τα, φυτικά, για μέσα φυτικής προέλευσης. Είναι εντελώ διαφορετική κατηγορία προϊόντων. Και ο κ. Σέκερ και ο κ. Σποκ τώρα έχουν θέσει ερωτήσεις που αφορούν τα νομοθετικά κείμενα. Έχουμε όντως μία απλουστευμένη διαδικασία καταχώρησης για τα μέσα φυτικής προέλευσης. Απλουστευμένη διαδικασία διότι τα μέσα φυτικής προέλευσης ε, είναι διαφορετικά από τα χημικά φάρμακα ε, και δεν μπορούμε εύκολα να αποδείξουμε την αποτελεσματικότητα. έχουμε δηλαδή απόδειξη ότι είναι αποτελεσματικά. Στα χημικά φαρμακευτικά προϊόντα είμαστε πιο αυστηροί Ζητάμε απόδειξη αποτελεσματικότητας ε, και πρέπει να απαιτούμε να αποδεικνύουν τα χημικής προέλευσης φάρμακα ότι είναι πιο αποτελεσματικά από άλλα φάρμακα. Ε, γι' αυτό δίνουμε μια ε, δυνατότητα, ένα προνόμιο στα μέσα φυτικής προέλευσης να μην χρειάζεται να έχουν τόσο βαριά διαδικασία, να έχουν μια απλουστευμένη διαδικασία. Λαμβάνουμε υπόψη τις ε, πτυχές ε, ασφάλειας και η ε, πτυχή της ασφάλειας λέει ότι υπάρχει παραδοσιακή προσέγγιση ότι έχουν χρησιμοποιηθεί τόσα χρόνια στην Ευρωπαϊκή Ένωση και είπε και ο κύριος τι γίνεται στο 16 γάμα 4 όταν το προϊόν λιγότερο από 15 χρόνια όταν χρησιμοποιείται στην Ευρωπαϊκή Ένωση λιγότερο από 15 χρόνια. Εγώ πιστεύω ότι ε, συνεχίζει να ισχύει αυτό το οποίο ισχύει και νομίζω ότι δεν χρειάζεται να αλλάξει κάτι από αυτού επί, της, ε, επί των όσων ε, ισχύουν για την προθεσμία. Προσπάθησα να ερευνήσω το θέμα όταν είδα την ερώτηση για να δω τι γίνεται σε σχέση με την θέση σε εμπορία. Όντως, ορισμένα προϊόντα μπορεί να μην υπόκεινται στην απλουστευμένη διαδικασία. Αλλά δεν μπορεί κανείς να υποχρεώσει τον ετούντα. Αν κάποιος δεν θέλει να καταφύγει στην απλουστευμένη διαδικασία, είναι δικαίωμά του να μην καταφύγει σε αυτή τη διαδικασία. Και σε διάφορα προϊόντα που έχουν συγκεκριμένα βιολογικά ή χημικά συστατικά, μπορεί ο κατασκευαστής, ο παρασκευαστής να αποφασίσει αν θέλει να επιλέξει την α ή τη β διαδικασία. Τα παραδοσιακά φάρμακα φυτικής προέλευσης από το 2004 έχουν μια επταετή προθεσμία για τη ε, διαδικασία έγκρισης. Αυτή η προθεσμία το 2004 λήγει το 2011. δεν ξέρω γιατί κάποιος ε, δεν ασχολήθηκε με το θέμα επί 7 χρόνια. Μπορεί κάποιος ε, να αποκοιμήθηκε και να μην ε, ενημερώθηκε, αλλά νομίζω ότι οι σύλλογοι ενημερώνουν τα μέλη του εγκαίρω. Μια άλλη πιθανότητα είναι να υπάρχει κάποιο ζήτημα με την ποιότητα των ε, φαρμακευτικών προϊόντων. Δεν μπορώ να το γνωρίζω. Μπορεί να μην θέλουν τη διαδικασία καταχώρησης ε, γιατί δεν έχουν ακόμη επαρκώς εξετάσει τα θέματα ποιότητας. Η άλλη εναλλακτική λίστα ήταν ότι είναι ένα σύνθετο φάρμακο ένα φάρμακο φυτικής προέλευσης που έχει όμως και ανόργανα συστατικά, όπως είπε ο κύριος Ρή. Μπορεί να περιλαμβάνει και άλλα ανόργανα συστατικά, οπότε θα πρέπει να θεωρηθεί όπως τα φάρμακα χημικής προέλευσης και ισχύουν διαφορετικά θέματα. Όπως και τότε που είχαμε συζητήσει για τα συμπληρώματα διατροφής, ένας παραγωγός ε, βιταμίνης C μας είχε ε, πραγματικά ασκήσει μεγάλο πόλεμο. Δεν ξέρω μήπως ο κύριος Ρής θέλει να μας πει αν σκέφτεται η Επιτροπή ε, να μας ε, υποβάλει και πρόταση για τα φάρμακα ανθρωποσοφιστικής προέλευσης ή ομοιοπαθητικής ή παραδοσιακής κινέζικης ιατρικής. Ευχαριστώ πολύ. Άφησε την Τάγμα να μιλήσει περισσότερο χρόνο για να μας υπενθυμίσει τη συλλογική μνήμη της Επιτροπής μας, μιας και υπάρχουν και νεότεροι στην Επιτροπή μας. Ε, και εγώ έχω λάβει παρόμοιες επιστολές όπου πολλοί φοβούνται ότι παραδοσιακά γιατροσόφια της γιαγιάς όπως χαμομήλι και φασκόμηλο θα, θα απαγορευτούν στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν νομίζω ότι πρέπει να φοβόμαστε όμως ε, ότι ε, τέτοια προϊόντα θα πρέπει να καταχωρηθούν και αν δεν καταχωρηθούν δεν θα μπορούμε πια να τα πίνουμε. Και υπάρχουν και εταιρείε που δεν είναι εταιρείε. Και πολλοί ανησυχούν ότι από τον Απρίλιο του 2011 προϊόντα ομοιοπαθητικής ε, και ανθρωποσοφιστικής δεν θα μπορούν να χρησιμοποιούνται ε, γιατί θα χρειάζεται διαφορετική διαδικασία καταχώρησης. Γι' αυτό θέλαμε τις καταχωρήσεις. Ο Κρίς Ντέιβις. Ε, ναι, Πρόεδρε, για την ερώτηση που μόλις θέσατε και εγώ ήθελα να αναφερθώ. Thank you, Mr. President. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εδώ δεν θέλω να μιλήσω για τις ε, βιταμίνες και για τα συμπληρώματα διατροφές, αλλά για τα προϊόντα φυτικής προέλευσης. Θέλω και εγώ να ακούσω την απάντηση στην ερώτηση που τέθηκε ταυτόχρονα. Συμφωνώ με, πώς, μέσα όσο υπόθηκαν από τη συνάδελφο στο τέλος. Ε, η Κομισιόν ε, προτίθεται να παρουσιάσει μια συγκεκριμένη νομοθετική πρόταση για τα μειοποθετικά φάρμακα και τα παραδοσιακά φάρμακα γιατί πιστεύω ότι αυτό είναι κάτι πολύ σημαντικό τουλάχιστον ε, εμείς στην Ελλάδα έχουμε πλούσια βιοπικιλότητα και έχουμε πάρα πολλά βότανα, έχουμε πάρα πολύ μεγάλες δυνατότητες ε, και για τη θεραπεία και αυτό είναι πολύ σημαντικό για το ποιο είδος θεραπείας ε, κάποιος επιλέγει και επίσης ε, έχουμε και τη δυνατότητα ανάπτυξης ε, ε, βιώσιμων εφόρων πρακτικών στη θεραπεία. Έχουμε τώρα κάποιες επιχειρήσεις που ε, παρασκευάζουν φυτικά σκευάσματα και είναι καλό το ότι ζητάμε από τους ανθρώπους να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες. Ήδη ξεκίνησαν να αναλαμβάνουν πρωτοβουλίες και οι άνθρωποι ανησυχούν για το πώς θα εφαρμοστεί αυτή η νομοθεσία. Έτσι λοιπόν είναι πολύ σημαντικό να έχουμε μια ειδική νομοθεσία για την παραδοσιακή ιατρική και για τα φάρμακα φυτικής προέλευσης. Και επίσης να δούμε αν κατά τη διαδικασία προπαρασκευής αυτής της νομοθεσίας, αν θα μπορούσαμε να συζητήσουμε και για μια μεταβετική περίοδο για την εφαρμογή σε σχέση με αυτά που έχουμε σήμερα. Ευχαριστώ. Κύριος Uh, για να απαντήσω στην ερώτηση τι θα γίνει με τα προϊόντα που δεν θα μπουν ε, στη διαδικασία αυτή υπό την οδηγία δηλαδή για τα παραδοσιακά προϊόντα φοιτικής προέλευσης θα παραμείνουν στην αγορά τα προϊόντα αλλά δεν θα μπορούν να ονομάζονται προϊόντα φοιτικής προέλευσης γιατί δεν θα έχουν λάβει άδεια από αυτό το καθεστώ. Θα μπορούσαν ε, να ενταχθούν σε άλλε κατηγορίε προϊόντων στην αγορά. Σε ό,τι αφορά τι πρωτοβουλίε τη Κομισιόν για τα παραδοσιακά φάρμακα, ε, μπορούμε να καλύψουμε όλα ε, τα είδη προϊόντων, ανθρωποσοφιστικής προέλευσης ε, για την κινέζικη ιατρική κτλ. Μέχρι τώρα δεν σχεδιάζουμε να αναλάβουμε νομοθετική δράση, νομοθετική πρωτοβουλία σε αυτό το τομέα. Όπως ε, γνωρίζετε έχουμε αρκετά φορτωμένη ατζέντα και ε, στοχεύουμε στο μέλλον να αναθεωρήσουμε την νομοθεσία για τα κτηνιατρικά φάρμακα ε, και είναι αυτό ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που θέλουμε να παρουσιάσουμε στο Κοινοβούλιο και στο Συμβούλιο. Σας ευχαριστούμε πολύ. Ωραία. Το συζητήσαμε λοιπόν αυτό το θέμα και θα συνεχίσει να μας απασχολεί. Παρακαλώ, κυρία Ροτμπέρεντ. Ο κύριος Ρης απάντησε στην ερώτησή μου γιατί δεν κατάλαβα. Απαντήσατε στην ερώτηση της Ντάγμαρ. Σε ό,τι αφορά την ρυθμιστική πρωτοβουλία για τα παραδοσιακά φάρμακα. Εκτός μικροφώνου, μιλήτρια. Δηλαδή πείτε απλώ ναι, αυτό θα ήταν καλό. Κοιτάξτε, πολύ θα ήθελα να πω ναι, γιατί εγώ όταν σπούδαζα ε, ήμουν και στην Ινδία και μελέτησα αυτό το θέμα. Αλλά είναι πάρα πολύ δύσκολο για μας ε, να, να παρουσιάσουμε μια τέτοια πρωτοβουλία σε αυτό το στάδιο του σχεδιασμού της ανάληψης νομοθετικών πρωτοβουλειών. Μάλλον όχι ήταν η απάντηση, λέει ο πρόεδρο, παρά ναι. Η απάντηση είναι θα ήθελα, αλλά μάλλον δεν μας επιτρέπεται. Πολλές ερμηνείες. Ναι, θα ναι, σας ακούσουμε για ένα σχόλιο για να επικεντρωθώ στο τελευταίο είδος απάντησης που δόθηκε, που είναι κατά κάποιο τρόπο όχι. Ήθελα να ξέρω τι συνέβη, γιατί το 2008 η Κομισιόν Εκθεσίτης δήλωσε ότι η καταλληλότητα ενό ξεχωριστού νομικού πλαισίου για προϊόντα ορισμένη παράδοση θα πρέπει να αξιολογηθεί. Τώρα λέτε δεν το πράττουμε αυτό, ούτε καν μια αξιολόγηση πλέον. Τι έγινε λοιπόν από το 2008 μέχρι σήμερα, αυτή είναι η ερώτησή μου. Not, not much happened in this Δεν έγιναν και πολλά από τότε. Και εγώ αυτό νόμιζα. Μιλητής, αλλά κοιτάξτε, αν ε, υπάρχει έκκληση από το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο να γίνουν περισσότερα πράγματα, από και η Κομισιόν ε, είναι υπεύθυνη να απαντήσει και φυσικά θα προετοιμάσει μια έκθεση αξιολόγηση. Αλλά η απάντησή μου αφορούσε την ομοθετική πρωτοβουλία και όχι την ε, αξιολόγηση. Κάτι τέτοιο μπορεί να γίνει τα επόμενα έτη. Θα πρότεινα να κάνει η Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ ένα ταξίδι στην Ινδία για να τα εξετάσει τα θέματα επιτόπου. Λοιπόν, σοβαρευόμαστε και περνάμε στο σημείο 8 της μέσης διάταξης. Α, στο σημείο 7. Στο σημείο 7 της μέσης διάταξης προφορική ερώτηση της Κορίν Λεπάζ σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για την αξιολόγηση των κινδύνων για την υγεία από γενετικώς τροποποιημένους οργανισμούς. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Κύριε Πρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αγαπητοί συνάδελφοι, ένα από τα πιο σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς είναι η αξιολόγηση κινδύνων για την υγεία και για το περιβάλλον. Αν κοιτάξουμε την ε, οδηγία του 2008, διαπιστώνουμε ότι απαιτεί ανάλυση κινδύνου, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα, των άμεσων και των έμεσων κινδύνων, των συσσωρευτικών ε, επίσης ε, δράσεων. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι οι ρυθμίσεις αυτές δεν έχουν τηρηθεί, και γι' αυτό μάλλον το Συμβούλιο ομόφωνα το Δεκέμβριο του 2008 ζήτησε ενίσχυση της αξιολόγησης κινδύνου όσον αφορά τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, κάτι το οποίο επανέλαβε και το Συμβούλιο της 14ης Οκτωβρίου του 2010. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το 2010 ενέκρινε μία πρόταση με στόχο να διευκρινίσει περισσότερο τι δεδομένα πρέπει να δίνει η ΕΦΣΕ, Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια Τροφίμων, νέους κανόνες δηλαδή, κατευθυντήριες γραμμές τόσο για την υγεία όσο και για το περιβάλλον. Ένα μέρος πάντως της επιστημονικής κοινότητας αλλά και πολλές χώρες μέλη πιστεύουν ότι οι νέες αυτές κατευθυντήριες γραμμές δεν ενισχύουν την αξιολόγηση αλλά αντίθετα αποδυναμώνουν τις απαιτήσει που υπήρχαν ε, και υπάρχουν μέχρι τώρα και που έτσι καλλιώς δεν φτάνουν, δεν είναι αρκετές. Εδώ δεν θέλω να μπω σε λεπτομέρειες, θέλω όμως να σας πω ότι οι μελέτες που θα έπρεπε βάσει του σημείου 25 της οδηγίας να δίνονται δεν δίνονται, ότι οι βιολογικές επιπτώσεις που στατιστικά έχουν νόημα όσον αφορά τους γενετικά τομένους οργανισμούς ε, δεν γίνονται όπως πρέπει γιατί γίνονται σε ποντικούς αλλά όχι σε μεγάλο αριθμό ζώων και μόνο για 90 μέρες ενώ για τα παρασιτοκτόνα γίνονται εξελογήσεις για δύο ολόκληρα χρόνια. Ξέροντα ότι εκατομμύρια ζώα πρόκειται να καταναλώσουν γενετικά τροπομένου οργανισμού, προτίθεται η Επιτροπή να αυξήσει τον αριθμό των ποντικών που επιβάλλονται σε μελίτε και να παρατείνει τη διάρκεια των μελετών σε 24 μήνες αντί για όπως προβλέπεται και για τα φυτοφάρμακα. Σκοπεύει επίσης να αναθέσει τη διεξαγωγή τοξικολογικών δοκιμών επί της αναπαραγωγής των γενετικά τροπημένων οργανισμών, καθώς και συναφών διαγενελογικών δοκιμών, έτσι όπως διατυπώνεται στην οδηγία του 2010 αλλά που ε, δεν ε, τηρείται προς το παρόν. Οι κατευθυντήριες γραμμές, εξάλλου, παρουσιάζουν και έλλειψη στατιστικής αξιοπιστίας όσον αφορά τις ε, αναλύσεις ταξικότητας. Αυτό το ζητάματος επαλήθευσης της ισχύως των θεστικών δοκιμών, μόνο εφόσον η μέθοδος τοξικολογικής ανάλυσης που χρησιμοποιείται δείχνει την ύπαρξη ψευδών θετικών αποτελεσμάτων, ενώ δεν προβλέπεται σχετική επαλήθευση για τις δοκιμές που θα μπορούσαν ενδεχομένω να παρέχουν ε, ψευδό αρνητικά αποτελέσματα. Οι θετικέ είναι πολύ πιο σπάνιε, οι αρνητικέ είναι πιο συχνέ. Διαπιστώνουμε εξάλλου ότι αποδυναμώνεται η διατύπωση. Το κείμενο γίνεται λιγότερο δεσμευτικό και ε, παφιόμεθα στις επιχειρήσεις να καθορίσουν πώς ε, θα προσφέρουν προστασία, ενώ ο στόχος προστασίας είναι ένα πολιτικό θέμα που θα έπρεπε να αποφασίζουν οι δημόσιες αρχές. Οι ελλείψει αυτέ και οι χαλαρέ διατάξει που προβλέπονται από τι ανατοέρω αναθεωρημένε κατευθυντήριε γραμμέ αντιβαίνουν στα συμπεράσματα του Συμβουλίου του 2008, το οποίο ζήτησε ακριβώ το αντίθετο. Δεν επιτρέπουν να έχουμε αποτελέσματα αδιαφυσβήτητη αξιοπιστία. Και είναι απαράδεκτο η έγκριση αυτού του κειμένου να προχωρήσει χωρί διαφάνεια και χωρί ευρεία συζήτηση. Οπότε η ερώτηση μου είναι εξή. Μπορεί η Επιτροπή να εξηγήσει με ποιο τρόπο θεωρεί ότι εν λόγω νέε κατευθυντήριε γραμμέ ανταποκρίνονται στι απαιτήσει του Συμβουλίου, με ποιο τρόπο ενισχύουν την αξιολόγηση του υγειονομικού κινδύνου των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών και δεν χαλαρώνουν τι απαιτήσει απέναντι στι επιχειρήσει που διαθέτουν γενετικά τροποποιημένους οργανισμού στην αγορά. Τρίτη πτυχή τη ερώτησή μου είναι το θέμα τη διαχείριση κινδύνου. Η Επιτροπή πρέπει να διασφαλίσει την ε, ορθή διενέργεια της αξιολόγησης κινδύνων. Γιατί αν δεν γίνεται ορθά η διενέργεια της αξιολόγησης κινδύνου, δεν μπορούμε να έχουμε και σωστή αξιολόγηση κινδύνου. Συνεπώ, η Επιτροπή πρέπει να διασφυλίσει ότι οι επιστημονικές επιφυλάξεις αναγνωρίζονται και αναφέρονται στη γνωμοδότηση της ΕΑΤ, όπω ορίζεται η οδηγία του 2001-18. Για ποιο λόγο δεν έχει μεριμνήσει η Επιτροπή για την εφαρμογή των απαιτήσεων της οδηγίας αυτή σχετικά με την αξιολόγηση και για ποιο λόγο δεν ποτέθεσε η Επιτροπή στη νέα το ερώτημα σχετικά με το γεγονό ότι δεν έχει αναγνωρίσει καμία επιστημονική επιφύλαξη, εξορμέ μια περίπτωση, ότι υπάρχουν πολλέ τέτοιε επιστημονικέ ε, επιφυλάξει. Πώ αντιλαμβάνεται η Επιτροπή το ρόλο τη ω διαχειρίστρια κινδύνου, καθώ και την εφαρμογή τη αρχή τη προφύλαξη. Τέλο, τι προτείνει η Επιτροπή για να μα διασφαλίσει μια διαδικασία εμπειρογνωμοσύνη αξιόπιστη, αμερόλεπτη, διαφανή και απελεγμένη από σύγκρουση συμφερόντων που πολύ συχνά τα βλέπουμε τελευταία. Ευχαριστώ. Όλες αυτές τις ερωτήσεις υποβάλλουμε στον κύριο Πούτλεϊ, Διευθυντή από τη Γενική Διεύθυνση ΣΑΝΚΟ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Εισαγωγικά να πω ότι η Κομισιόν ε, και ο Επιτροπός ε, Νταλή συμφωνούν απόλυτα με, τις, ε, με τα τελευταία λόγια τη κυρία Λεπάζ για την αξιολόγηση που έγινε από την ΕΦΣΑ, την Ευρωπαϊκή Αρχή για την ασφάλεια του τροφίμων. Εμεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκή Επιτροπή αναγνωρίζουμε ότι χρειαζόμαστε μια επιστημονική ανάλυση από την ΕΦΣΑ, η οποία να είναι διαφανή και αμερόληπτη και αξιόπιστη. Φυσικά το έχει επαναλάβει επανειλημμένο και ο Επίτροπο. Δεν υπάρχει κανένα ερώτημα λοιπόν σχετικά και πρέπει να βελτιώσουμε την κατάσταση γιατί είναι αλήθεια ότι αναγνωρίζουμε ότι υπάρχουν σημεία προς βελτίωση. Για να απαντήσω τώρα στις διάφορες ερωτήσεις της κυρίας Λεπάζ και καταρχήν την πρώτη η αξιολόγηση των γενετικά τροποποιημένων οργανισμών είναι μια συγκριτική αξιολόγηση. Συγκρίνει ένα φυτό γενετικά τροποποιημένο με ένα κανονικό φυτό, με ένα συμβατικό φυτό ε, και συγκρίνει τα χαρακτηρισμό, τα χαρακτηρισμό της γενετικής τροποποίησης δεν ε, έχουμε την ίδια περίπτωση με τα παρασιτοκτόνα. Για ορισμένε περιπτώσει έχουμε για τα παρασιτοκτόνα μελέτε τοξικότητα που φτάνουν ω και Μπορούμε όμω να μιλήσουμε και για την ε, σπονγκοδή κεφαλοπάθεια, όπου έχετε τέτοιε μελέτε τοξικότητα μακροπρόθεσμε που φτάνουν μέχρι και τα 10 χρόνια. Όλοι λοιπόν εξαρτώνται από το είδο τη νόσου, από το χαρακτήρα τη νόσου εδώ για του ε, γάμματα φωμικρών δεν ε, έχουμε πρόβλημα τοξικότητας παρόμοιο. Ε, γιατί ξέρετε ότι οι φωμικρών ε, στην πλειονότητά τους είτε είναι φυτά ανθεκτικά στα ζυνοκτώνα είτε ανθεκτικά στις νόσους και ενίοτε και στα έντομα. Αυτά που ανθίστανται στα έντομα αξιολογούνται σύμφωνα με τις ίδιες αρχές που έχουμε και για τα παρασιτοκτόνα έχουν τις ίδιες ιδιότητες. Δηλαδή έχουμε τα ε, BT που σκοτώνουν ε, τα έντομα και έχουμε τις ίδιες διαδικασίες αξιολόγησης μεταξύ των κανονικών παραστοκτόνων BTAF, BT και των γενετικά τροπομένων φυτών BT. Είναι λοιπόν ε, ίδιες ε, διαδικασίες αξιολόγησης. Είναι αλήθεια όμως ότι έχουμε μελέτες ε, ε, στους ποντικούς ε, ε για τις 90 ημέρες, όχι για όλα, γιατί πολλές φορές η ΕΦΣΑ δεν θεωρεί ότι είναι απαραίτητο, αλλά άλλες φορές θεωρεί ότι είναι απαραίτητο. Και αυτό είναι ο προβληματισμό που υλοποιούμε αυτή τη στιγμή. Δεν έχουμε όμως ε, ολοκληρώσει τον προβληματισμό μας για να δούμε τι θα κάνουμε με αυτή τη μελέτη των 90 ημερών. για μια πιο μιακοπρόθεσμη μελέτη 24 μηνών όπως ε, θέλει η κυρία Λεπάς ε, για τους αρουραίους. Δηλαδή να τρέφονται τα ποντίκια με γάματα φόμικρον επί 24 μήνες. Για να γίνει κάτι τέτοιο θα πρέπει να έχουμε διαδικασίες δοκιμών που να έχουν επικυρωθεί σε κοινοτικό επίπεδο βεβαίως αλλά και σε διεθνές επίπεδο δεν θα έπρεπε να ζητήσουμε μελέτες 24 μηνών ε, όταν ε, δεν αναγνωρίζονται από καμία επιστημονική κοινότητα στον κόσμο. Θα πρέπει όλοι να εργαστούμε από κοινού για να μπορεί να γίνει κάτι τέτοιο, αλλά για αυτό το πρωτόκολλο των 90 ημερών ε, εξετάζουμε αυτή τη στιγμή πώς θα το ενισχύσουμε. Ερώτηση παριθμών 2. Για το σχεδίο κανονισμού που χαλαρώνει τους κανόνες της ΕΦΣΑ. Τους αποδυναμώνει. Εμείς δεν έχουμε την ίδια άποψη, πιστεύουμε, ότι πρόκειται για ενίσχυση των σημερινών κανόνων σε πολλαπλά επίπεδα. Καταρχήν, σε νομικό επίπεδο. Γιατί σήμερα μιλάμε για κατευθυντήριες γραμμές που δεν είναι δεσμευτικές. Ενώ, αν ε, έχουμε θέτηση μέσω ενός κανονισμού της Κομισιόν, Αυτές οι κατευθυντήριες γραμμές ε, καθίστονται νομικά δεσμευτικέ και αυτό δίνει νομικό πλεονέκτημα. Επίσης, θεωρούμε ότι έχουμε ενίσχυση της αξιολόγησης ε, από επιστημονική σκοπιάς, γιατί συμπεριλαμβάνονται στόχοι που πρέπει να πληρούνται για κάθε στάδιο της ε, αξιολόγησης κινδύνων. Έτσι λοιπόν για την καθολική αξιολόγηση Ισχύει αυτό και έχουμε και το πρωτόκολλο που αναγνωρίζεται σε διεθνέ επίπεδο. Επιμένουμε τα μάλα στο ότι δεν πρέπει να φανταζόμαστε πράγματα που κανείς δεν αναγνωρίζει σε διεθνέ επίπεδο. Εμείς στην πραγματικότητα επιθυμούμε αυτή η διεθνή συνεργασία να μπορεί να καταστεί πιο συγκεκριμένη μέσω των κατευθυντηρίων γραμμών, προκειμένου οι αξιολογήσει της ΕΦΣΑ ε, να μην είναι δυνατόν να αμφισβητηθούν σε διεθνές επίπεδο. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό. Κατόπιν. Θεσπίζεται ένα πρωτόκολλο για τις ε, δοκιμές ε, στους αγρούς και με αυτές τις συγκριτικές αναλύσεις, με συγκεκριμένους κανόνες για τις στατιστικές αναλύσεις. Πιστεύουμε ότι αυτό προβαίνει στην ενίσχυση των κανόνων δεν ε, έχουμε ε, κάποια σημεία που να έχουν καταργηθεί σήμερα. Πιστεύουμε ότι υπάρχει ενίσχυση, ίσως όχι προς την κατεύθυνση που επιθυμεί η κυρία Λεπάζ για την ε, δοκιμή των 24 μηνών, αλλά εμεί πιστεύουμε ότι ενισχύσαμε το σημερινό πρωτόκολλο. Για την ερώτηση 3. Για τους μικροπρόθεσμους κινδύνους. Θεωρούμε ότι είναι σημαντικό να ξεκαθαρίσουμε και θα το πράξουμε μάλιστα σε κάποιο άλλο νομοθέτημα να προβλέψουμε ένα monitoring, μια εποπτεία όταν θα έχει δοθεί άδεια στο γενετικά τροποποιημένο οργανισμό. Είναι σημαντικό να θεσπίσουμε ένα αριθμιστικό πλαίσιο για να μπορέσουμε να κάνουμε την παρακολούθηση των πτυχών της καλλιέργειας όταν θα έχει δοθεί άδεια στο γενετικά τροποποιημένο οργανισμό. Για να επανέλθουμε στο θέμα της αδειοδότησης. Νομίζω ότι δεν πρέπει εδώ να μπλέκουμε τις απόψεις με μειοψηφίας με τις επιστημονικές γνωμοδοτήσεις. Κοιτάξτε, εμφισβητεί τα πράγματα. Η επιστήμη αυτή είναι και η αρχή της. Αλλά γι' αυτό συνεχίζεται η έρευνα και η πρόοδος. Αν πούνε οι επιστήμονες ότι δεν αμφισβητούν, δεν αμφιβάλλουν πλέον, σταματούν να ερευνούν και δεν έχουν και βρήματα. Για μας η επιστημονική βεβαιότητα αποτελεί τμήμα του πανοράματος της επιστήμης. Όμως, ε, οι απόψεις της μειοψηφίας είναι επίσης σημαντικές. Όπως λέει η κυρία Λεπάς, ε, είχαμε μόνο και μία γνωμοδότηση της Ευρωπαϊκής Αξίας Ασφαλής των Τροφίμων, της ΕΦΣΑ, για τους γάμματα φόμικρον, όπου περιλαμβανόταν μία μειοψηφική άποψη σε σχέση με την ανθεκτικότητα ε, στα αντιβιωτικά. κάθε μέλος του επιστημονικού πάνελ έχει την ευθύνη να διασφαλίσει αν συμφωνεί, ότι συμφωνεί ή όχι με τη γενική άποψη του πάνελ, καθώς εμείς θέλουμε το πάνελ να εκδίδει μη γνωμοδότηση που θα τη χάνει μεγαλύτερες μεγαλύτερης δυνατής τη μεγαλύτερη δυνατή συνένεση. Γιατί στην ίδια έχουμε μία ε, πλειοψηφική άποψη που λέει άσπρο και μία ε, μειοψηφική άποψη που λέει μαύρο. Είναι πολύ δύσκολο για το διαχειριστή το κινδύνου, δηλαδή την Κομισιόν, να φτάσει σε μια απόφαση. Έτσι λοιπόν, ε, κατά τη διάρκεια τη επιστημονική αξιολόγηση, ζητάμε κατευθείαν από την ΕΦΣΑ να ξεκαθαρίσει αυτό το σημείο. Ζητούμε η ΕΦΣΑ να ξανασυζητήσει με τους επιστήμονες που είχαν αυτή τη μειοψηφική άποψη, έτσι ώστε να δοθούν καλύτερες εξηγήσεις και να προσπαθήσουμε να κατανοήσουμε γιατί υπήρξε αυτή η μειοψηφική άποψη. Και να ενταχθεί στη γενική γνωμοδότηση του πάνελ. Δηλαδή δεν αρνούμαστε την άποψη της μειοψηφίας, απλώς θέλουμε ξεκάθαρες γνωμοδοτήσεις που να μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε στη συνέχεια γιατί θα τις έχουμε κατανοήσει ορθά και θα μπορούμε να τις μεταφράσουμε σε μια ξεκάθαρη νομοθεσία. Και γι' αυτό το λόγο υπάρχουν λίγες αρνητικές απόψεις για τους γαμματαφόμικρων και γι' αυτούς τους λόγους αυτές οι γνωμοδοτήσεις καθυστερούν. Ξέρετε ότι οι βιοτεχνολογικές εταιρείες κατηγορούν την Κομισιόν και την ΕΦΣΑ ότι πολλές φορές χρειάζονται τρία και πέντε χρόνια για την κατάρτιση της νομοδότησης. Γιατί κάθε φορά που υπάρχουν είτε βεβαιότητες είτε με ψηφικές απόψεις, αντί να δοθεί μια αρνητική γνωμοδότηση, η ΕΦΣΑ συνεχίζει να εργάζεται ε, σε αντίθεση με το τι γίνεται σε άλλου τομεί, όπω για τα παραστοκτόνα όπου η ΕΦΣΑ, ε, παραδείγματο χάρη, εκδίδει αμέσω μία αρνητική γνωμοδότηση. Και είδαμε ένα παράδειγμα σήμερα με το Α3D, ε, A3D, με μια, ένα παραστοκτόνο που συζητήθηκε στο Συμβούλιο σήμερα το πρωί και δεν ε, τοποθετήθηκε το Συμβούλιο και η Κομισιόν θα πρέπει να δράσει στο ίδιο πλαίσιο με τη διαδικασία γαματόφα ομικρών για να το αποκλείσει από τον κατάλογο των ε, αδειοδοτημένων παραστοκτών γιατί υπήρξαν αιτήματα από την εταιρεία να δοθεί μια παράτηση για να παρουσιάσει προς τα στοιχεία και η είπε όχι. Έτσι λοιπόν ακολουθούμε τη γνωμοδότηση της ΕΦΣΑ. Ενώ στο σχηματογραφό μικρούν ε, δεν το πράττει. Ζητά πρόσθετες πληροφορίες στην εταιρεία και γι' αυτό το λόγο είχαμε είτε λίγες ε, μειοψηφικές ε, απόψεις, ε, είτε καθόλου αρνητικές απόψεις. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την Ευρωπαϊκή Επιτροπή για τη λεπτομερή απάντησή της. Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί όταν μιλάμε για απόψει μειοψηφία και πλειοψηφία πάνω σε αυτό το ζήτημα. Για τον απλούστατο λόγο ότι πολλέ από τι μελέτες δεν είναι εντελώ ανεξάρτητες από τη βιομηχανία. Είναι πιο εύκολο να έχουμε μια μελέτη για γενετικά τροπημένους οργανισμού όταν έχουμε πρόσβαση και άδεια από την επιχείρηση που τους χρησιμοποιεί. Πρέπει λοιπόν να αξιολογήσουμε όχι μόνο το πόσες μελέτες έχουμε, αλλά να δούμε και τι αποδείξεις έχουμε για την ανεξαρτησία των μελετών αυτών. Συμφωνώ λοιπόν με την κυρία Λεπάζ και με τις προτάσεις της. Δεν μας ε, δεν κατηγορούμε ότι δεν έχουν γίνει αρκετά, αλλά ότι δεν τηρούμε την αρχή της προφύλαξης. Ότι γίνεται έγκριση χωρίς να υπάρχουν τέλειες διαδικασίες όσον αφορά την αξιολόγηση των γενετικά δεδομένων οργανισμών. Και ένα άλλο ζήτημα τώρα. Όπως ε, και οι σοσιαλιστές είχαμε μια κρόαση και η ΕΦΣΑ παραδέχεται ότι υπάρχει ένα θέμα με τις ε, αντίστοιχες ποσότητες. Φαίνεται ότι δεν είναι αποτελεσματική αυτή η αρχή των ισοδύναμων τιμών, ισοδύναμων της σύγκρισης που γίνεται ανάμεσα στους γενικά οργανισμούς και τις παραδοσιακές καλλιέργειες. Θέλω όμως μια διευκρίνηση. Στο διαδίκτυο ακούμε πολύ ότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σκέφτεται να σταματήσει την ε, εφαρμογή της μηδενική αρχής για τους γενικά τροπομένους οργανισμούς. Υπάρχει κανένα τέτοιο νέο από πλευράς Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Είναι ενδιαφέρον να έχουμε μια γενική συζήτηση για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αλλά λόγω έλλειψης χρόνου θα πρέπει να περιοριστούμε στα συγκεκριμένα ερωτήματα και στη συγκεκριμένη ερώτηση της κυρίας Λεπάζ, αλλιώς δεν θα μας φτάσει ο χρόνος. Μπαρτ που και ο ίδιος έχει στο επόμενο σημείο μια ερώτηση και του δίνω το λόγο τώρα. Ευχαριστώ. Θέλω κι εγώ να παρέμβω για την ερώτηση αυτή για την ερώτηση της κυρίας Λεπάς. Πολύ συγκεκριμένα μιλάει για κινδύνους επί της υγείας. Η Επιτροπή, λοιπόν, βλέπουμε ότι δεν μπορεί εύκολα να απαντήσει για τις αξιολογήσεις, για τις συγκριτικές μελέτες, ότι είναι αλλιώς ε, από ό,τι με τα εντομοκτώνα, έπειτα αναφέρθηκε και στο ρόλο της ΕΦΣΑ. Όμως, ακούγοντας την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, πραγματικά ε, νιώθω κι εγώ ότι λείπουν συγκεκριμένα δεδομένα. Αρχές αυτού του μήνα υπάρχει μια θετική γνωμοδότηση, για παράδειγμα της ΕΦΣΑ για ένα συγκεκριμένο προϊόν, της Μονσάντο και της Dow AgroSciences, για τον, ε, το καλαμπόκι υπό την επωνομασία Smart που επιτρέπεται η εμπορία του με την έρευνα που έγινε η ΕΦΣΑ καταλήγει σε αποτελέσματα από μεμονωμένες περιπτώσεις και όχι από το συνδυασμό. Γιατί μπορεί κάλλιστα βλέπετε να υπάρχουν μεμονωμένα αποτελέσματα που δεν βλάπτουν την υγεία, αλλά σε συνδυασμό το ένα με το άλλο, ναι, να βλάπτουν την υγεία. Γι' αυτό λοιπόν είναι πολύ σωστό αυτό που θέτει η κυρία Λεπάζ δεν θα πρέπει έτσι χωρίς δισταγμούς να κοιτάμε αυτές τις ε, υποθέσεις. Αντίθετα, πρέπει πολύ συγκεκριμένα να μας απαντήσει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή σε αυτήν την πολύ συγκεκριμένη ερώτηση της κυρίας Λεπάς για τον συνδυασμό παραγόντων. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Η κυρία Χριστίνα Κουτιέρης έχει το λόγο. Ευχαριστώ. Ε, η συνάδελφος εδώ, η κυρία Γιούσο, που έχει το λαιμό της και δεν μπορεί να μιλήσει, μου ζήτησε να πω και μερικά πράγματα και εκ μέρους της. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, δεν μπορεί να τα βάζουμε με τους πανεπιστημιακούς των πανεπιστημίων μας ε, και με τα ερευνητικά κέντρα και να λέμε ότι επηρεάζονται από την ε, βιομηχανία. τη βιομηχανία που παράγει γενετικά τροπημένους οργανισμούς. Νομίζω ότι υπάρχουν πάρα πολλοί ερευνητές που δουλεύουν πάνω στους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς και κανένας από όλους αυτούς δεν έχει πει ότι υπάρχουν και κίνδυνοι. Αυτό όμως που συμβαίνει είναι ότι υπάρχουν και μελέτες που λένε ότι διάφοροι ε, φυσικοί οργανισμοί βλάπτουν την υγεία, που δεν είναι γενετικά τροποποιημένοι. Η πατάτα για παράδειγμα, που μερικές φορές έτσι έχει μια τρυπούλα ε, δημιουργεί μεγάλο πρόβλημα στις εγγύους, αν φάνε τέτοια πατάτα. Μην έχουμε την αίσθηση ότι η φύση δεν ελοχεύει κινδύνους. Αυτό είναι ένα. Έπειτα, θέλω να οργανώσουμε ακρόαση εδώ με ερευνητές οι οποίοι ερευνούν που να είναι ανεξάρτητοι και να μας εξηγήσουν τα επιχειρήματά τους. Γιατί αυτό που είπε ο πράσινος συνάδελφος για τους διάφορους παράγοντες και τα προϊόντα, το συνδυασμό τους, εγώ όταν μιλάω με επιστήμονες γι' αυτό μου λένε ότι όχι δεν ισχύει και μου εξηγούν γιατί. Εγώ δεν έχω την επιστημονική γνώση για να σας το εξηγήσω, εκείνοι όμως μου το εξηγούν και δεν έχουν καμιά σχέση με τις επιχειρήσεις. Η επιστήμη έχει προχωρήσει αρκετά. Δεν είναι ε, η φύση που μας προστατεύει από όλα και εμείς την καταστρέφουμε. Όχι, την δυσχυδή ράχη την προκαλεί αυτό που σας είπα που υπάρχει μέσα ε, στην πατάτα. Δεν είναι ότι τα γενετικά τροπημένα δημιουργούν το πρόβλημα και ότι η φύση δεν δημιουργεί κανένα πρόβλημα. Όχι. Γι' αυτό να οργανώσουμε ακρόαση εδώ. Το δηλώνω επίσημο ότι το ζητάω από τον πρόεδρο. Ευχαριστώ. Δεν έχουμε χρόνο και γι' αυτό σας παρακαλώ να μην μακρηγορείτε, όχι να πω δύο λεπτά, ούτε καν δύο λεπτά. Βικτώρια Πρόντι. Ευχαριστώ. Συγγνώμη που καθυστέρησα, αλλά καθυστέρησα το αεροπλάνο μου. Θα προσπαθήσω να είμαι πάρα πολύ σύντομος. Εγώ προσωπικά δεν βλέπω να ενέχονται κίνδυνοι στους ε, γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, αλλά το κύριο πρόβλημα μπορεί να είναι ότι κατά κάποιο τρόπο μπορεί να εξαρτηθεί η διατροφή ολόκληρου του πλανήτη από ένα περιορισμένο αριθμό ποικιλιών και επομένως το να θέσουμε σε κίνδυνο την περίπτωση που έχουμε επίθεση παρασίτων την διατροφική ασφάλεια. Εγώ νομίζω ότι αυτό είναι ο μεγάλος κίνδυνος που ενέχεται εδώ και νομίζω ότι θα πρέπει εμείς να λάβουμε μέτρα κατά αυτού του κινδύνου μέσω της διασφάλισης ενός ελάχιστου αριθμού ποικιλιών. Γιατί δεν μπορούμε να εξαρτώμαστε, ε, να εξαρτώμε τη διατροφή ολόκληρης της ανθρωπότητας από ε, ένα πολύ περιορισμένο φάσμα ποικιλιών. γιατί εδώ μπορεί να διακυβεύεται πραγματικά η ε, διατροφική ασφάλεια, αν περιορίσουμε δηλαδή υπερβολικά τις ποικιλίε. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Λεπάζ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Κύριε Πούτλη, στην απάντησή σας ε, κυρίως μιλήσατε για τη συγκριτική αξιολόγηση και την αντιστοιχία ουσιών. Αυτό χρησιμοποιείται και στις Ηνωμένες Πολιτείες ακριβώς για να μην γίνουν μελέτες ε, και να μην, ε, δεν, δεν επαφιέμεθα στα αμερικανικά πρωτόκολλα γιατί δεν υπάρχουν τέτοια πρωτόκολλα. Ε, στην οδηγία 2018 όμως δεν λέει ότι εφαρμόζεται η αρχή της ισοδυναμίας ουσιών και γι' αυτό δεν γίνονται μελέτες. Ζητούνται μελέτες για τις άμεσες και έμεσες επιπτώσεις βράχη πρόθεσμα και μακροπρόθεσμα για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς χωρίς να αναφέρεται αυτή η αρχή. Αυτή είναι η πρώτη μου παρατήρηση. Δεύτερον, κάτι που με ανησυχεί. Το, το θέμα των συγκριτικών μελετών αξιολόγησης για να μην πούμε αντιστοιχεία ουσιών γιατί το ίδιο πράγμα με άλλα λόγια λέμε ο κύριος Χάρη Κούιπερ που προεδρεύει της Επιτροπής Γενετικά Τροποποιημένων Οργανισμών ε, έχει αποκαλυφθεί ότι έχει σχέσεις με το χώρο και αν δούμε ε, τις προτάσεις ε, του κύριου Κούιπερ και τις αντίστοιχες εταιρείε, βλέπουμε σαφώς ότι υπάρχει αυτό το θέμα των ισοδύναμων ουσιών. Κύριε Πούντλη, νομίζετε ότι εφαρμόζουμε την οδηγία 2001-18 εφαρμόζοντας αυτή την αρχή. Εγώ δεν είμαι καθόλου βέβαια για κάτι τέτοιο και για να είμαι και σύντομη όπως ζήτησε ο Πρόεδρος, η συνένεση σε επιστημονικό επίπεδο τι σημαίνει, ότι διαγράφουμε τις απόψεις της μειοψηφία ε, και φροντίζουμε ε, να τις τυλίγουμε σε ένα γενικό αποτέλεσμα. Εγώ ε, θέλω να σας πω ότι ως διαχειριστής του κινδύνου θέλω να γνωρίζω τι προβλήματα μπορεί να υπάρχουν. Ακόμη και αν αυτός που εκφράζει τα προβλήματα είναι μειοψηφία και μικρή μειοψηφία μάλιστα. Και το θέμα της συνένεσης είναι αυτό το οποίο τίθεται επιτάπητος. Χρειάζεται αντίθετη γνώμη και όχι γνώμη συνένεσης. Κύριε Πούντλη, πέντε λεπτά για να απαντήσετε. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε αρκετέ ερωτήσει, θα προσπαθήσω να είμαι σύντομο. Στι μελέτε ε, του κλάδου που ανέφερε ο κύριο Αρσένη, στι μελέτε τη βιομηχανία, δεν το συζητήσω γιατί είναι ένα ε, δεν ήθελα να το συζητήσω γιατί είναι ένα άλλο τομέα που έχει σχέση με την παρακολούθηση. Το σκεπτόμαστε πρώτον για να δούμε πώ μπορούμε να έχουμε χρήματα και δεύτερον για να ξεκινήσουν κάποιε μελέτε, για να ε, επαναληφθούν κάποιε μελέτε που έχουν γίνει από βιοτεχνολογικέ εταιρείε. Γνωρίζετε ότι η διαδικασία απαιτεί σοβαρότητα. Αυτές είναι ε, μελέτες που επαληθεύονται από ομοτήμους, peer review studies, και προσπαθούμε για ορισμένε από αυτέ τι μελέτε, όχι βέβαια για όλε, να δούμε πώ μπορούν να ξαναγίνουν αυτέ οι αναλύσει, ιδίω αυτέ οι περίφημε αναλύσει των 90 ημερών σε ποντικού, όπου ανεξάρτητα εργαστήρια ε, που θα πληρώνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μπορούσαν να μας δώσουν μια ουδέτερη ανεξάρτητη γνώμη. Δεύτερον, για τη μηδενική ανοχή για τις εισαγωγές. Ναι, προσπαθούμε να εφαρμόσουμε ένα νομοθετικό σύστημα για να επιτρέψουμε 0,1% ε, ανοχή για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς τους οποίους αξιολογεί τώρα η ΕΦΣΑ, που τώρα αξιολογεί επαναλαμβάνω, και για τις ζωοτροφές. Μόνο για αυτά όχι για τα υπόλοιπα που απευθύνονται για την ανθρώπινη διατροφή. Το 0% λοιπόν πρέπει να το προσδιορίσουμε με τεχνικό τρόπο ε, για να δούμε και πώς μπορούμε να ανταποκριθούμε στις απαιτήσει των εισαγωγών. Και είναι κάτι που θα υποβάλουμε σε ψηφοφορία στα κράτη-μέλη τον Ιανουάριο. Αλλά όχι για όλους τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς, επαναλαμβάνω, για αυτούς που αξιολογεί τώρα η ΕΦΣΑ και μόνο για τις ζωοτροφές. Ακόμη προς τον κύριο Στάς και την κυρία κορτίνα θα ήθελα να πω ότι υπάρχουν κανόνες εμπιστευτικότητας που ισχύουν για τους γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς υπό πολύ αυστηρές προϋποθέσεις. Επί τη βάση συγκεκριμένων ερωτημάτων, οι μελέτες αυτές μπορούν να ανακοινωθούν για θέματα διπλώματος ευρεσιτεχνίας, για λόγους εμπιστευτικότητας, υπάρχουν κάποια τμήματα που δεν μπορούν να δημοσιευθούν προς τα έξω, αλλά η διαφάνεια είναι πλήρης στο θέμα αυτό, επί τη βάση επίσημου αιτήματο όμως πρέπει να υποβληθεί. Για, την, για τον περίφημο καλαμπόκι Smart, είναι ένα σαραβόσιτος ε, για ε, ε, είδη διατροφής και για ζωοτροφές. Δεν έχει εκριθεί στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Προσπαθούμε να δούμε υπό ποιες προϋποθέσεις αυτή η γνωμοδότηση μπορεί να μετατραπεί σε έγκριση. Δεν έχει γίνει τίποτα όμως προς το παρόν. Για την ισοδυναμία ουσιών, όντως κυρία Λεπάζ υπάρχει η αρχή. Οι Αμερικανοί χρησιμοποιούν αυτή την αρχή για να μην κάνουν ε, επιστημονικές αξιολογήσεις ε, ε, και προσπαθούν να πούνε ότι το γενετικά τροποποιημένο φυτό είναι ίδιο με το συμβατικό φυτό, αλλά είναι κάτι το οποίο εμεί δεν χρησιμοποιούμε, γιατί ξέρετε ότι οι μελέτες χρειάζονται 4-5 χρόνια για την ΕΦΣΑ και αυτό σημαίνει ότι η αξιολόγηση είναι πολύ πιο σοβαρή από τις, τις χώρες της Βόρειας της Νότιας Αμερικής. Αυτό δεν είναι αμφισβητήσιμο. Δεν θα θέλαμε βέβαια να έχουμε συνένεση για τις επιστημονικές απόψεις. Θέλουμε να υπάρχει συνένεση για τα πρωτόκολλα των μελετών. Αυτό είναι διαφορετικό. Τα πρωτόκολλα μελέτης μπορεί να καταλήγουν σε θετικές ή αρνητικές απόψεις ε, και με απόψεις μειοψηφίας παράλληλα, αλλά κυρίως επί των πρωτοκόλων αυτών θέλουμε πληροφορίες. Αυτά κύριε Πρόεδρε, προσπάθησα να είμαι πολύ σύντομο και να απαντήσω σε όλε τι ερωτήσει, αλλά αν θέλετε μπορούμε να συνεχίσουμε και να δώσω και άλλε απαντήσει. Ευχαριστούμε πολύ. Κυρία Κουτιέρες, ε, αν θέλετε ακρόαση θα πρέπει να το πείτε στους ε, συντονιστές για να το συζητήσουμε. Είναι κάτι που πρέπει να συζητηθεί και να αποφασιστεί από τους συντονιστές αν θέλουμε να οργανώσουμε μια τέτοια ακρόαση. Λοιπόν, περνάμε στο επόμενο σημείο. Στο σημείο 8, ο Μπαρτ Στάση έχει επίση μια προφορική ερώτηση σχετικά με την εφαρμογή τη νομοθεσία για του γενετικά τροποποιημένου οργανισμού και θα δώσω κατευθείαν τον λόγο στον κύριο Πούτλη. Τα θέματα είναι γνωστά, νομίζω. Κύριε Πούτλη, θέλετε να πείτε κάτι για το θέμα αυτό, για την εφαρμογή τη νομοθεσία. Εσεί είστε ειδικό επί του θέματο και στην κατάλληλη θέση. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Θα προσπαθήσω να απαντήσω και σε αυτό το θέμα που μελετήσαμε ιδιαίτερα προσεκτικά. ξέρετε ότι μια προσέγγιση που αναπτύχθηκε στις 13 Ιουλίου για τις καλλιέργειες με αυτή τη νέα νομοθεσία για την συνύπαρξη, αυτή η νέα πολιτική δεν τροποποιεί τις αρχές της συνύπαρξης που έχει να κάνει με το εξή, να λάβουν τα κρατημέλη τα απαραίτητα μέτρα για να ε, πετύχουν ε, την τυχαία παρουσία γενετικά τροπημένου οργανισμού στα συμβατικά προϊόντα. Ο στόχο αυτή τη νέα σύσταση ε, είναι να ληφθούν καλύτερα υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου του Περιβάλλοντος του 2008 ε, σε αυτά τα συμπεράσματα γινόταν μνήα στη δυνατότητα που έχουν τα κράτη-μέλη να λάβουν μέτρα σχετικά με τη συνύπαρξη και μέσω της δημιουργίας ε, ζωνών χωρίς γενετικά τροποποιημένους οργανισμούς. Υπάρχουν ορισμένα κράτη-μέλη που θεωρούν ότι το κατόφλι του 0,9 είναι επαρκή στόχος, αλλά άλλα κράτη-μέλη οθέτησαν μέτρα για να αποφύγουν κάθε παρουσία γενετικά τροποποιημένων οργανισμών με μηδενική ενοχή. Και άλλα κρατημέλη ακόμη προέβλεψαν ε, διαφορετικούς κανόνες απομόνωσης ε, για τα προϊόντα βιολογικής καλλιέργειας. Ξέρετε ότι η Κομισιόν ε, σύστασε ένα ευρωπαϊκό γραφείο συνύπαρξη ε, στην Ισπανία με εμπειρογνώμονε που διορίζονται από τα κράτη-μέλη και που προσφέρει τεχνική υποστήριξη στα κράτη-μέλη που θέλουν να ε, καθορίσουν μέτρα σχετικά με τη συνύπαρξη. Υπήρξε ήδη δημοσίευση στι 27 Σεπτεμβρίου του 2010 ενό οδηγού των πρακτικών για την καλλιέργεια του αραβοσίτου κατόπιν ε, για τις ε, ερωτήσεις ε, που έχουν να κάνουν με τα ποια κράτη-μέλη έχουν θεσπίσει μέτρα. 15 κράτη-μέλη μέχρι σήμερα έχουν θετήσει μέτρα περί συνύπαρξης και τρία ακόμη κοινοποίησαν το σχέδιό τους στην Κομισιόν γιατί φυσικά αυτό αφορά τα κράτη-μέλη που θέλουν να προβούν σε τέτοια καλλιέργεια. Και ξέρετε υπαρχουν 6-7-6 κράτη-μέλη τα οποία έχουν ε, επιτρέψει την καλλιέργεια είτε του ορβασίτου είτε της πατάτας και τα κράτη-μέλη που δεν έχουν ε, επιτρέψει την καλλιέργεια γάμματα φαμικρά αυτή τη στιγμή, μάλλον δεν μπορεί να μην ενδιαφέρονται από αυτά τα μέτρα συνύπαρξης. Μεταξύ αυτών των 15 κρατών μελών ε, υπάρχουν 10 περίπου που προβλέπουν τη δημιουργία ενός δημοσίου μητρώου που συμπεριλαμβάνει την αναφορά της ε, τοποθεσίας της καλλιέργειας και μπορούμε εκεί να βρούμε πληροφορίες για το πού βρίσκεται η συγκεκριμένη καλλιέργεια. Υπάρχουν άλλα κρατημέλη που προβλέπουν ε, μια αναφορά στο μητρό του Γιωργού ή ε, της φάρμας. Ε, είναι δυνατό κάτι τέτοιο, αν και μπορεί να είναι λιγότερο διαφανές. Ένα κράτος προβλέπει δεδομένα που θα παρέχονται βάση γραπτού αιτήματο κάποιον ενδιαφερομένου. Και σχεδόν τρία κρατημέλη δεν προβλέπουν κοινοποίηση αυτών των πληροφοριών. συντομία αυτές είναι οι απαντήσεις, ε, Πρόεδρε, της διαφορετικής του κύριου Στάση. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε κύριε Πουλέο. Ο Μπάρτ Στάς. Θα είμαι πολύ σύντομος, Πρόεδρε. Ευχαριστώ. Είναι ένα θέμα που έπρεπε να καλυφθεί την Τετάρτη το θέμα που θα συζητούσαμε για την εφαρμογή, αλλά ζητήθηκε να συζητηθεί τώρα, γιατί είχαμε και την ερώτηση της κυρίας Λεπάζ. Και για να υπάρχει και ο αρμόδιος εκπρόσωπος της Επιτροπής. Ελπίζω να μας δώσει γραπτό στις απαντήσεις η Επιτροπή, γιατί θα με ενδιαφέρει να πάρουμε ένα αντίγραφο των απαντήσεων της Επιτροπής. Θα πρέπει να μπορούμε να ξέρουμε πώς θα τα χρησιμοποιήσουμε όλα αυτά στο μέλλον και στις επόμενες συζητήσεις που έχουμε. Νομίζω ότι ο κατάλογος των 100 μελών είναι γνωστός. Ο κ. Πούλη μπορεί να μας τα δώσει αυτά τα στοιχεία. Και... Να σας τα πω και αμέσω, άμα θέλετε. Να μας τα πείτε τότε, παρακαλώ. Ανάμεσα στους εννέα που προβλέπουν τη δημιουργία ενός εθνικού μητρώου έχετε την Αυστρία, τη Γερμανία, τη Δανία, τη Γαλλία, την Ουγγαρία, Λιθουανία, Λουξεμβούργο, κάτω χώρες και Σουηδία. Από τις δύο χώρες που προβλέπουν την ε, μνήα αυτή για το Μητρό είναι η Λετωνία και η Πορτογαλία. Το κράτος που ζητάει γραπτή αίτηση από αυτό που θέλει οι πληροφορίες είναι η Τσεχία. Και στη συνέχεια σε τρεις χώρες μέλη δεν προβλέπεται η απευθείας ανακοίνωση. Είναι η Σλοβακία, η Ρουμανία και το Βέλγιο. Αλλά για το Βέλγιο πρέπει να είμαστε προσεκτικοί διότι αυτό το περίφημο μητρό είναι ένα σχέδιο. Δεν υπάρχει δηλαδή σήμερα. Όμως οι βελγικές αρχές, από όσο ξέρω και ξέρω ότι σας ενδιαφέρει το Βέλγιο πολύ, προσοχή με το Βέλγιο, προσοχή. Αυτά λοιπόν είχα να πω για τον κατάλογο που αφορά τα κράτη-μέλη. τώρα ξέρουμε λοιπόν ποιος είναι ποιος. Κάτι ακόμα. Η Ισπανία είναι η χώρα, αναφέρεται και στην ε, ερώτησή μου, είναι η χώρα που έχει τους περισσότερους γελτικούς, ε, γελτικά οργανισμούς. Για την Ισπανία δεν σας άκουσα να αναφέρετε την Ισπανία, δεν έχετε τίποτα. y de... Όχι, δεν υπάρχει κοινοποιημένο σχέδιο επί του παρόντος όσον αφορά την Ισπανία. Αυτά λοιπόν. Έχουμε τώρα συγκεκριμένα στοιχεία. Τα έγραψε ο Μπάρτιστας, τα σημείωσε όλα. Αν υπάρχουν συμπληρωματικέ ερωτήσεις. Είναι ένα θέμα που σαφώ έχει σχέση και με την ερώτηση της Κονίλ Λεπάζ ε, και αν φτάσει το θέμα της νομοθεσία στην Επιτροπή μας θα μα απασχολήσει εκ νέου. Τώρα, Περνάμε στο σημείο 10. 9. Στο σημείο 9 της ημερήσιας διάταξης. Μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εδώ έχουμε την Εντίτα Εστρέλο, η συγγήτρια. Θα σας δώσω το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Το σχέδιο της έκθεσης είναι διαθέσιμο σε όλες τις γλώσσες. Έτσι λοιπόν όλοι οι συνάδελφοι έχουν λάβει γνώση. Βέβαια, σε ορισμένε γλωσσικέ εκδοχέ υπάρχουν κάποιε ελλείψει ε, και κάποια λάθη που θα διορθωθούν οι ανισότητες στην υγεία διαφέρουν ένα χώρα σε χώρα, από χώρα σε χώρα, από περιφέρεια σε περιφέρεια, συνεχίζονται με τις οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες και μπορεί να επιβεβαιωθούν από λόγους ε, ε, φίλου, εθνοτικούς, ε, θρησκευτικούς ή σχετίζονται με παράγοντες πολύ διαφορετικούς όπως οι συνθήκες ζωής, η συμπεριφορά της υγείας, η παιδεία, το επάγγελμα και τα, ο μισθός ε, ή οι ε, υπηρεσίες πρόληψης ε, των νόσων και πρόθεση της υγείας όπως και οι δημόσιες πολιτικές που επηρεάζουν την ποσότητα, την ποιότητα και την κατανομή των παραγόντων αυτών. Η υγεία και το προσδόκιμο της ζωής σχετίζονται επίσης με τις κοινωνικές συνθήκες και με την ανέχεια κατά την παιδική ηλικία παρά Τότε σημειώθηκαν κάποια κάποια πρόοδο σε διάφορα κράτη-μέλη, συνεχίζουν να υπάρχουν πολύ μεγάλες ε, ανισότητε ε, στα 27 κράτη-μέλη. Από την άλλη, ε, όταν η φτώχεια σχετίζεται με άλλη βάλλοντη κατάσταση, όπως η παιδική ηλικία ή τα γυρετιά, ή όταν κάποιο ανήκει σε μια μειονοτική ομάδα, τότε αυξάνονται οι κινδύνοι τη υγεία. Γι' αυτό πρέπει να παρέχεται νομική υποστήριξη ποιότητα και υπηρεσίε πληροφόρηση που να μπορούν να βοηθήσουν του πολίτε ε, να γνωρίζουν καλύτερα τα δικαιώματά του και αυτό βέβαια θα συνεισφέρει στη μείωση των ανισοτήτων. Οι ανισότητες στην υγεία, όπως ε, είπα, μπορεί να ξεκινούν από την παιδική ηλικία, να επιμηκύνονται μέχρι τα γυρατιά και να περνούν από γενιά σε γενιά. Εξού και η σημασία του θέματος και η επιτακτική ανάγκη να βρεθεί λύση. Το σημερινό πλαίσιο της παγκόσμιας κρίσης τίνει να επιδεινώνει το status quo. Όπως είναι προφανές η κρίση έχει τεράστιο αντίκτυπο στον τομέα της υγείας σε διάφορα κράτη-μέλη, τόσο σε επίπεδο προσφοράς όπως ε, και ζήτησης. Σε επίπεδο προσφοράς η κρίση οδηγεί στη μείωση της χρηματοδότησης για τη δημόσια υγεία, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει την παροχή υπηρεσιών υγεία σε μακροπρόθεσμα λόγω, σε ένα, λόγω ενός συνδυασμού παραγόντων που συνεισφέρουν για την επιδείνωση της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού γενικά. Ορισμένα κράτη-μέλη συμπεριλαμβάνουν στα προγράμματα ανάκαψης οικονομίας μέτρα για την για το μετριασμό των αντίκτυπου της οικονομικής κρίσης στον τομέα της υγείας με επένδυση στις υποδομές, ε, με την ε, βελτιστοποίηση της χρηματοδότησης και την αναδιάρθρωση των συστημάτων ε, υγείας. Ενώ άλλα κρατημέλη απλά έκαναν περικοπές στους διάφορους προϋπολογισμούς. Κάποιοι λένε ότι η κρίση είναι αποτέλεσμα των κοινωνικών ενσωτήτων. Επίσης και γι' αυτό είναι σημαντικό ε, ο περιορισμός ε, των ανισοτήτων να είναι προτεραιότητα σε όλα τα επίπεδα πολιτικής δράσης και για το λόγο αυτό εμείς ε, δηλώνουμε την ικανοποίησή μας με αυτή την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και με τους στόχους που έχει καθορίσει η ανακοίνωση αυτή σε σχέση με την έκθεσή μου. Θέλω να πιστήσω την προσοχή σας σε ορισμένες προτάσεις που θεωρώ πλέον σημαντικές πολύ συγκεκριμένα σε ό,τι αφορά στην αναγκαιότητα να προσδοθεί ιδιαίτερη προσοχή στις ανάγκες ε, των ατόμων που βρίσκονται σε κατάσταση ανέχειας, ε, στις ευάλωτες ε, ομάδες όπως τους μετανάστες, στους ηλικιωμένους, στα φτωχά παιδιά και στα άτομα με αναπηρία. Μια άλλη πρόταση έχει να κάνει με τα μέτρα για το μετριασμό του αντικτύπου της οικονομικής κρίσης στον τομέα της υγείας, κυρίως ε, στους ε, ακόλουθους τομείς. Επένδυση στις ε, υγειονομικές υποδομές, στη δημόσια υγεία, πρόθεση της υγείας και πρόληψη των νόσων, βελτιστοποίηση της χρηματοδότησης του τομέα της υγείας, αναδιάφρωση και αναδιοργάνωση του συστήματος υγειονομικής περίθαλψης. Τρίτον, έκκληση στα κράτη-μέλη για να υιοθετήσουν πολιτικές ε, που θα προσφέρουν ε, καλές συνθήκες ζωής ε, σε όλα τα παιδιά, δράση στήριξης, επίσης στις εγγύους και στους γονείς. Τέταρτον, ε, καλό το Συμβούλιο και την Κομισιόν να γνωρίσουν καλύτερα στο πλαίσιο στρατηγική ε, για την Ευρώπη του 2020 ε, το ότι η υγεία αποτελεί σημαντικό ρόλο για την καταπολέμηση του αποκλεισμού και να συμπεριληφθούν δείκτε για την κοινωνική και οικονομική κατάσταση συνοδευτικά τη στρατηγική για την Ευρώπη του 2020. Ζητώ από την Επιτροπή και τα κράτη-μέλη να παρακολουθούν τι ανισότητε στον τομέα τη υγεία Τη κοινωνική και οικονομική κατάσταση, ε, τη ηλικία του φύλου και τη γεωγραφική Διάσταση. και επίση να καταρτιστεί με μεθοδολογία για να αξιολογηθεί η κατάσταση υγεία στα κράτη-μέλη έχοντα ε, κατά νου τον προσδιορισμό των προβληματικών τομέων, τον καθορισμό προτεραιοτήτων και τη διάδοση βελτιστών πρακτικών. Τέταρτο, επίσης, τέλος, ε, είναι επιθυμητό τα διαρθρωτικά ταμεία και το Ταμείο συνοχή να υποστηρίξουν σχέδια που να συνδέονται με παράγοντε που συνεισφέρουν για την ύπαρξη ισοτήτων στην υγεία. Ε, περιμένω τα σχόλια των συναδέλφων ε, που σίγουρα θα συμβάλλουν ε, στη βελτίωση των προτεσιών μου. Εγώ θα παρουσιάσω και κάποιες προτάσεις τροπολογιών γιατί είχα ένα περιορισμό λέξεων στην αρχική έκδοση έτσι λοιπόν δεν μπορούσα να συμπεριλάβω εκεί όλα όσα επιθυμούσα. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Αντίτα Στρέλα. Θέλουμε να υπάρχει ισότητα στις υπηρεσίες υγείας και εδώ όταν υπάρχουν θέματα ανισότητα, σαφώς πρέπει να μας απασχολήσουν. Θα δώσω σε συντονιστές ε, τρία λεπτά. Φιλίπ Ζουβά από το ΕΛΚ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Καταρχήν θα ήθελα να ευχαριστήσω την κυρία Στρέλα για τη δουλειά που έκανε πρώτη μου παρατήρηση, σε μια τέτοια έκθεση που είναι πολύ σημαντική, θα πρέπει να προσέξουμε αυτά τα οποία δηλώνουμε με ιδιαίτερα έντονο χαρακτήρα. Και υπάρχουν δύο-τρία σημεία στο κείμενο ε, που αποτελούν ε, κάπως αξιωματικές διατυπώσεις. Όταν λέει ότι οι γυναίκες ζουν ε, περισσότερο, όντω αυτό είναι αλήθεια. Αλλά το ότι υποφέρουν από νόσους κατά μεγαλύτερο τμήμα της διάρκειας ζωής τους, νομίζω ότι είναι μια δήλωση που δεν ξέρω σε τι βασίζεται. Όπως επίσης όταν λέμε ότι έχουν μειώσει τα κράτη-μέλη τις δαπάνες υγείας και αυτό έχει επιπτώσει επί της υγείας, εγώ δεν γνωρίζω να υπάρχουν αποδείξεις ότι υπάρχουν λόγω της κρίσης επιπτώσεις επί της υγείας γιατί τα κράτη έχουν μειώσει τις δαπάνες. Ε, πρέπει να διακρίνουμε δύο στοιχεία στις ανισότητες υπηρεσιών υγείας που είναι πολύ διαφορετικά. Γιατί τα εργαλεία που χρησιμοποιούμε για να τα επιλύσουμε αυτά τα προβλήματα είναι διαφορετικά. Καταρχήν υπάρχουν ανισότητες που έχουν σχέση με τους περιβαλλοντικούς και κοινωνικούς παράγοντες. Ε, στέγαση, ε, επαγγέλματα που έχουν ιδιαίτερε δυσκολίε, κακή διατροφή. Όλα αυτά δημιουργούν συνθήκε ανισότητα στον τομέα τη υγεία βαθύτατε και μείζωνα σημασία ε, και μπορεί κανείς όταν, είναι, όταν δουλεύει σε ορυχεία, όταν ζει σε συνθήκες που δεν είναι ε, ε, υγιεινές, μπορεί ακόμη και να πεθάνει από αυτό. Είναι πραγματικά συνθήκες που δημιουργούν ε, ανισότητες. Ένα άλλο θέμα είναι το θέμα της πρόσβασης στις υπηρεσίες υγείας. Είναι εντελώ διαφορετικό. Όταν δεν έχουμε εύκολα πρόσβαση σε γιατρό ή σε συνθήκες περίθαλψης γιατί δεν υπάρχει γιατρός, γιατί δεν ε, ε, έχουμε πρόσβαση στα συστήματα κοινωνικής ασφάλισης που θα μας επιστρέψουν τα χρήματά μας και εδώ υπάρχει, θέματα, υπάρχει θέμα ανισότητας. Δημιουργούνται και εδώ λοιπόν συνθήκες ανισότητας εντελώς διαφορετικού χαρακτήρα. Δηλαδή να σας τα πω πολύ χονδρικά, όταν έχει κάποιος ε, μία πολύ σοβαρή νόσο στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ε, λίγο πολύ την ίδια αντιμετώπιση έχουν όλοι σε όλα τα κράτη-μέλη. Ε, σε αυτή την περίπτωση δεν έχουμε ανισότητα. Όμως στις φροντίδες ε, που δεν επιστρέφονται τα χρήματα, ε, οι συνθήκες ε, έχουν μεγάλη ανισότητα. Παραδείγματο χάρη το ότι δεν επιστρέφονται τα χρήματα για τα γυαλιά μοιοπίας δημιουργεί ανισότητες. Υπάρχουν λοιπόν ανισότητες ή για τα στοιχεία της ανείχνευσης του καρκίνου, παραδείγματο χάρη, για τις εξετάσεις ανείχνευση του καρκίνου του μαστού στις γυναίκες όταν δεν γίνονται αυτές οι εξετάσεις που είναι εξετάσεις πρόληψης οι ανισότητες που δημιουργούνται είναι μεγάλες. Λοιπόν υπάρχουν ε, ανισότητες λόγω της έλλειψης σωστής πρόσβασης σε υπηρεσίες υγείας γιατί δεν παίρνουμε πίσω τα χρήματα που δίνουμε γιατί δεν έχουμε πρόσβαση σε προληπτικές εξετάσεις σε γιατρό και οι διαφορετικές και αυτή η περίπτωση ανισοτήτων είναι διαφορετική από την προηγούμενη που αναφέρθηκα. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ πολύ. Μίλιαν Τσάπρανοχ από τους κοιόδη συζητητές ο επόμενος. Ευχαριστώ. Σας ευχαριστώ για τη σημερινή συζήτηση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό αυτό το θέμα. και θέλω να τονίσω τα μέτρα που θα μπορούσαν να ληφθούν ε, υγεία και ανισότητε. Αυτό αποτελεί μια πραγματικότητα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Παρ' όλα αυτά, δεν ε, καθορίζεται μόνο από τους κοινωνικούς και οικονομικούς παράγοντες. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες όπως ε, γενετικοί παράγοντες, η πρόσβαση στη υγειονομικό σύστημα, ε, πρόσβαση σε πληροφορίες που αφορούν ε, την υγιεινή ζωή, τον υγιεινό τρόπο ζωής και επίσης μιλάμε και για νησότητες λόγω διαφορετικής ε, και άνησης πρόσβασης στις ε, μοντέρνες τεχνολογίες. Εγώ θέλω να τονίσω την ε, πρόσβαση στις πληροφορίες για τους ασθενείς. Πιστεύω ότι η υγεία εξαρτάται από τις ε, ποιοτικές πληροφορίες τις οποίες μπορεί να έχει κάποιος ε, πρόσβαση ε, σε σχέση με τον υγιεινό τρόπο ζωής και τη σωστή διατροφή. Αν θέλουμε να ενισχύσουμε τη θέση των ασθενών, τότε θα πρέπει να παράσχουμε στους πολίτες καλές και ποιοτικές πληροφορίες και θα πρέπει να επιτρέψουμε στους πολίτες να κάνουν ενημερωμένε επιλογές και να λογοδοτούν και για τις επιλογές που κάνουν, ευθύνονται για τις επιλογές αυτές θέλω να καταθέσω κάποιες τροπολογίες για τις ανισότητες ε, γεωγραφικού χαρακτήρα και για την τηλεϊατρική. Σας ευχαριστώ. κύριος Λίζα. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστώ και την εισηγήτρια Εντιτές Στρέλα και τον Φιλίπ Ζουβάνς και ο δισηγητή Ακούσαμε τις παρεμβάσεις τους ε, και ε, βλέπουμε ότι είναι αρκετά δύσκολη η κατάσταση στον τομέα της υγείας. Εμείς ε, ως εκπρόσωποι των πολιτών της Ευρώπης πρέπει να τονίσουμε το ενδιαφέρον μας για το θέμα αυτό και να τονίσουμε ότι οι διαφορές μέσα στα κράτη της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μέσα σε κάθε κράτος μέλος πρέπει να μειωθούν και πρέπει όλοι οι πολίτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης να έχουν δικαίωμα σε ορθή πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας λόγω πολλών παραμέτρων βλέπουμε ότι δεν είναι καθόλου απλό και καθόλου εύκολο. Και αυτό το λέει και το έγγραφο της Επιτροπής. Φαίνεται ότι υπάρχει ένα πρόβλημα και δεν είναι τόσο σαφές ότι υπάρχει μία ξεκάθαρη λύση την οποία να μπορούμε εύκολα να εφαρμόσουμε και να λύσουμε το πρόβλημα. Είναι πολλοί οι λόγοι για τις διαφορές συνθήκες υγείας, ακόμη και για τα ίδια νοσήματα. Και στο σημείο 2 υπάρχει ένα πρόβλημα. Ένα πρόβλημα είναι ε, οι κοινωνικές ελλείψεις και το χάσμα στις κοινωνικές υπηρεσίες που υπάρχει. Ε, είναι δύσκολο να προσφέρονται ακριβές ε, θεραπείες όταν δεν υπάρχουν οι κοινωνικο-οικονομικές προϋποθέσεις. Και είναι πολύ δύσκολη η εξισορρόπηση εδώ. Ξέρουμε ότι υπάρχουν κοινωνικές ανισότητες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και δεν μπορούμε ξαφνικά με πολιτική βούληση να τα επιλύσουμε. Υπάρχουν βέβαια στο σχέδιο έκθεση της Δίτα ε, Στρέλλα κάποια ενδιαφέροντα στοιχεία. Πρέπει να τονίσουμε την πολιτική της υγείας στο πλαίσιο της στρατηγικής 2020. Αυτό είναι ευκταίο και είναι σημαντικό το να παίξουν πιο σημαντικό ρόλο το Ταμείο Συνοχής και άλλα. Και ο συνάδελφος Μικολάσης που δεν είναι σήμερα εδώ έχει εργαστεί ως μέλος της Περιφερειακής Επιτροπής και στη δική μας Επιτροπή για το θέμα αυτό. Υπάρχουν λοιπόν δυνατότητες. Πρέπει τα κράτη-μέλη να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες πιο προσεκτικά και θα ήθελα τέλος να δώσω ένα παράδειγμα όπου ανεξάρτητα όπου με ίδιες γενετικές προδιαθέσεις υπάρχει μεγάλη ε, διαφορά για την ε, μειοπάθεια. Ε, ε, νομίζω ότι ε, αυτό είναι ένα παράδειγμα όπου μπορούμε να βοηθήσουμε τους ασθενείς και εδώ θα μπορούσε να γίνει μια συγκεκριμένη μελέτη για να δούμε ότι με, ίδιες γενετικές, με ίδια γενετική προδιάθεση μπορούμε να μειώσουμε την επίπτωση. Ευχαριστώ. Πρόντι. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, ήθελα να ευχαριστήσω την συγκήτρια για το έργο της και να υπογραμμίσω πως ε, τον περασμένο αιώνα είχαμε πολύ μεγάλες κατακτήσεις σε κοινωνικό επίπεδο και πρέπει να είναι και σημείο αναφοράς για αυτό τον αιώνα. Δεν μπορούμε αυτές τις κοινωνικές κατακτήσεις να τις εγκαταλείψουμε. Όμως ε, υπάρχουν προβλήματα που οφείλονται στην οικονομική κρίση και θα έπρεπε να επαγρυπνούμε εμείς επί του κινδύνου αυτού. Δηλαδή, τη στιγμή που οι άνθρωποι είναι ιδιαίτερα αδύναμοι, θα μπορούσαν να δημιουργηθούν νέες ανισότητες ε, που να αφορούν την υγεία. Αυτό είναι ένας ε, πάρα πολύ σχετικός κινδυνός και εμείς πρέπει να προσπαθήσουμε να τον αποφύγουμε. Είδαμε με πόση δυσκολία και πόσε αντιδράσεις ε, αντιμετώπισε ο πρόεδρος Ομπάμα στις ΗΠΑ για να μπορέσει να προωθήσει ένα λόγο ισότητας. Και αυτό πρέπει να μας κάνει να προβληματιστούμε και να είμαστε και ιδιαίτερα προσεκτικοί για το θέμα αυτό. Ακριβώς γιατί οι τελευταίες εξελίξεις ε, μας έχουν δείξει πως ε, οι ανισότητες μεταξύ των πολιτών αυξάνονται σε ό,τι φορά το εισόδημα. Έτσι λοιπόν ε, όλα αυτά ε, μπορούν επίσης να έχουν επίπτωση και στον τομέα της υγείας. Νομίζω ότι αυτή είναι πάρα πολύ σημαντική στιγμή για να ανασχεδιάσουμε και να διοργανώσουμε τον τομέα της υγείας ε, έχοντας ε, φυσικά κατά νου και το διασυνοριακό χαρακτήρα προκειμένου να μπορέσουμε να διασφαλίσουμε μια ισότιμη πρόσβαση στην υγεία εξελίφοντας αν είναι δυνατό όλες τις διαφορές και διαφοροποίησεις που υπάρχουν μεταξύ των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ. Ντάγμα Ροτ Μπέρεντ. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ο κύριος Λίζε είπε κάτι πολύ σημαντικό. Στο τέλος της ομιλίας του μας υπενθύμησε ότι υπάρχουν απλές μέθοδοι να μπορούμε σε ασθενείς μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, σε ασθενείς που έχουν ε, ίδια γενετική προδιάθεση, ε, να δώσουμε ε, ίση ίση υγειονομική ε, περίθαλψη και να τους βοηθήσουμε. Εγώ τους του είπα εκτός μικροφώνου ότι πρέπει να το θέλουμε για να το κάνουμε, πρέπει να υπάρχει η βούληση. Ε, βέβαια υπάρχουν και δυνατότητες που ήδη υπάρχουν και δεν χρησιμοποιούνται από τα κράτη-μέλη το Ταμείο Συνοχής και τα Διαθετικά Ταμεία έχουν πολύ λίγες δυνατότητες γιατί δεν είναι μέσα τα οποία έχουν θεσπιστεί προς τούτο. Η πολιτική υγείας που αρχικά ήταν αρμοδιότητα των κρατών μελών είναι κάτι στο οποίο μπορούν τα κράτη-μέλη να κάνουν κάτι. Μόνο που τα κράτη-μέλη δεν θέλουν, δίνουν για άλλα θέματα χρήματα, για οδικό δίκτυο, για σιδηροδρομικές υποδομές, για βιομηχανικές υποδομές κλπ. και όχι για την υγεία. Και γι' αυτό μας ενδιαφέρει πολύ η έκθεση της κυρίας Εστρέλα. Υπάρχει όμως ένα σημαντικό θέμα ότι τα κράτη-μέλη ε, θα πρέπει από μόνα τους να αναγνωρίσουν τη σημασία της υγείας και να ζητηθεί αυτό από τα κράτη-μέλη. Γι' αυτό νομίζω ότι θα πρέπει να στυλιτεύσουμε τα κράτη-μέλη, να κάνουμε μια πολιτική name and shame εδώ να μην περιμένουν 10-15 χρόνια τα κράτη-μέλη για να δουν ότι δεν έχουν επενδύσει στον τομέα της υγείας τελικά. Να μπορούν ε, να ε, να, να μπορούμε να βλέπουμε πόσο της 100% του ΑΕΠ τους ε, δίνουν για το τομέα της υγείας. Να δούμε ότι κάποια κράτη-μέλη δίνουν μεγάλο ποσοστό του ΑΕΠ, αλλά κράτη-μέλη πολύ μικρό ποσοστό του ΑΕΠ και να βάλουμε ένα πίνακα που να το δείχνει αυτό και να ορίσουμε ότι θα πρέπει να επενδύουν ένα ποσοστό του ΑΕΠ τους. Να δούμε πόσο επενδύουν στην εκπαίδευση, πόσο επενδύουν ε, στις υποδομές και στο οδικό δίκτυο, γιατί θα εκπλαγούμε το πόσο λίγο επενδύουν ε, στην υγεία. Αν δούμε την ε, ποσοστιαία συμμετοχή των κρατών μελών, μπορεί αυτό να δείξει ότι είναι και αρμοδιότητα των κρατών μελών που δεν τηρείται και δεν είναι αρμοδιότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης μόνο. Ευχαριστώ πολύ. Υπάρχει η έννοια της κοινωνικής σύγκλησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μπορούμε να δούμε το ποσοστό του ΑΕΠ που δίνεται για την παιδεία και την υγεία, αλλά δεν είναι το άμεσο στοιχείο που πρέπει να μας ενδιαφέρει εδώ. Ευχαριστώ. Είναι μια θλιβερή κατάσταση. υπάρχει λίγη πρόσβαση και στην κατάρτιση για θέματα υγείας και στην υγεία γενικότερα. Υπάρχουν ομάδες οι οποίες πλήττονται περισσότερο λόγω καπνίσματος, λόγω κατάχρησης αλκοόλ ή και εξαιτία κακής διατροφής. Επειδή είναι πιο φθηνό να αγοράζει κανείς ε, μεταπημένα τρόφιμα, Πολλέ φορές υπάρχουν κατηγορίε ανθρώπων που καταναλώνουν πολύ περισσότερα τέτοια έτοιμα φαγητά από ότι τα φαγητά που μαγειρεύονται στο σπίτι, με αποτέλεσμα διάφορες ασθένειες όπως είναι ο διαβήτη και άλλες. Και τα πράγματα θα χειροτερέψουν εφόσον έχουμε οικονομική κρίση. Πρέπει λοιπόν να κάνουμε ό,τι μπορούμε για να περιορίσουμε τι βλάβε στι πιο φτωχέ κατηγορίε πληθυσμού. Ελπίζω η έκθεση αυτή να αποτελεί μόνο το σημείο κίνησης για να αντιμετωπίσουμε όλα αυτά τα πολύπλοκα ζητήματα που είναι πολλά. Και ελπίζω όλες οι χώρες να πάρουν στα σοβαρά αυτό το θέμα, διότι η οικονομική κρίση δεν είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί σαν άλοθη για να κάνει τους φτωχού να υποφέρουν ακόμα περισσότερο στις κοινωνίες μας. Αντίθετα, πρέπει να κάνουμε κάτι θετικό με αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε, Κρυς Ντέιβις. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Αντώνιο Παγανόβα είναι σκιώδη. δυστυχώς δεν μπορεί να είναι εδώ, αλλά εκ μέρου της θα πω εγώ κάποια πράγματα και θα προσθέσω και κάποια δικά μου σχόλια. Ε, και εκείνη και εγώ στηρίζουμε την ε, εισηγήτρια στην προσπάθειά της για αυτό το θέμα που είναι σημαντικό για τους πολίτες μας. Ξέρουμε ότι δουλεύει για το θέμα της διασυνοριακής υγείας με αντίθεση από το Συμβούλιο στις προτάσεις που θέλει να προωθήσει το Κοινοβούλιο. Λέει η συγγήτρια ότι αν θέλουμε να περιορίσουμε τις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν τα κράτη-μέλη για να προχωρήσουμε, ε, τι να κάνουμε, να αυξήσουμε τις ανισότητες μεταξύ μας. Τα επόμενα χρόνια θα αντιμετωπίσουμε διάφορα προβλήματα πιο έντονα, όπως την οικονομική κρίση, που είπε και η συνάδελφος πριν. Οι ανισότητες αυξάνουν εξαιτίας της οικονομικής κρίσης, οι ανισότητες μεταξύ χωρών μελών. Έπειτα υπάρχει και το δημογραφικό ζήτημα, γύρανση του πληθυσμού. Σε τι βαθμό αυτό το φαινόμενο θα προκαλέσει αλλαγές και διαφορές μεταξύ των χωρών μας. Υπάρχουν πράγματα που θα μπορούσαμε να προσθέσουμε στην έκθεση. Το ένα είναι η αναγνώριση της ε, ε, πολυπλευρούς φύσης του ζητήματος της ανισότητας και της άνησης πρόσβασης στην υγεία. Απασχόληση, οι ευκαιρίες που έχει κανείς στην απασχόληση δηλαδή, η ένταξη των μειονοτήτων και άλλα τέτοια. Δεύτερον, πρέπει να δούμε και κάποιες ανισότητες που δεν είναι τόσο προφανείς καταρχήν. Πράγματα που λείπουν από τις στατιστικές. Κάτι που έχει να κάνει με τα προβλήματα υγείας της απασχόλησης. Αν δούμε τι κάνουν τα κράτη-μέλη, τα επίπεδα αυτοκτονίας που διαφέρουν από τη μία χώρα στην άλλη και που μπορεί να έχουν να κάνουν ε, με την έλλειψη βιταμίνης δέλτα που λέγαμε και πριν ή με την έλλειψη ήλιου ή έπειτα τα ποσοστά που έχουμε για κάπνισμα, για κατανάλωση αλκοόλ. Εδώ καταλαβαίνω ότι υπάρχουν τεράστιες ανισότητες και μέσα στο Ηνωμένο Βασίλειο στις πόλεις. Μπορεί σε ένα κομμάτι μιας πόλης να έχουμε προσδόκιμο ζωής πολύ μεγαλύτερο από ότι σε ένα άλλο κομμάτι της ίδιας πόλης. Άρα δεν έχει να κάνει με την πρόσβαση στη δημόσια υγεία τελικά. Μόνο υπάρχουν και ένα σωρό άλλοι παράγοντες που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη. Τέλος, υπάρχει το θέμα στην, προ, της πρόσβασης σε ειδικέ θεραπείες. Σε ορισμένες χώρες υπάρχουν ε, διευκολύνσεις για θεραπείες που δεν υπάρχουν σε άλλες χώρες, γιατί έχουμε τους ειδικού, έχουμε τους γιατρούς που έχουν καταρτιστεί για να εφαρμόζουν κάποιες θεραπείες, πολλοί δεν υπάρχουν. Πρέπει να υπάρχει κάποια ισορροπία λοιπόν και στα θέματα της επικουρικότητας. Και ξέρω ότι η Αντώνια Παβανόβα θα ήθελε να πει ότι δεν θα πρέπει να θεωρείται αυτό πρόσχημα για να επωφελούμαστε από υπηρεσίες αλλού. Πρέπει να κάνουμε όλοι προσπάθειες. Καντίνες. Ε, κύριε Κουτιέρε, συγγνώμη, κύριε κουτιέρε, ευχαριστώ. Πρέπει να υπάρχει αρκετά κοινή λογική μεταξύ μας εδώ. Εγώ φοβάμαι ότι θα οδηγηθούμε σε μία συζήτηση χωρίς τέλος για τα θέματα υγείας. Ακούσαμε μερικά σημαντικά εδώ. Αυτό που είπε ο Πίτερ Λύση, ότι δεν είναι μόνο οικονομικό το ζήτημα. Βέβαια, αν υπήρχαν άπειρα χρήματα θα ήταν πιο εύκολα τα πράγματα. Όμως, ο δείκτης του προσδόκιμου ζωής και της υγείας εξαρτάται από τα χρήματα και από αυτά εξαρτάται και το μοντέλο υγείας που προσφέρουμε. Αν είχαμε κάποιους δείκτες και το έγραφο αυτό βοηθούσε να αποκτήσουμε αυτούς τους δείκτες με τους οποίους θα μπορούσαμε να μετρήσουμε την κατάσταση. Για μένα αυτό που λείπει από εδώ είναι ναρκωτικά και κατανάλωση αλκοόλ. είναι πράγματα το που οδηγούν ακόμη και πολλούς νέους να μειώνουν φοβερά το επίπεδο της ζωής τους. Για τους νέους πάντα έχουμε πολύ θλιβερές μελέτες που λένε και για την αύξηση του AIDS μεταξύ τους. Αυτά θα έπρεπε να σκεφτούμε. Επειδή όλες οι χώρες δεν είναι ίδιες μεταξύ τους. Όταν ξεκινήσαμε να δουλεύουμε στην προηγούμενη θητεία για την οδηγία αυτή για τη διασυνοριακή υγεία, αντιμετωπίσαμε το πρόβλημα ότι πολλές χώρες δεν θέλανε να γίνεται σύγκριση των υπηρεσιών υγείας. Τέλος, κάτι που είπανε διάφοροι συνάδελφοι. Η πρόληψη έχει να κάνει με την οτροπία που επικρατεί σε μια κοινωνία. Θα έπρεπε να υπάρχουν εκστρατείες στο εσωτερικό των χωρών, στις διάφορες αγορές. Πρέπει δηλαδή από κάτω προς τα πάνω να υπάρχει αυτή η στήριξη. Ο κόσμος να σκέφτεται από μόνοι τους διάφοροι, να μαζεύονται και να εξηγούν στον κόσμο πώς πρέπει να τρώει καλύτερα. Ή έπειτα να προσφέρουμε καλύτερες υπηρεσίες φροντίδας προς τους ηλικιωμένους. Ελίνα uh, Ευχαριστώ πολύ, Ελένα Αντωνέσκο. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Θέλω να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για τη δουλειά που έχει κάνει και να ευχαριστήσω και τον κύριο Ζουβά που ήταν εισηγητής από τη δική μας ομάδα. Για μας έχει ιδιαίτερη σημασία αυτή η συζήτηση, ιδίως διότι προέρχομαι από μια χώρα που κατονομάζεται ως πρώτη χώρα όσον αφορά την επίπτωση ορισμένων ασθενειών. Είναι μια συζήτηση λοιπόν που με ενδιαφέρει πάρα πολύ και ελπίζω να αποτελέσει απλώς την αφετηρία για να συνεχίσουμε τις προσπάθειές μας σε αυτό τον τομέα. Όντως υπάρχουν μεγάλες διαφορές μεταξύ κρατών μελών και στο εσωτερικό του ίδιου κράτους μέλους. Και θα ήθελα να τονίσω ορισμένα σχετικά ε, σχόλια που πιστεύω ότι και στο, στην έκθεσή μας πρέπει να τα αναφέρουμε. Λοιπόν, πρέπει να επιμείνουμε περισσότερο ε, μνήμα των διαθροτικών ταμείων και πρέπει να αναφέρουμε την επίπτωση των, των κοινοτικών πόρων, των πόρων της Ευρωπαϊκής Ένωσης επί της υγείας. Και όταν μιλάμε για τα διαθροτικά ταμεία, πρέπει να πούμε ότι μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για τη μείωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Όταν είναι στα χέρια των τοπικών αρχών αυτοδιοίκησης που είναι πιο κοντά στους πολίτες και μπορούν να ανταποκριθούν καλύτερα στις ανάγκες των τοπικών κοινωνιών. Επίσης πρέπει να αναφέρουμε τα μέσα τα οποία έχει στη διάθεσή της η Ευρωπαϊκή Ένωση και να δούμε ποια είναι η καλύτερη μέθοδος για αποτελεσματική παρέμβαση. Και τα κράτη-μέλη θα πρέπει να αναλάβουν συγκεκριμένες ευθύνες και πρέπει να τηρήσουν τις δεσμεύσεις που αναλαμβάνουν. Υποστηρίζω επίσης την ιδέα της δημιουργίας δικτών ανισοτήτων υγείας και τα διορθωτικά ταμεία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με βάση αυτούς τους δείκτες ανισότητα υγεία. Ένα τελευταίο σημείο που θέλω να αναφέρω είναι ότι ε, η μετανάστευση εργαζομένων είναι επίσης ένα θέμα που δημιουργεί ανισότητες ε, υγείας. Υπάρχει διαρροή εγκεφάλων σε πολλές χώρες Κεντρικής και Ανατολικής Ευρώπης. Φεύγουν γιατροί, παραδείγματος χάρη, και υγειονομικό ε, προσωπικό και επαγγελματίε υγείας που πάνε και εγκαθίσεται σε πιο πλούσιες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Στη Ρουμανία περίπου 6.000 γιατροί έφυγαν από τη Ρουμανία πέρυσι για να εγκατασταθούν σε πιο πλούσιες χώρες της Ευρωπαϊκής η Ρουμανία ήδη είχε σημαντική έλλειψη ιατρικού προσωπικού και καταλαβαίνετε ότι αυτή η κατάσταση επιδεινώνεται. Θα υποβάλω σχετικές τροπολογίες. Ευχαριστώ πολύ και τελευταία ομιλήτρια Ρίτα Μάνερ που σας καλωσορίζω και επισήμως στην πρώτη σας συνεδρία στην Επιτροπή μας. Ευχαριστώ. Αναφερθήκαν πάρα πολλές πτυχές. Έτσι λοιπόν καταρχήν να ευχαριστήσω την εισηγήτρια για το εξαιρετικό σχεδίο κειμένου. Είναι πάρα πολύ σημαντικό το θέμα αυτό, νομίζω όλοι συμφωνούμε. Και μάλιστα θέτει και πολλές προκλήσεις, γιατί όπως ε, έχει υποθεί η εδώ αναφερόμαστε και ε, στην κατάσταση που επικρατεί στα κράτη-μέλη και πρέπει να δούμε τι εργαλεία έχουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση για να ασκήσουμε πίεση στα διάφορα κράτη-μέλη. Αν δούμε ποιες διαφορές υπάρχουν ε, στα κράτη-μέλη σε ό,τι αφορά την πρόσβαση στις ε, υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, μπορούμε να δούμε ότι υπάρχουν πολλές διαφορές και στις περιφέρειες μιας ίδιας χώρας. Δηλαδή, εμείς στη Φιλανδία βλέπουμε ότι η κατάσταση διαφέρει ανάμεσα στις διάφορες πόλεις σε ό,τι αφορά την πρόσβαση πρόσβαση στις υπηρεσίες περίθαλψης. Πολλά υπόθηκαν και για την πολιτική συνοχή και για το πώς η πολιτική συνοχή μπορεί να υποστηρίξει την ε, ανάπτυξη των υπηρεσιών υγείας. Ε, εγώ είμαι και μέλος της Επιτροπής ε, Περιφερειακών Υποθέσεων και με τα διαφορετικά ταμεία υπάρχει δυνατότητα να χρησιμοποιηθούν κονδύλια για τις υπηρεσίες υγείας και αυτό έχει γίνει πολύ αποτελεσματικά στη χώρα μου. Έτσι λοιπόν πρέπει να δούμε πώς πρέπει να γίνει ο συντονισμός σε επίπεδο κράτους μέλους και σε ποιους τομείς. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να χρησιμοποιήσουμε τα διαφορετικά τομεία για την πρόθεση της υγείας. Μια ακόμη πτυχή που συζητείται και στην Επιτροπή ΕΝΒΗ έχει να κάνει με τους ε, δείκτες της πολιτικής συνοχής. Ε, έχουμε αυτή τη στιγμή ένα σύστημα που βασίζεται στο ΑΕΠ, αλλά ε, υπάρχει και μία συζήτηση για το αν θα πρέπει να συμπεριλάβουμε και κάποιους δείκτες που να βασίζονται σε δεδομένα της υγείας. Κάτι τέτοιο θα μπορούσαμε να το υποστηρίξουμε. Το θέμα της γύρανσης είναι πολύ σημαντικό όταν ε, μιλάμε για τη διαθεσιμότητα των υπηρεσιών περίθαλψης. Ε, σε ορισμένε ε, περιοχές βλέπουμε ότι οι άνθρωποι γερνούν πάρα πολύ γρήγορα. Αυτό πρέπει να το λάβουμε υπόψη, γιατί φυσικά θα υπάρχουν μεγαλύτερες ανάγκες στις περιοχές αυτές για πρόσβαση στις υγειονομικές υπηρεσίες. Αντρερίς, πέντε λεπτά για να λάβετε θέση επί του θέματος από πλευρά της Επιτροπής. Uh, Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Είναι πολύ σημαντική αυτή η έκθεση για το θέμα των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή έχει αναλάβει τη δέσμευση να καταπολεμήσει τις ανισότητες μέσα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μεταξύ των κοινωνικών ομάδων σε κάθε κράτος μέλος. Η επικοίνωση για την αλληλεγγύη στον τομέα της υγείας δημιουργεί το πλαίσιο για δράση της Ευρωπαϊκής Ένωσης ε, για να ε, βελτιωθούν οι πολιτικές της Ευρωπαϊκής Ένωσης στον τομέα της υγείας, ε, της απασχόλησης και για να δημιουργηθούν ίσες ευκαιρίες και στην περιφερειακή πολιτική. Τα διορθωτικά ταμεία και το Ταμείο Συνοχή συγκεκριμένα χρησιμοποιούν ε, ε, πόρους ε, και η αποτελεσματική τους χρήση είναι κάτι που πρέπει να έχουμε κατά νου για τη βελτίωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Όπως ήδη ελέγχθη, δεν υπάρχει εύκολη λύση για το θέμα αυτό. Πρέπει να έχουμε κατά νου την πολυμορφία που υπάρχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση τον πολύπλοκο χαρακτήρα. Θέλουμε να διευκολύνουμε τη δράση των ε, θεσμικών οργάνων της Ευρωπαϊκής Ένωσης καθώς και των κρατών μελών και των ε, τοπικών φορέων και εδώ η εταιρική σχέση είναι η λέξη κλειδί για το μέλλον. Η πρόταση ψηφίσματος ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου θα υποστηρίξει αυτή την προσπάθεια και όπως ήδη αναφέρθηκε αυτή τη στιγμή με την οικονομική κρίση υπάρχει άλλη μια απειλή για επιδείνωση των ανισοτήτων στον τομέα της υγείας. Η υγεία είναι ο πιο πολύτιμος πόρος των πολιτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης, συνδέεται άμεσα με την απασχόληση και είναι ενδιαφέρον να δούμε και τα θέματα ε, δαπανών των κρατών μελών για τον τομέα της υγείας ως ποσοστό του ΑΕΠ. Η στρατηγική Ευρώπη 2020 είναι επίσης σημαντική σε αυτό τον τομέα γιατί θέλει να μειώσει τις ανισότητες και ελπίζουμε ότι ε, θα βοηθήσει να ανταποκριθούμε στις ανάγκες στον τομέα αυτό. Για την υγεία, την πρόληψη και την πρόσβαση σε υπηρεσίες υψηλής ποιότητας υγείας είναι άλλο ένα σημαντικό θέμα που αναφέρεται στην έκθεση. Αναφερθήκατε και στην οδηγία και στην συνεργασία μεταξύ διαμεθοριακών περιοχών, ούτως ώστε να υπάρχει βελτιωμένη πρόσβαση σε υπηρεσίε υγεία και να χρησιμοποιείται ε, και οι, ε, χρησιμοποιούνται και οι γεωγραφικές παράμετροι και η τεχνολογία που μπορεί να τεθεί στην υπηρεσία της υγείας. Σας ευχαριστώ όλους σας που συμμετείχατε σε αυτή τη συζήτηση. Και μέσα στα επόμενα χρόνια, το 2012, θα ετοιμάσουμε μια έκθεση σχετικά με τους δείκτες τους οποίους ζητήσατε κι εσείς για να μπορούμε να κατανοήσουμε καλύτερα αυτά τα σημαντικά φαινόμενα που συζητάμε σήμερα. Σας ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστούμε κύριε Ρης και ευχαριστούμε και όλους ε, σας που λάβατε το λόγο για αυτό το σημαντικό θέμα. 10 Δεκεμβρίου είναι η προθεσμία για τις τροπολογίες ε, στις 12. Τον Ιανουάριο θα συζητήσουμε την έκθεση της κυρίας Αστρέλα στην Επιτροπή και το Μάρτιο στην Ολομέλεια. Περνάμε στο επόμενο σημείο, στο σημείο 10. Έντιτε, θέλει το λόγο άλλη μια φορά, σύντομα παρακαλώ. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να ευχαριστήσω τους συναδέλφους για τις συνεισφορές τους. Όπως και εγώ εμένα είναι ιδιαίτερα εμπλουτιστικά τα σχόλια που ακούστηκαν και θέλω να υπογραμμίσω ότι δεν υπάρχουν πράγματι εύκολες λύσεις. Ε, πόσο μάλιστα λάβουμε υπόψη ότι είναι πολύ μεγάλες ε, οι διαφορές μεταξύ των κρατών μελών. Όμως ε, είναι αλήθεια ότι οι ανισότητες στην υγεία ε, είναι συνέπεια άλλων υφιστάμενων ανισοτήτων στην κοινωνία. Και θα έπρεπε να καταβάλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια για να τις καταπολεμήσουμε και για να επιλύσουμε αυτή την κατάσταση. Πολύ γρήγορα θα ήθελα να αναφερθώ σε ορισμένα από τα σχόλια που ακούστηκαν συγκεκριμένα στο ζήτημα της πρόληψης. Εγώ πιστεύω ότι αυτή η προσέγγιση πρέπει να γίνει σε δύο επίπεδα. Δηλαδή, στο επίπεδο της πρόληψης ε, πρέπει να καταπολεμήσουμε τους παράγοντες ε, που προκαλούν τις ανισότητες στην υγεία και αφετέρου σε ένα δεύτερο επίπεδο πρέπει να δημιουργήσουμε καλύτερες προϋποθέσεις ε, για την πρόσβαση στις υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης για όλους τους πολίτες. Επίσης αυτό έχει να κάνει και με την ενημέρωση των πολιτών για τα δικαιώματά τους, ε, για το τι είναι διαθέσιμο και πώς μπορούν ε, να επωφεληθούν οι πολίτες. Σε ό,τι αφορά τώρα τα κοινοτικά ταμεία που αναφέρθηκαν από διάφορους συναδέλφους, συμφωνώ απόλυτα ότι πρέπει να εκμεταλλευτούμε καλύτερα τους υφιστάμενους μηχανισμούς το υπογραμμίζω αυτό εκ νέου. Τα διαρθρωτικά ταμεία θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν καλύτερα. Υπάρχουν βέλτιστες πρακτικές ε, σε πολλά κράτη-μέλη για το πώς έχουν χρησιμοποιηθεί ορθά οι κοινοτικοί πόροι στον τομέα της υγείας. Και όλο ένα και περισσότερο θα είναι απαραίτητο να γίνει κάτι τέτοιο, γιατί έχουμε τη γύρω του πληθυσμού, δημογραφικές ε, εξελίξεις στη σύνθεση του πληθυσμού και είναι προφανώς ότι το κόστος ε, της υγειονομικής περίθαλψης θα αυξηθεί. Και φυσικά αυτό θα προκαλέσει και μεγαλύτερες ανισότητες, γιατί υπάρχουν ε, πολλά άτομα που έχουν μεγαλύτερη δυσκολία να έχουν πρόσβαση στη υγειονομική περίθαλψη. Αυτό αναφέρθηκε και από κάποια συνάδελφο Παίρνοντα χάρη πρέπει να ε, υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες και δυνατότητα πρόσβασης στις πληροφορίες για να γίνει παίρνοντα χάρη η ανείχνευση κάποιων ε, νόσων. Και για να ολοκληρώσω όλα τα στοιχεία που εγώ αναφέρω στο σχέδιο της έκθεσης ναι, προέρχονται από μελέτες ή από την ίδια την ανακοίνωση της Κομισιόν και από τη σύνοψη της μελέτης αντικτύπου που συνοδεύει την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Έτσι λοιπόν μιλάμε για στατιστικά στοιχεία αξιόπιστα κατά την απόψή μου καθώς προκύπτουν από μελέτες. Σας ευχαριστώ. Ευχαριστούμε την Εντίτα Στρέλα για τη δουλειά που έκανε για αυτή την απαιτητική έκθεση. Και τώρα περνάμε στο σημείο 10, δυναμικό μείωση ε, του διοξιδίου του άνθρακος που εκπέμπουν τα βαρέα οχήματα επαγγελματική χρήση. Ο κ. Φίλιπ Όουεν από πλευρά τη Επιτροπή. Σας ευχαριστώ Πρόεδρε. Καλό απόγευμα σε όλους και σας ευχαριστώ που μου δίνετε την ευκαιρία να έρθω και να σας μιλήσω για το έργο της ε, ΓΑΜΑ ΔΕΛΤΑ για την καταπολέμηση της κλιματικής αλλαγής για το θέμα αυτό. Θα σας προσθέσω το σκηνικό. Οι μεταφορές αποτελούν ένα πάρα πολύ σημαντικό τμήμα των συνολικών εκπομπών του διοξιδίου του άνθρακα 25% στην Ευρωπαϊκή Ένωση των ε, εκπομπών ε, προέρχονται από βαρέα οχήματα. Έτσι λοιπόν ε, αυτό μεταφράζεται στο 25% των συνολικών εκπομπών ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Μία αύξηση στις εκπομπές ε, μεταξύ του 60% και του 70% αναμένεται μεταξύ του 2019 και του 2050. Τότε θα μιλάμε για το μεγαλύτερο μέρος που θα καλύπτουν αυτές οι εκπομπές στις συνολικές εκπομπές εκπομπέ τη Ευρωπαϊκή Ένωση Δεξιδίου του Άνθρακα. Έτσι λοιπόν, θέλουμε να πετύχουμε του στόχου μα, θα πρέπει να μειώσουμε τι εκπομπέ αυτέ. Έτσι λοιπόν, οι εκπομπέ των βαρύνων οχημάτων αναμένεται να αυξάνονται σε σχέση και με την ανόδο του ΑΕΠ, αν δεν αναλάβουμε δράση, αν ε, με την ε, ρύθμιση των ε, εκπομπών για τα αγιοταχή. Είδαμε ότι δεν ήταν επαρκής η ρύθμιση αυτή που τέθηκε πέρσι σε ισχύ. Ε, αν δούμε τα δεδομένα από το 2009, βλέπουμε ότι υπάρχει σημαντική μείωση ε, στις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα από τα οχήματα επίσης. Ε, ε, υπάρχει και σημαντικός ανταγωνισμός μεταξύ των αυτοκινητών και αυτό θα ισχύσει και στο μέλλον. Πρέπει να διασφαλίσουμε ότι τα πρότυπα της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την αποδοτικότητα είναι τα πιο αποτελεσματικά παγκοσμίω. Όπως το γνωρίζετε, ένας προφανής τομής δράσης είναι τα βαρέα οχήματα επαγγελματική ε, χρήση. Δεν έχουμε μια στρατηγική, πάντως την άνοιξη φέτος, η στρατηγική της Κομισιόν για τα πιο καθαρά και πιο αποδοτικό οχήματα μετά ανέφερε ότι θέλει να αναπτύξει μια στρατηγική, αλλά δεν έχει δέσει συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα. Υπάρχουν ε, πολλές αυτοκινητοβιομηχανίες ε, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, όμως η βιομηχανία βαρέων οχημάτων είναι αρκετά κατακαιρματισμένη. Ε, είχαμε πάρα πολλούς και μεμονωμένους ιδιοκτήτες και άλλους εταιρείες που κατέχουν στόλους λοιπά. Έτσι λοιπόν η Κομισιόν θέλει να ξεκινήσει μία μελέτη φέτος για να κατανοεί αναλύσουμε τον αριθμό της ε, κατανομής των χρηστών, των οχημάτων, τον, τον, σημερινό ε, μέγεθος ε, του στόλου και θέλουμε να δούμε και πόση ενέργεια καταναλώνεται από, αυτό, αυτά τα οχήματα και ποια, υπάρχει, ε, ποια είναι η σχέση που υπάρχει μεταξύ της κατανάλωσης ε, βενζίνης και της εκπομπής διεξουδίτου του άνθρακα και να κατανοήσουμε τις υφιστάμενες τεχνολογίες, να κάνουμε μια μελέτη για τις μηχανές και μια μελέτη για τις νέες τεχνολογικές δυνατότητες. Είναι Επίσης η μελέτη θέλει να περάσχει μία αξιολόγηση των ε, επιλογών πολιτικής που θα μπορούσαν να δουν όπως η εμπορία εκπομπών, ε, νομοθεσία για να θέσουμε απαιτήσει επιδόσεων για όλα τα οχήματα και τα μέρη ε, των αυτοκινήτων. Επίσης ένα σύστημα παρακολούθησης που ανακαλύπτει την επίδοση των οχημάτων που πολλούνται καθώς και τα καύσιμα και ίσως να μπορέσουμε να αλλάξουμε και την νομοθεσία για το βάρη και τις διάστασεις και της διαστάσης ε, για να ε, δούμε αν πρέπει επίσης να μειώσουμε τα όρια της ταχύτητας για τα βαρέα οχήματα. Όλα αυτά θα ολοκληρωθούν την άνοιξη του χρόνου. Όμως η αγορά είναι μόνο το πρώτο βήμα. Ε, ένα ακόμα εμπόδιο είναι ότι δεν έχουμε μία μέθοδο για να αποστικοποιήσουμε ε, τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για τα βαρεοχήματα επαγγελματικής χρήσης. Όταν έχουμε μία τέτοια μέθοδο ε, είναι δυνατό να καταλήξουμε σε συμπεράσματα. Ξέρουμε ότι η βιομηχανία θέλει να αναπτύξει μία μέθοδο για να μειώσει τις εκπομπές ε, και η Κομισιόν υποστηρίζει αυτή τη διαδικασία και γι' αυτό αναλαμβάνουμε και ένα δεύτερο έργο, αυτή είναι μία μελέτη που έχει να κάνει με τη δοκιμή ε, μεθόδων πιστοποίησης για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα και για την κατανάλωση βενζίνης των οχημάτων αυτών. Αυτό θα ε, μελετήσει, μάλλον θα καταρτήσει μία μέθοδο με πιστοποίηση σε αυτών των οχημάτων ε, παγκοσμίω. Θέλουμε να δούμε τα γραμμάρια το χάρη ανά ε, χιλιόμετρο ανάλογα με το βάρος που μεταφέρεται και ε, αυτό θα έχει να κάνει με τα βαρέα οχήματα επαγγελματική ε, χρήση. Ε, είναι πολύ δύσκολο. Ε, θέλουμε να καταλήξουμε σε μία δοκιμή ακρίβεια και να χρησιμοποιήσουμε και εξομοίωση με υπολογιστέ. Βάσει των αποτελεσμάτων αυτή τη διαδικασία, ελπίζουμε να μπορέσουμε να καταλήξουμε σε ένα σύστημα προκειμένου να μπορέσουμε να αιμοδοποιήσουμε τι διάφορε δομέ και τα διάφορα οχήματα και τα τρέλερ και να να έχουμε διάφορες κατηγορίες επιδόσεων. Όλα αυτά ελπίζουμε να ολοκληρωθούν την άνοιξη του 2012 αυτό το έργο δεν θα πρέπει να ειδωθεί μεμονωμένα. Η Κομισιόν ε, ξέρει ότι προωθούνται ε, διάφορες σχετικές νομοθετικές προτάσεις από την EPA στις Ηνωμένες Πολιτείες ε, και από την Βουλή των Αντιπροσώπων και θέλουμε επίσης να δούμε πώς όλα αυτά επηρεάζουν και τους υπόλοιπους φορείς αυτή τη στιγμή αυτό αποτελεί η προτεραιότητά μας Θέλουμε να διασφαλίσουμε ότι ο κανονισμός ε, για τα φορτηγά θα τεθεί σε εφαρμογή. Δεν υπάρχει αυτή τη στιγμή ε, βέβαια χρονοδιάγραμμα για το πώς θα προωθήσουμε το νομοθετικό έργο μας για τα βαρέα οχήματα. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε πολύ κύριε Όν για την εισαγωγή σας. Ο Chris Davis έχει ήδη ζητήσει το λόγο. Μπορεί να μην υπάρχει χρονοδιάγραμμα, αλλά εσείς είπατε ότι σε 7 σταθμούς θα σταματήσει το τρένο σε διάφορες ημερομηνίες. Πότε θα φτάσει στον τελικό του προορισμό δεν ξέρουμε, κάπου πάντως κινείται. Πρώτα απ' όλα, ζητάω από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να σταμα... θα σταματήσει να τονίζει το θέμα του διοξιδίου του άνθρακα. Νομίζω ότι όλη η νομοθεσία θα κάνει περισσότερο πρόεδρο στο Συμβούλιο αν μιλάμε για ε, αποτελεσματικότητα καυσίμων πιο πολύ. Είναι βλέπετε και αυτός ένας ε, τομέας όπου υπάρχουν αυτοί που πιστεύουν ότι πρέπει να γίνουν μεγάλες αλλαγές και αυτοί που θέλουν να χρησιμοποιήσουν καλύτερα τους σπόρους. Το θέμα είναι πόσο αποτελεσματικοί μπορούμε να είμαστε. Αποτελεσματικότητα καυσίμων λοιπόν, έτσι ώστε να χρησιμοποιούμε με καλό τρόπο τους φυσικούς σπόρους μειώνοντας τα έξοδα. Αυτό που λέτε εσείς, ε, μείωση διοξιδίου του άνθρακα, εντάξει, δεν φαίνεται τι εννοείτε. Τώρα, την νομοθεσία αυτή τη χρειαζόμαστε όταν πρόκειται για τα βαρέα οχήματα. Έχει καλές επιδόσεις μέχρι τώρα η Ευρωπαϊκή Ένωση. Για τα επιβατικά, εκεί όπου έχουμε νομοθεσία, έχει υπάρξει δράση από πλευρά της βιομηχανία προ όφελο των οδηγών και όσον αφορά την κατανάλωση καυσίμων κλπ. κλπ. Είναι πρόοδο. Οι μηχανικοί πάντα λένε ότι μπορούν, ναι. Αλλά πάντα μπαίνουν φραγμοί στο να τα καταφέρουν. Τελικά γίνεται όμως. Οπότε είμαι υπέρ της Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας σε αυτό το τομέα μάλλον. Βέβαια τα προβλήματα που εντοπίσετε κι εσείς τα αναγνωρίζω. Πώς κάνετε συγκρίσεις, πώς ε, βάζετε ένα σύστημα αξιολόγησης, πώς τα εφαρμόζετε. Όταν όμως πρόκειται για την μεταφορά τα βαρέα οχήματα, εκεί δεν χρειάζεται. Γιατί σε αντίθεση με ό,τι συμβαίνει με τα επιβατικά ή με τα ελαφρά οχήματα, αυτοί που αγοράζουν τα φορτηγά γνωρίζουν πάρα πολύ καλά ποια είναι η κατανάλωση σε καύσιμα που έχουν και η εμπορία τους γίνεται βάση της χαμηλής κατανάλωσης καυσίμων. Έτσι τα διαφημίζουν αυτοί που θέλουν να τα πουλήσουν. Όταν πρόκειται για απόδοση καυσίμων, οι κατασκευαστές οχημάτων, οι ίδιοι τονίζουν στις διαφημίσεις τους το θέμα αυτό της κατανάλωσης καυσίμων. Το θέλει ο κόσμος. Αντίθετα, με τα φορτηγά δεν γίνεται αυτό. Ας δούμε λοιπόν πώς γίνεται η διαφήμισή τους και πόσο μεγάλη σημασία δίνουν οι κατασκευαστές για να πουλήσουν τα φορτηγά τους σε αυτό το θέμα της ενεργειακής απόδοσης, της ε, κατανάλωσης καυσίμων. Χρειάζεται δηλαδή τελικά γι' αυτά. Αυτό πρέπει να δούμε. Μακάβεν, Λίντα Μακάβεν. Μας δώσατε τα στοιχεία για οχήματα. Αυτά τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα, σε τι αναλογία ε, δημιουργούν εκπομπές διοξιδίου του άνθρακα για να δούμε κατά πόσο το χρειαζόμαστε. Και έπειτα υπάρχουν και τα λεωφορεία, τα πούλμαν. Εκεί ποια είναι η κατανάλωση και ποιες είναι οι εκπομπές. Ξέρω ότι έχουν υπάρξει πρωτοβουλίες από επιχειρήσεις, πολλές πόλεις έχουν τη δικιά τους πολιτική για την χρήση λεωφορείων εκεί. Λοιπόν, έχετε στοιχεία όσον αφορά τα λεωφορεία και τα πούλμαν. Δεν θέλει κανείς άλλο το λόγο και ο αν θέλετε να απαντήσετε εσείς τώρα στις ερωτήσεις. Θα προσπαθήσω από, την αρχή, το τέλος προς την αρχή να απαντήσω. 25% της, ε, των εκπομπών τις οδικές ε, μεταφορές εκπροσωπούνται από τα, οχήματα, από τα βαρέα οχήματα, τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Όσον αφορά τα λεωφορεία, σαφώς είναι διαφορετικά από άλλα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Δεν είναι η ίδια η κατηγορία. Γιατί υπάρχουν και μεταξύ των λεωφορείων τα αστικά λεωφορεία που έχουν πολλές τάσεις, σταματάνε, ξεκινάνε κλπ. Και υπάρχουν πολλά θέματα τα οποία πρέπει να λάβει κανείς υπόψη να μιλάμε για τα λεωφορεία και πούλμαν όταν μιλάμε για τις μετρήσεις, για το πώς θα υπολογίσουμε, θα πρέπει να πούμε διοξείδιο του άνθρακος ανά χιλιόμετρο που ταξιδεύει κάθε επιβάτης ή κάτι τέτοιο. Δεν είναι το ίδιο όπως με τη μεταφορά εμπορευμάτων. Έχουμε δύο ε, καθήκοντα. Καταρχήν να κατανοήσουμε την αγορά για να δούμε αν είναι βαρέα επαγγελματικά οχήματα λεωφορεία. Είναι αλλά είναι διαφορετικά. Την περσμένη εβδομάδα συναντήθηκα με τους UITP και είδα ότι και για τα λεωφορεία έχουν θέματα υπόψη τους ε, και ε, στα φορτηγά, στα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Έχουμε ε, τα απορριμματοφόρα, έχουμε τα αστικά φορτηγά, έχουμε τα 40 τόνων. Πολύ διαφορετική τομή και πρέπει να καταλάβουμε ποια οχήματα θα έπρεπε ε, ε, ε, να μας απασχολήσουν περισσότερο. Το πρώτο δηλαδή που πρέπει να κάνουμε είναι να καταλάβουμε την αγορά και τους σκοπούς για τους οποίους διατίθενται αυτά τα οχήματα. Και η βιομηχανία, η Volvo, η Scania κλπ. έχουν πάρα πολλούς υποτομείς και πρέπει να κατανοήσουμε τις ιδιαιτερότητες αυτής της αγοράς. Περνώ στις ερωτήσεις του κυρίου Ντέιβις τώρα, αν χρειαζόμαστε νομοθεσία. Ε, όπως σας είπα πρέπει να κατανοήσουμε την αγορά και αφού κατανοήσουμε την αγορά πρέπει να δούμε πώς μπορούμε να προετοιμάσουμε την νομοθεσία, πώς μπορούμε να κάνουμε τη μέτρηση των εκπομπών από τα οχήματα αυτά και ακόμη αυτό δεν το γνωρίζουμε. Από την άλλη πλευρά συμφωνώ πλήρως μαζί σας ότι πρέπει να αλλάξουμε την παρουσίαση, το marketing. Δηλαδή θα πρέπει να τονίσουμε τη σημασία της ανάπτυξης, των θέσεων απασχόλησης, της καινοτομίας. Γιατί να μιλάμε για το καύσιμο και να μιλάμε για την κατανάλωση καυσίμου. Ε, δεν θα έλεγα ότι δεν πρέπει να συζητάμε για τις εκπομπές διοξιδίου του άνθρακος, γιατί και αυτό πρέπει να το βάλουμε. Αλλά όντως το πώς θα το παρουσιάσουμε, το πώς θα πουλήσουμε το όλο πακέτο είναι σημαντικό όπως είπατε. Και πρέπει ε, να τονίσουμε την καινοτομία, την ανάπτυξη της θέσης απασχόλησης και παράλληλα το ότι θα κάνουμε και κάτι καλό για το περιβάλλον. Έτσι πρέπει να το παρουσιάσουμε στον κλάδο. Εδώ μα ενδιαφέρουν και οι διεθνεί εξελίξει. Είπα ότι οι ΗΠΑ αναπτύσσουν τώρα νομοθεσία για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Το ίδιο κάνει και η Ιαπωνία. Και νομίζω ότι είναι σημαντικό αυτά που θα κάνουμε να το κάνουμε έχοντα κατά νου τον κλάδο. Γιατί αν δούμε ότι οι Ευρωπαίοι παραγωγή είναι πιο αποτελεσματική από τους άλλους, αυτό θα μας βοηθήσει να πουλάμε οχήματα διεθνώς. Παράλληλα πρέπει ε, να αναπτύξουμε την νομοθεσία μας ε, ε, παράλληλα με άλλες χώρες για να μην χρειάζεται οι κατασκευαστές οχημάτων να πληρούν διαφορετικές προδιαγραφές εδώ και σε άλλα μέρη του κόσμου, τόσο ώστε να είναι ισόφελος των παραγωγών αυτό το οποίο κάνουμε. Ευχαριστώ πολύ. Σας ευχαριστώ. Ερωτήσεις Chris Davis. Η ερώτησή μου ήταν αν έχετε κάνει κάποια εξέταση ε, του τρόπου με τον οποίο διατίθεται στην αγορά αυτά τα οχήματα. Πώς λαμβάνουν οι κατασκευαστές υπόψη την αποδοτικότητα σε σχέση με το, με καύσιμο όταν πουλάνε τα οχήματά τους. Ακόμη ετοιμάζετε τις μελέτες σας, λέει ο Έτσι δεν είναι, δεν θα ξέρετε ακόμη. Ε, Επιτροπή. πρέπει να είναι τμήμα τη μελέτης και αυτό από τον ε, ο κλάδο σαφώ μα λένε ότι πρέπει να λάβουμε υπόψη και πώ λειτουργεί το θέμα των εκπομπών ε, και τη κατανάλωση καυσίμου. Από ό,τι μα έχει πει ο κλάδο, η αποδοτικότητα του καυσίμου είναι πολύ σημαντικό γιατί είναι μεγάλο κόστο για τα βαρέα επαγγελματικά οχήματα. Σα ευχαριστώ πολύ. Θα περιμένουμε λοιπόν με μεγάλο ενδιαφέρον τη μελέτη και τι ε, νομοθετικέ πρωτοβουλίε που ενδέχεται να προκύψουν. Και τώρα έχουμε ένα τελευταίο σημείο στην ημερήσια διάταξη την έμεση αλλαγή χρήση γη και τα βιοκαύσιμα. Το σημείο 13 που είπαμε ότι θα συζητήσουμε. Ένα θέμα που έχει δημιουργήσει πολλέ συζητήσει, υπάρχουν και πολλέ μελέτε και γι' αυτό πρέπει και εμεί να το συζητήσουμε. Ο Φίλιπ Όουεν από τη Γενική Διεύθυνση Κλίμ θα μα πει και ο Γιάννη Φανστέν από τη Γενική Διεύθυνση Ενέργεια. Δεν ξέρω ποιο θέλει να ξεκινήσει, ο κ. Φανστέν, για να πάρει ανάσα ο κ. Όουεν λίγο που μίλησε πολύ. Παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και καλησπέρα σε όλους σας. Όπως φαντάζεστε, θα σας μιλήσω εκ μέρους της Γενικής Διεύθυνσης Ενέργειας, τα and Action, μια που είμαστε υπεύθυνοι για θέματα περιβάλλοντος. Καταλαβαίνω πολύ καλά γιατί έχετε βάλει στην ημερήσια διάταξη αυτό το θέμα. Είναι σημαντικό το να συζητάμε τα βιοκαύσιμα και την αηφόρα ανάπτυξη. Βέβαια είναι πράγματα πολύ σημαντικά επί του παρόντος. Την Κυριακή ε, ξεκινάνε να εφαρμόζονται τα κριτήρια για τα βιοκαύσιμα και την αηφορία. Χρειάστηκε μεγάλη πολιτική και τεχνική προσπάθεια. Θα χρειαστεί και διοικητική προσπάθεια από πλευράς της αγοράς για να δείξει ότι τα βιοκαύσιμα που βρίσκονται στην αγορά ανταποκρίνονται στα κριτήρια εφορίας. Εφόσον είναι έτσι, τα κράτη-μέλη θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν τα βιοκαύσιμα αυτά για να πετύχουν τους στόχους της χιλιετίας και ε, θα μπορέσουν έτσι να πετύχουν και τους στόχους για την μείωση εκπομπών διοξιδίου του άνθρακα που επίσης αναφέρονται στους στόχους. Επιπλέον τα βιοκαύσιμα θα μπορούν να τύχουν ε, οικονομική στήριξης από το δημόσιο εφόσον όντω ανταποκρίνονται στα κριτήρια αυτά. Πρέπει να συζητήσουμε για αυτό το θέμα, διότι η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το Δεκέμβριο πρέπει να παρουσιάσει μία μελέτη. Εφόσον πρέπει, θα συνοδεύεται και με νομοθετική πρόταση η μελέτη μας αυτή. Δεν θα σας εκπλήσει να ακούσετε ότι ετοιμάζοντας την έκθεσή μας αντιμετωπίσαμε πολλές δυσκολίες, πολλές αλλαγές, έτσι κι αλλιώς είναι περίπλοκο το θέμα. Έχουμε τα κριτήρια βιωσιμότητας που έχουν να κάνουν με την αλλαγή χρήσης γης. Όμως, μπορούν να υπάρξουν και διαρροές κατά κάποιο τρόπο. Δηλαδή υπάρχουν έμεσες αλλαγές χρήσης της γης, αλλαγές στην καλλιέργεια από το ένα μέρος στο άλλο ή από ένα λόγο για κάποιον άλλον, έμεσα έχουν σαν αποτέλεσμα να υπάρχει επέκταση της καλλιέργειας σε κάποιο άλλο σημείο. Αν αυτό συμβεί σε μέρη που υπάρχει ε, μεγάλη ε, ελευθέρωση διοξιδίου του άνθρακα, μπορεί να υπάρξουν ακόμα περισσότερα αέρια του θερμοκηπίου. Αυτή η έμεση μερη που υπαρχει μεγαλη ε ελευθερωση διοξιδιου του ανθρακα μπορει να υπαρξουν ακομα περισσοτερα αερια του θερμοκηπιου αυτη η εμεση αλλαγη στη χρήση γης είναι κάτι που δεν μπορούμε εύκολα να μετρήσουμε και να υπολογίσουμε. Γίνεται εκτίμηση. Χρησιμοποιούμε μοντέλα γι' αυτό. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή λοιπόν ξεκίνησε με τέσσερις διαφορετικές αναλύσεις για να αντιληφθεί καλύτερα την εξέλιξη και τη διαδικασία. Βάσει αυτών των μελετών είχαμε και διαβούλευση από τον Ιούλιο μέχρι τέλη Οκτωβρίου. Τα κύρια ερωτήματα που τέθηκαν στις διαβουλεύσεις αυτές ήταν πρώτον, κατά πόσο αυτή η αναλυτική δουλειά αποτελεί καλή βάση για να καθορίσουμε πόσο σημαντική είναι η έμεση αλλαγή χρήση γης. Και δεύτερον, κατά πόσο χρειάζεται ευρωπαϊκή δράση και αν ναι, τι είδους δράση χρειάζεται από πλευρά της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είχαμε 140 περίπου απαντήσεις που πήραμε από οργανώσεις, από πολίτες και από κράτη-μέλη. Επί του παρόντος ετοιμάζουμε την έκθεσή μας, σε αυτή τη διαδικασία βρισκόμαστε, βάσει της αναλυτικής δουλειάς που κάναμε και βάσει των αντιδράσεων που είχαμε από το κοινό κατά τη διάρκεια της διαβούλευσης αυτής, όσο ήταν αυτή ανοιχτή. Θα έχουμε και πάλι συζήτηση με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, όταν θα έχουμε ολοκληρώσει την έκθεσή μας και θα έχουμε κάτι πιο συγκεκριμένο να συζητήσουμε μαζί σας. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε, κύριε Φανσένα, κύριε Thank you, Mr. Chairman. Ευχαριστώ. Όπως αναφέρει και ο Χάνης, μίλησε εκ μέρους και των δύο γενικών και εδώ ενέργειας και climate action. Ε, εμείς ε, παρακολουθούμε από πάρα πολύ κοντά αυτό το έργο και έχουμε και μια ομάδα ανθρώπων που εργαζονται και για τις δύο γενικές διευθύνσεις ε, επί της παρούσας έκθεσης. Δεν έχω τίποτα να προσθέσω αυτή τη χρονική στιγμή. Νομίζω ότι θα είναι το καλύτερο αν μας θέσετε ερωτήσεις όπου μπορούμε να απαντήσουμε πληρέστερα. Ευχαριστώ. Yeah. Έχουμε αρκετούς που έχουν ζητήσει το λόγο. Κρήτον Αρσένης είναι πρώτο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Πρώτη ερώτηση για το θέμα της ε, αν σκοπεύετε να λάβετε υπόψη ε, σε ό,τι αφορά τις επιπτώσεις που υπάρχουν ε, στα δάση σε σχέση με την έμεση αλλαγή χρήσης ή αν, ε, όταν θα μετρήσετε ε, τις εκπομπές ε, διοξιδίου του άνθρακα θα λάβετε υπόψη άλλες μελέτες τώρα για τις διαπραγματεύσεις στο Κανκούν που λαμβάνουν χώρα τώρα. Ποια θα είναι η στάση της ε, Ευρωπαϊκής Ένωσης σε σχέση με το Red Plus. Ja, dann äh, gebe ich das Wort an Claude Thomas, der frühere Berichterstatter über die Renewable Energy. Thomas είναι εισηγητής ε, για τις ανανεώσιμες ενέργειες, για την οδηγία. Θα σας δώσω το λόγο λοιπόν. Κύριε τούρμες, Ευχαριστώ Πρόεδρε. Να υπενθυμίσω από πού ξεκινήσαμε και βλέπω και την κυρία Γκροστέτ που επί Γαλλικής Προεδρίας μας βοήθησε πολύ να προχωρήσουμε και έχω και μία παρατήρηση για την καινοτομία. Όλοι οι συνάδελφοι, ιδίω όσοι ήρθαν μετά το 2009, πρέπει να κατανοήσουν ότι όταν διαπραγματευόμαστε το θέμα αυτό, ως κοινοβούλιο στην ψηφοφορία μας στην Επιτροπή Ήτρε και στην, και στην Επιτροπή ΕΝΒΗ έχουμε ε, τροπολογίες και η δικιά μου τροπολογία η 199 ψηφίστηκε με 50 υπέρ ε, στην ε, Επιτροπή Ήτρε και δύο κατά και ο Άντρες Βίκμαν ε, είχε κάτι άλλο, ε, κάποια άλλη γνωμοδότηση παράλληλα στην Επιτροπή ε, Ήτρε. Τελικά, στο Κοινοβούλιο έγινε αποδεκτό να μην αποφασίζουμε λαμβάνοντας υπόψη όλους τους παράγοντες. Και αν εμείς ως Κοινοβούλιο στις διαπραγματεύσεις μεταξύ Κοινοβουλίου, Συμβουλίου, όπου ήταν παρούσα και η Επιτροπή βέβαια, αν εμείς τελικά αποδεχθούμε να αποσύρουμε κάποιες τροπολογίες ή να μην επιμείνουμε σε κάποιες τροπολογίες μας, Υπάρχουν ε, υπάρχει συγκεκριμένη στάση για το iLook. Αν περάσουμε σε μια διαδικασία που ζητάμε από την Επιτροπή να το λάβει υπόψη σε μια έκθεση και να προτείνει σχετική νομοθεσία το 2011 ή αργότερα, αρχίζει να είναι ε, πηγαίνει ανησυχία αν βλέπουμε ότι τμήμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής όχι μποϊκοτάρει γιατί είναι πολύ έντονο αυτό αλλά τουλάχιστον δεν ε, ανταποκρίνεται σε αυτό το οποίο σαφώς ε, είχε αναλάβει ως πολιτική δέσμευση στην συμφωνία του Δεκεμβρίου του 2008. Και στην οδηγία αιτιολογική σκέψη 85, καθώς και το άρθρο 19.6, σαφώς αναφέρουν ότι πρέπει να βασίζεται σε επιστημονικά στοιχεία και στον παράγοντα iLook και από τις 31 Δεκεμβρίου και μετά και το 2011 είναι κάτι το οποίο πρέπει να επιληθεί. Καταλαβαίνω λοιπόν από αυτά που μας λέει η Επιτροπή ότι ακόμη δεν είναι σε θέση να μας δώσει μια έκθεση στις ημερομηνίε που είχαν ε, μπει στα σχετικά κείμενα. Και αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι στο πρόγραμμα δράσης για το 2011 πουθενά δεν γίνεται μνήα της έκθεσης ή της ε, συναπόφασης. Χρειαζόμαστε λοιπόν κάποια διασφάλιση από εσά ότι όντως σας απασχολεί σοβαρά το θέμα Γιατί μιλάμε για την πρακτική εφαρμογή, την εφαρμογή στην πράξη ενό θέματο που αποφασίστηκε από το Συμβούλιο και το Κοινοβούλιο. Ο Μπάς Άικουτ, που τον ενδιαφέρουν ιδιαίτερα τα μοντέλα χρήση γη, σίγουρα θα μιλήσει για το θέμα αυτό. Πιστεύουμε ότι το iLook είναι μια παράμετρος πολύ σημαντική και δεν υπάρχουν παράμετροι που να δείχνουν ότι το iLook δεν είναι αρκετά σημαντικό. Ένα άλλο δεύτερο θέμα και ως εισηγητής για την οδηγία αυτή. Έλεγα πάντοτε ότι το κρίσιμο τεστ για αυτή τη νέα νομοθεσία είναι το πώς αντιδρούν σε αυτή οι παράγοντες της αγοράς. Είδαμε τις επενδύσεις στους διάφορους τομείς ανανεώσιμων πηγών ενέργειας. Από τον τομέα των βιοκαυσίμων δεν έχουμε σχετικές ε, αναλύσεις και από τους αναλυτές από την Bloomberg παραδείγματος χάρη μας λένε ότι όλος ο τομέας γύρω από τα βιοκαύσιμα δεν κάνει επενδύσεις είναι επιφυλακτικοί στις επενδύσεις γιατί δεν ξέρουν πώς θα εξελιχθεί η αγορά. Και αν μιλήσουμε σε αυτούς που είναι έτοιμοι να μπουν στη δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων, που είναι πιο εξελιγμένα βιοκαύσιμα, τα βιοκαύσιμα που θα έχουν πολύ χαμηλότερο παράγοντα iLook, η απάντησή τους είναι ότι το πλαίσιο που έχουμε σήμερα, που έχει διπλή επιβράβευση για τη δεύτερη γενιά, δεν είναι αρκετά ισχυρό για να ε, για τα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς. σκεφτήκαμε τι αντικαθιστά την κυροζήνη και αν έχουμε και πιο αποτελεσματικά ε, φορτηγά και εξετάσουμε τι θα αντικαταστήσει την ε, ε, το καύσιμο μετά το 2020-2030, αν δεν είναι η βιομάζα, τι θα είναι. Χρειαζόμαστε επενδύσεις στα βιοκαύσιμα δεύτερης γενιάς για να έχουμε και μία ε, αξιόπιστη λύση μακροπρόθεσμα για να έχουμε τις μειώσεις που συμφωνήσαμε. Ζητάμε λοιπόν από την Επιτροπή να εξετάσει αυτήν την παράμετρο του iLook για να μπορέσουμε να καταλάβουμε καλύτερα την αγορά. Ευχαριστούμε πολύ, Κλοντ. Κρις Τέιβις. Ευχαριστώ. Ελπίζω ότι θα υπάρξουν πολλοί στην Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα θέλουν να σώσουν τα προσχήματα για αυτό το θέμα. Γιατί σε αυτή την Επιτροπή πολλοί θα σας πούνε «σας το είπαμε» αν αλλάξετε την νομοθεσία. Σας είχαμε νομοθεσια σας ειχαμε προειδοποίησει», θα σας πούμε. Εγώ Προσωπικά ήμουν ενθουσιώδης με τη χρήση των βιοκαυσίμων πριν από μερικά χρόνια. Όσο προχωρούσε η νομοθεσία άρχισαν να μπαίνουν αφιβολίες στο μυαλό μου, συζητώντας και με διάφορους. Ο χρόνος προχώρησε. Σήμερα η ζήτηση της Ευρώπης οδηγεί στην καταστροφή οικοτόπων. Καταστρέφεται η επικοινομορφία και αυτό που είπε ο Κλοντ είναι σωστό. ότι είναι και θέμα επενδύσεων στη δεύτερη και στην τρίτη γενιά βιοκαυσίμων. Θα έλεγα λοιπόν περιμένετε δεν μπορούμε να εφαρμόσουμε την αρχή της προφύληξης, δεν μπορούμε δηλαδή να ανακαλέσουμε, δεν μπορούμε να το ξαναδούμε και να μας δώσετε μια ιδέα για το χρονοδιάγραμμα που έχετε στο μυαλό σας. Πώς θα θεωρηθεί, θα επαναξιολογηθεί η κατάσταση κτλ. βάσει της παρούσας νομοθεσίας. Λίντα Μακάβεν όπως και ο Κρίς, έτσι και εγώ. Πριν από δύο χρόνια όταν συζητήσαμε, δεν ήμουν υπέρ της καμπάνιας Stop Biofuels. Είχαμε συζητήσει για τα κριτήρια βιωσιμότητας και είχαμε πει ας συνεχίσουμε, ας προσπαθήσουμε να προχωρήσουμε στη δεύτερη γενιά βιοκαυσίμων. Μετά όμως άρχισα να διαβάζω τις εκθέσεις από διάφορους οργανισμούς, από το Ινστιτούτο για την Ευρωπαϊκή Πολιτική Περιβάλλοντος, από τη UNEP, ε, του Ηνωμένου Βασιλείου, ε, περιβαλλοντικές οργανώσεις της Ολλανδίας κλπ. Και πρόκειται για οργανώσεις διεθνούς φήμης, αξιόλογοι οργανισμοί είναι όλοι αυτοί, που έβαλαν και στο δικό μου το μυαλό αμφιβολίες. Και πριν από μερικές εβδομάδες συζητούσαμε για δεκάδες χιλιάδες οικογένειες στην Ανατολική Αφρική που θα έπρεπε να μετατοπιστούν από ε, κάποιες επιχειρήσεις που ανέπτυσαν τα βιοκαύσιμα. Δεν είναι δυνατόν να κάθεσαι και να τα κοιτάς αυτά, επειδή όπως είπε και ο Κρίς πριν από δύο-τρία χρόνια είχαμε πει ναι, ναι, Τώρα η Ευρωπαϊκή Επιτροπή θα μας πει αν είναι αλήθεια. Τελικά μήπως η Ευρωπαϊκή Επιτροπή το βρίσκει πολύ δύσκολο και δεν θέλει να βουτήξει. Δεν θέλει να μας προτείνει τον ε, παράγοντα αυτόν που ανέλησε πριν και ο συνάδελφος. Γιατί είναι και θέμα επενδύσεων και εσείς κάνατε επενδύσεις. Πρέπει να είμαστε ξεκάθαροι τι μηνύματα στέλνουμε, τι θέλουμε. Δεν νομίζω ότι πρέπει να πιέσουμε λοιπόν, ώστε τα Χριστούγεννα να την έχουμε αυτή την πρόταση της Επιτροπής, αν δεν είμαστε σίγουροι ότι θα έχουμε τη σωστή πρόταση, αν χρειαστεί παραπάνω χρόνο, σας χρειαστεί. Και δεν βλέπω γιατί δεν έχουμε το χρονοδιάγραμμα. Δεν ξέρω. Χρειάζεται μεγαλύτερη σαφήνεια και μηνύματα από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή ότι η Επιτροπή είναι ομόφωνα υπέρ. Όλες οι γενικές διευθύνσεις δηλαδή. Μάλιστα. Πρόεδρε. Ευχαριστώ και ευχαριστώ και την Κομισιόν ε, για όσα δήλωσε για το θέμα αυτό. Όλα αυτά είναι ζωτική σημασία, κυρίως για την αξιοπιστία ε, των στόχων που θέλουμε να πετύχουμε το 2020 σε ό,τι αφορά τις εκπομπές. Ε, η συζήτηση συνεχώς συνεχίζεται και πάντοτε το ερώτημα είναι έτοιμη η επιστήμη για κάτι τέτοιο. Και πρέπει να είμαστε σαφείς αν δούμε όλες τις μελέτες που υπάρχουν δεν αναφέρθηκαν ε, και από τους συναδέλφους, δεν υπάρχει καμία μελέτη που να λέει ότι δεν υπάρχει ε, μέση αλλαγή χρήση της γης. Όλες οι μελέτες δείχνουν ότι υπάρχει αντίκτυπος ε, μέση μεσιαλλαγής της χρήσης της γης και υπάρχει αντίκτυπος στους στόχους που θέλουμε να πετύχουμε το 2020. Και αναφέρομαι μόνο στο διοξείδιο του άνθρακα, δεν μιλάω καν για τον αντίκτυπο της αμεσής αλλαγής χρήσης γης για τη βιοπικιλότητα. Ε, τουλάχιστον αυτά δεν λαμβάνονται υπόψη στη διαδικασία, στην οδηγία περί ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και νομίζω ότι είναι σημαντικό να παρουσιάσουμε μια τέτοια πρόταση γιατί κανένα επιστημονικό ίδρυμα δεν λέει ότι δεν θα πρέπει να παρουσιάσετε ε, κάτι τέτοιο. Φυσικά υπάρχουν ε, κάποιες βιομηχανίες ε, που δεν είναι έτοιμες για κάτι τέτοιο, κάποιοι τομείς, ναι, μπορώ να το καταλάβω και κάποια κράτη-μέλη δεν είναι ακόμη πεπισμένα, αλλά εγώ δεν έχω δει καμία επιστημονική απόδειξη που να λέει ότι δεν υπάρχει εδώ αξία. έτσι λοιπόν, Κομισιόν, σας παρακαλώ, εντάξει, εγώ δεν θέλω με λίγα και με δόντια εδώ να υπερασπίσω την προθεσμία του Δεκεμβρίου, αλλά νομίζω ότι είναι πιο σημαντικό να έχουμε εδώ τα ορθά στοιχεία για αυτή την ε, έμεση αλλαγή χρήσης ε, της γης ε, εδώ. Είχαμε πάρα πολλές φορές διάφορες υποθέσεις. Αν δούμε τι είχε γίνει στην αρχή, ότι αν το κάνουμε αυτό για τη γάμα δέλτα εμπορίου, τότε θα δουν μόνο την εφαρμογή 5,6% και θα δουν το 50% της εθανόλης και το 50% του δίζελ. Ξέρουμε ότι αυτές οι υποθέσεις δεν ισχύουν για το τι θα γίνεται το 2020. Δείτε τα σχέδια εφαρμογή από την οδηγία για τις ανανεώσιμες. Βλέπετε εδώ ότι πάνω από το 90% προέρχεται από τα βιοκαύσιμα και μάλλον θα έχουμε 25 με 75% ε, για το βιοδίζελ ε, έτσι λοιπόν ε, έχουμε αυτό το JRC, το, αυτό το ίδρυμα ε, το οποίο σας παρακαλώ ε, όταν εργάζεστε με τέτοιες υποθέσεις δείτε και το διαχωρισμό μεταξύ diesel και βιοθανόλης και τότε θα ξέρουμε ότι έχουμε ε, πραγματικές τιμές και στοιχεία για την έμεση αλλά και της χρήσης γης. Εφαρμόστε τα αυτά το 2011 και μπορούμε να δώσουμε τα σωστά μηνύματα σε αυτούς τους τομείς και τις βιομηχανίες που αναζητούν αυτά τα στοιχεία για να πετύχουμε όλο αυτό που θέλουμε τελικά. Ευχαριστώ κύριο Πρόντι. Ευχαριστώ Πρόεδρε. Εγώ είμαι παντότε πάρα πολύ σκεπτικός ε, μεταξύ της διάκρισης βιοκαυσίμων ε, πρώτης και δεύτερης γενιάς. Εγώ νομίζω ότι η διαφορά είναι μόνο αυτή ότι στη δεύτερη γενιά ολόκληρη η βιομάζα το σύνολο της βιομάζας θα έπρεπε να, το, να είναι αντικείμενο εκμετάλλευση. Και έτσι στην περίπτωση αυτή εγώ θα ήθελα να αναφερθώ και στο μας της ε, στα βιολογικά δηληστήρια γιατί θα μπορούσαμε να έχουμε και την κατάσταση του πετρελαίου με πρώτες ε, ύλες που προέρχονται από τα υπολείμματα της βιομάζας. Εδώ τώρα θα ήθελα να πω το εξής πριν ε, να μπούμε στην εξέταση ενός ζητήματο που έχει να κάνει με την έμεση αλλαγή της ε, χρήση να πούμε ότι το έδαφος είναι ένας ε, σπάνιος πόρος που πριν να κάνουμε λοιπόν αλλαγές θα πρέπει να σκεφτούμε πολύ καλά. Δεύτερον, καθώς ήδη υπάρχουν σημαντικές ποσότητες βιομάζας διαθέσιμες, πριν να αναλάβουμε πολύ ισχυρέ δεσμεύσεις, ε, ίσως θα μπορούσαμε να παγιώσουμε τις τεχνολογίες που έχουμε για τα κατάλοιπα πριν να κάνουμε αλλαγές στη χρήση της γης. Και σκεφτόμενοι πάντοτε το έδαφος που είναι ένα σπάνιος πόρος, πριν να κάνουμε τα πράγματα αυτά θα μπορούσαμε ακόμη να ε, λειτουργήσουμε έτσι ώστε να και να έχουμε όλα τα κατάλληλα εργαλεία για να προβούμε σε μια παρατήρηση. Ε, κυρίως του χώρου μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε και τα συστήματα GMS, ε, παρατήρησης της γης, που είναι απολύτως απαραίτητα. Έτσι λοιπόν ε, πρέπει να χρησιμοποιήσουμε τα εργαλεία αυτά για να γνωρίζουμε ποια είναι ακριβώς η κατάσταση του εδάφους και πώς ακριβώς χρησιμοποιείται. Και στη βάση αυτή θα μπορούσαμε να προσπαθήσουμε και να επιταχύνουμε την εφαρμογή του δορυφορικού συστήματος για να μπορέσουμε στη συνέχεια να είμαστε σίγουροι ότι διαχειριζόμαστε σωστά τις πολιτικές μας. Ευχαριστώ. Grazie, Επόμενη ομιλήτρια, Ρίτα Μάνεν. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ τον εκπρόσωπο της Επιτροπής για την πολύ καλή περιγραφή του θέματος που μας έδωσε και όπως είπαν και πολλοί οι προηγούμενοι ομιλητές είναι σημαντικό να καταλήξουμε σε κάποια συμφωνία για το θέμα αυτό και να επιτύχουμε τους στόχους του 2020. Δεν θα επαναλάβω αυτά τα οποία ήδη ελέγχθησαν. Θέλω να κάνω μια ερώτηση προς την Επιτροπή όμως όσον αφορά τη χρήση της τύρφης ως τμήμα της βιοενέργειας και των δύο Ξέρω ότι διχάζονται οι απόψει από αυτού και ότι υπάρχουν σχετικέ συζητήσει που διεξάγονται. Αλλά θα ήθελα να πω ότι στην Ευρωπαϊκή Ένωση η τύρφη είναι διαθέσιμη. Και είναι πόρος που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε αντί να αγοράζουμε άνθρακα ή οτιδήποτε άλλο από άλλες χώρες εκτός Ευρωπαϊκής Ένωσης. Άρα πιστεύω ότι πρέπει να χρησιμοποιούμε την τύρφη. Παραδείγματο χάρη στη Φινλανδία αυτή τη στιγμή πάνω από 100 σπίτια ε, θερμαίνονται με τη χρήση τύρφης. Η τύρφη είναι ένας φυσικός πόρος που ανανεώνεται με αργούς ρυθμούς και θα ήθελα να ζητήσω από την Επιτροπή να μας πει ποια είναι η γνώμη της για τη χρήση τύρφης. Ο κύριος Φανστέν και ο κύριος Όουεν θα μας απαντήσουν. Ποιος θα ξεκινήσει, όπως πριν ή αντιστρόφως. Ε, Φανστέν. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Και ευχαριστώ για όλα τα ωραία σχόλια που ακούσαμε. Κοιτάξτε, δεν θα επαναπαυθούμε, θα δούμε χρονολογικά λίγο. Για το πρώτο θέμα, δεν έχουμε σήμερα την ενημέρωση. Για το δεύτερο, για το Red Plus και το Cancun. Ξέρουμε πολύ καλά βέβαια τι γίνεται στο Cancun, εννοείται, και ελπίζουμε ότι θα ληφθεί κάποια απόφαση, θα υπάρξει κάτι θετικό για το ΡΕΤ. Βέβαια πρέπει να δούμε πώς θα επιδράσει αυτό στη δουλειά μας για το άλλο γενικότερα. Είναι κάτι που το παρατηρούμε. Θα δούμε τι θα γίνει στο Κανκούν και τι μπορούμε να κάνουμε στη συνέχεια με αυτό. Σε σχέση με το άλλο. Πολλές ερωτήσεις. Στέρνες, Ντέιβις, Λίδα Μακάβεν και άλλοι. Όλοι με ρωτήσατε για το χρονοδιάγραμμα. Μπορώ να σας πω πού βρισκόμαστε και πού πιστεύουμε ότι πάμε χρονικά. Ο και εγώ μόλις ερχόμαστε από μια συνάντηση όπου συζητήσαμε την έκθεση που προβλέπεται για τα τέλη της χρονιάς να προταθεί για νομοθεσία. Ελπίζουμε ακόμα ότι θα είναι έτοιμη πριν από τα Χριστούγεννα, ίσως λίγο μετά, γύρω στις 31 Δεκεμβρίου ας πούμε ότι πιστεύουμε πως θα βγει. Και θα λέει τι έχουμε κάνει όσον αφορά τις μελέτες μας τους τελευταίους 12 μήνες και θα αντικατοπτρίζει λίγο και αυτά τα οποία λαμβάνουν χώρα στη διαβούλευση. Δηλαδή τι μας ε, απάντησαν οι άνθρωποι στις ερωτήσεις που θέσαμε εγώ. Και από εκεί και πέρα θα τίθεται και κάποιες ε, επιλογές προς τα που θα ήθελε να πάει η Ευρωπαϊκή Επιτροπή. Με αξιολόγηση για το 2011, ώστε το καλοκαίρι του 2011 να έχουμε ολοκληρώσει. Προσπαθούμε πρώτα απ' όλα να πετύχουμε την προθεσμία του Δεκεμβρίου για πράγματα που δεν έχουμε ασχοληθεί τα τελευταία χρόνια. Ξέρετε, είναι ένας δύσκολος τομέας. Υπάρχουν αβεβαιότητες και επιστημονικά, αλλά υπάρχουν και πολλά προβλήματα με τα μοντέλα. Προσπαθούμε να τα αναπτύξουμε λοιπόν όσο γίνεται καλύτερα για να έχουμε μια καλή βάση για να γίνει η αξιολόγηση του χρόνου. Το θέμα δεν είναι το νομοθετικό πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, μην περιμένετε κάτι εκεί. Owen. Συμφωνώ με αυτά που είπε ο Φίλιπ Φανέστερ για το χρονοδιάγραμμα πάνω στο οποίο δουλεύουμε. Πάντως, να πω και μερικά πράγματα ακόμα. Δεν μ' αρέσει να διορθώνω τον κύριο Τέρνες, αλλά η οδηγία περιλαμβάνει τον όρο εφόσον ε, πρέπει, εφόσον κριθεί επιθυμητό. If appropriate. Δηλαδή, η Επιτροπή θα μελετήσει το θέμα δεν λέει ότι πρέπει οπωσδήποτε να φέρει τον παράγοντα ILOC. Λέει ότι η Επιτροπή πρέπει να μελετήσει το θέμα και να κάνει πρόταση if appropriate. Για τα άλλα θέματα που θέσατε, με τον κύριο πρώτη πολύ σωστά λέτε ότι η γη είναι ένα σπάνιο αγαθό. Και όντω γι' αυτό και υπάρχει και αυτή η έμεση αλλαγή στη χρήση γης. Έχει να κάνει με το πώς θα χρησιμοποιήσουμε τη γη μας και με το πώς χρησιμοποιούνται οι εκπομπές του εξωτερικού του Τώρα στην Ευρώπη είναι ενδιαφέρον να δούμε ότι δεν επεκτείνουμε τη γη που χρησιμοποιείται για γεωργία και ότι επεκτείνουμε τα δάση μας. Είναι καλό δηλαδή να πούμε ότι εδώ δεν υπάρχουν επιπτώσεις από την ε, χρήση ή την καλλιέργεια βιοκαυσίμων. Για την κυρία Μάνε τώρα. Δεν είναι ένα καινούριο θέμα αυτό της στήρφης που θέτεται συζητήθηκε και κατά τις διαπραγματεύσεις για την οδηγία τότε η Επιτροπή είχε τη θέση και ξεκολουθεί να την έχει ότι δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας η τύρφη. Σύμφωνα με την οδηγία είναι η βιομάσα και η τύρφη δεν είναι βιομάσα. Βέβαια δεν σημαίνει αυτό ότι η τύρφη δεν έχει πολλά πλονεκτήματα την έχουμε στις χώρες μας, είναι μια πηγή που μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε. Και ίσως θα μπορούσαμε να χρησιμοποιήσουμε την τύφη σε ε, περιπτώσεις δεύτερης γενιάς βιοκαυσίμων. Αλλά από μόνη της δεν είναι ανανεώσιμη πηγή ενέργειας και γι' αυτό δεν περιλαμβάνεται, δεν, δεν καλύπτει τις προϋποθέσεις δηλαδή που περιλαμβάνονται στους στόχους της χιλιτίας. Νομίζω ότι κάλυψα τα διάφορα σημεία. Α, ένα τελευταίο. Αναφερθήκατε σε μια μελέτη και τώρα βέβαια μπαίνουμε σε τεχνικά ζητήματα. Τέτοια ώρα είναι λίγο δύσκολο. Πάντως, όχι, ούτε μας μας φοβίζει. Αν δούμε διάφορα σενάρια, το 5-6% που είπατε εσείς, αλλά υπάρχει και ένα άλλο 8,6% που αναφέρεται σε μια άλλη μελέτη. καλυπτόμαστε. Αλλά όπως είπε και ο κύριος ε, και συνάδελφος, είναι τα μοντέλα που μας δημιουργούν δυσκολία και γι' αυτό χρειαζόμαστε, αυτός είναι ένας από τους λόγους για τους οποίους χρειαζόμαστε περισσότερο χρόνο πριν ε, ολοκληρώσουμε την πρότασή μας. Πάντως μόλις έχουμε την έκθεσή μας και ελπίζουμε γρήγορα, θα είμαστε πάλι στη διάθεσή σας. Ευχαριστούμε πολύ την Επιτροπή και ευχαριστούμε και όλους τους συναδέλφους. Ευχαριστούμε και τους διερμηνείς. Τέλος συνεδρίασης και από το πρωί στις 9 αρχίζουμε με την ψηφοφορία για διάφορες εκθέσεις.